Monsieur le euh, Χαιρόμαστε πάρα πολύ που σας υποδεχόμαστε εδώ, κύριε για αυτή την πρώτη επίσημη παρουσία σας ε, στην ε, Επιτροπή Μεταφορών. Υποδεχόμαστε στο πρόσωπό σας στην Βελγική Προεδρία και πραγματικά υποθέτουμε τις ελπίδες μας σε εσάς. Έτσι λοιπόν θα σας δώσω το λόγο για να σας ακούσουμε. Merci, euh, Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι αξιότιμοι κύριοι βουλευτές, καταρχήν θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που με καλέσατε να παρευρεθώ ενώπιόν σας εδώ στην Επιτροπή Μεταφορών για να σας παρουσιάσω τις προτεραιότητες της Προεδρίας για την κινητικότητα και τις μεταφορές. Είμαστε πεπισμένοι ότι θα υπάρξει επικοδομητική συνεργασία μεταξύ της Επιτροπής Μεταφορών, της Κομισιόν και του Συμβουλίου. Και φυσικά η δική σας υποστήριξη είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να προωθήσουμε τα θέματα της κινητικότητας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είδα, έχω έλθει σε δημαρίες επαφές με τους Ευρωπαίους ε, συναδέλφους μου, με την Κομισιόν, με τη Γραμματεία του Συμβουλίου και με κάποια μέλη της Επιτροπής ε, Μεταφορών και αυτές οι διμερείς ε, επαφές ε, μας έκαναν να κατανοήσουμε ότι το πρόγραμμά μας είναι φιλόδοξο. Οι προτεραιότητες που έχουμε θέσει είναι ρεαλιστικές, επίκαιρες και εφικτές. Το πρόγραμμα, το πρόγραμμα μας βασίζεται σε έξι προτεραιότητες και σε μία σειρά εκδηλώσεων που θα τις πλαισιώσουν. Ε, αυτές οι προτεραιότητες συνδέονται συχνά με τη συνέχιση των ε, φακέλων που είναι ήδη υπό εξέταση και φυσικά με το πρόγραμμα εργασίας της Κομισιόν. Χαίρομαι που διαπιστώνω ότι τα ευρωπαϊκά όργανα ήδη το 2010 κατέληξαν σε συνένεση επί ουσιαστικών ζητημάτων, εκ των οποίων και η ηλεκτρονική εξέταση των εγγράφων στις ελεύθερες μεταφορές, οι διάδρομοι για τις συνδρομικές μεταφορές, το κανονισμός για την πρόληψη των ατυχημάτων στον, στις αερομεταφορές και Επίσης, ο κανονισμός που αναφέρεται στην τροποποίηση του ρόλου των αποπτικών αρχών του Γαλιλαίου και επίσης ε, για τα δικαιώματα των επιβατών στις θαλάσσιες και πλωτές μεταφορές. Θα πρέπει να εγγυηθούμε ένα βιώσιμο μέλλον για τις μεταφορές, δίνοντας έμφαση στην ασφάλεια. Σε όλους τους τρόπους μεταφοράς θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε την καινοτομία Πρόκειται για ένα βασικό στοιχείο για το πρόγραμμα της Βελγικής Προεδρίας αλλά και για το σύνολο των προκλήσεων που έχουμε στα πλαίσια της ανάπτυξης της κινητικότητας. Καταρχήν θα ασχοληθούμε με τη Λευκή Βίβλο για το μέλλον των μεταφορών. Αυτή η λευκή βίβλος θα περιλαμβάνει ε, ουσιαστικά μία απάντηση στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε στον τομέα των μεταφορών. Το Βέλγιο θέλει να συνεισφέρει επικοδομητικά στην εκπόνηση και στην εφαρμογή αυτής της λευκής βίβλου και μας φαίνεται σκόπιμο να οργανώσουμε μία γενική ανταλλαγή προαπόψεων στην συνάντηση του Συμβουλίου τον Οκτώβριο προκειμένου να έχουμε ένα τελικό κείμενο το Δεκέμβριο το οποίο θα υιοθετηθεί. Και θα πρέπει να σκεφτούμε και τη διεθνοποίηση των εξωτερικών συνιστοσών σε μια διατροπική προοπτική. Θέλουμε να ξανανοίξουμε λοιπόν τη συζήτηση αυτή. Επίσης θα πρέπει να αναφερθούμε με την αναθεώρηση της οδηγίας για την Ευρωβινιέτα και θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο η Λευκή Βίβλος σε αυτό. Επίσης η Λευκή Βίβλος θα συνεισφέρει στο να προωθήσει την ανάπτυξη των πολιτικών των διευρωπαϊκών δικτύων μεταφορών. Κατά τη διάρκεια της Προεδρίας μας, όπως ήδη προτάθηκε στην διάσκευση για τα διευρωπαϊκά δικτύα της Σαραγώσα, θέλουμε να αναπτύξουμε την πολιτική και τη μεθοδολογία που θα μας επιτρέψουν να υλοποιήσουμε ένα ολοκληρωμένο διευρωπαϊκό δίκτυο μεταφορών με σαφείς προτεραιότητες. Επίσης, αναμένουμε τις προτάσεις της Κομισιόν για την αναθεώρηση του πρώτου σιδηροδρομικού πακέτου. Και μία συζήτηση για το θέμα αυτό θα πρέπει οπωσδήποτε να γίνει κατά τη διάρκεια της Βελγικής Προεδρίας. Επίσης, δίνουμε πολύ μεγάλη σημασία στην προώθηση της ασφάλειας ε, των μεταφορών και θέλουμε να λάβουμε γρήγορα από την Κομισιόν ε, το τέταρτο πρόγραμμα δράσης. Στο Συμβούλιο του 2 Δεκεμβρίου θα παρουσιάσουμε συμπεράσματα που θα μας επιτρέψουν να δώσουμε έμφαση κυρίως στους ποσοτικούς στόχους που θα συμπεριλαμβάνονται σε αυτό το πρόγραμμα δράσης. Το σχέδιο δράσης, οι ποσοτικοί στόχοι είναι οι πλέον κατάλληλοι για να μετρήσουν τα αποτελέσματα των μέτρων που έχουν ληφθεί, επιτρέποντας και μία αντικειμενική σύγκριση μεταξύ των κρατών μελών μέσω benchmarking. Επίσης θα αναπτύξουμε τις βέλτιστες τις δυνατές πρακτικές προκειμένου να μπορέσουμε να έχουμε τα καλύτερα διδάγματα ο ένας από τον άλλο. Τον Οκτώβριο το Βέλγιο οργανώνει με την Κομισιόν και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τις Ευρωπαϊκές ημέρες ασφάλειας στις μεταφορές. Η υλοποίηση της ε, ενίας αγοράς ε, και ε, η κυκλοφορία προσώπων και υπηρεσιών καθιστούν ε, απαραίτητη την υλοποίηση ενός ηλεκτρονικού συστήματος σε επίπεδο κρατών μελών σε σχέση με τους οδικούς κώδικες. Και αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει προοδευτικά να προωθήσουμε και τους υπόλοιπους τρόπους μεταφοράς πέρα των οδικών μεταφορών. Θα πρέπει να άρουμε όλα τα εμπόδια. Αυτό κυρίως για τις θαλάσσιες μεταφορές και πιο συγκεκριμένα για τις μεταφορές μικρών αποστάσεων. Ήδη έχουμε ε, αρκετή δυναμικότητα στις μεταφορές αυτές. Ό,τι αφορά τώρα την εφοδιαστική, εκεί πρέπει να έχουμε μια ολοκληρωμένη προσέγγιση και όχι μια προσέγγιση ανά τρόπο μεταφοράς. Έτσι λοιπόν στις 15 και 16 Σεπτεμβρίου θα οργανωθεί ένα άτυπο συμβούλιο στην Αμβέρσα το οποίο θα εξετάσει το θέμα της ε, ένταξης ε, των θαλάσσιων μεταφορών και των πλωτών μεταφορών στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς Αγαθών. Η παρουσία και η συνεισφορά της Επιτροπής Μεταφορών αναμένεται με ανυπομονησία. Παράλληλα, αναμένουμε και τη συνεισφορά του Επιτρόπου Συνκάλες και φυσικά και άλλων συναδέλφων από τα κράτη-μέλη. Είναι σημαντικό να θέσουμε σε εφαρμογή το σχέδιο δράσης Ναϊάδης. Πρόκειται για μια ενδιάμεση αξιολόγηση και αυτό θα γίνει και μέσω της διοργάνωσης μιας διάσκεψης για την μεταφορά των εμπορευμάτων στις αστικές περιοχές και επίσης θα έχουμε και μια συνδιάσκεψη σχετικά με τις πλωτές μεταφορές. Ε, η ΕΜΣΑ θα υποστηρίξει από τεχνική σκοπιά τις δραστηριότητες για ε, την ασφάλεια στη θάλασσα. Θα υπάρχει κατάρτιση των ε, αρμοδίων των κρατών βελών, θα υπάρξει εφαρμογή μέτρων περιβαλλοντικής προστασίας κτλ. Κάθε μέρα ο οργανισμός αυτός, ο ΕΜΣΑ, δείχνει πόσο χρήσιμος μας είναι. Οι αρμοδιότητες ε, αυτού του οργανισμού περιγράφονται στον κανονισμό 1406 του 2002. Αυτός ο κανονισμός ε, θα πρέπει να υιοθετηθεί και να, θα πρέπει συγγνώμη, να προσαρμοστεί. Το δεύτερο πακέτο θαλάσσιων μέτρων προβλέπει μια νέα σειρά μέτρων για την ασφάλεια στη θάλασσα. Σε ό,τι αφορά τώρα τις εναέριες μεταφορές, η κρίση που προέκυψε από το κλείσιμο του Ευρωπαϊκού Αέριου Χώρου κατόπιν της έκρησης του Ιρλανδικού, Ιρλανδικού, Ισλανδικού φεστίου προκάλεσε πολύ μεγάλες ε, αναταραχές αλλά μας οδήγησε και στο να σκεφτούμε, να προβληματιστούμε για τα δικαιώματα των επιβατών και για την αναγκαιότητα να έχουμε αποτελεσματικά διευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών. Φυσικά θα πρέπει να εξακολουθήσει να υπάρχει βελτίωση στις ενέργειες μεταφορές χάρη στην υλοποίηση του σταδίου 2 του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Ορανού και με την ανάπτυξη των ΦΑΠΣ το φθινόπωρο στην Μπρίζ θα λάβει χώρα μία διάσκεψη ε, για την εναέρια ασφάλεια και για το SS2, δηλαδή για το δεύτερο στάδιο του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Ουρανού. Εκεί θα μπορέσουμε να συζητήσουμε όλα αυτά τα θέματα. Η Κομισιόν ε, με είναι κίνηση για την διάμεση αναθεώρηση το 2010 για ε, τα συστήματα ε, πλοήγησης μέσω δορυφόρου, έγνος και γαλιλαίο. Και θα πρέπει η ανάλυση να γίνει από κοινού με την Κομισιόν και από τα κράτη-μέλη και το ε, γραφείο Ρολάν Μπερζέ. Εμείς ε, ελπίζουμε ότι αυτή η ενδιάμεση αναθεώρηση θα μας επιτρέψει να προβούμε σε ανάλυση των κινδύνων και έτσι θα μπορέσουμε να βελτιώσουμε την αποτελεσματικότητα του συστήματος αλλά και να προβλέψουμε και μια πολυετή χρηματοδότηση. Έτσι λοιπόν από τα τέλη του 2013 το Καλλιλέο θα πρέπει να έχει υλοποιηθεί πλήρως. Ο Επίτροπος Αντώνιο Ταζάνη κατά το Συμβούλιο Μεταφορών στις 24 του Ιουνίου παρουσίασε ένα σχέδιο δράσης για την εφαρμογή του Καλλιλέου. Θα αναφερθώ και εγώ στο θέμα αυτό στο Συμβούλιο προκειμένου να μπορέσουμε να φτάσουμε όσο το δυνατόν γρηγορότερα στην επιτέξη της για το GNSS μεταξύ κρατών μελών και Νορβηγίας και Ένωσης. Είναι επίσης σημαντικό να τονίσουμε τη σημασία του σχεδίου δράσης STE εμείς ε, θέλουμε η διαλειτουργικότητα των διαφορών συστημάτων να προωθηθεί και από την άλλη επιθυμούμε η εφαρμογή της οδηγίας πλαισίου STE να μην αποτελέσει πρόσκομα ε, στην ανάπτυξη της έρευνας και της καινοτομίας. Η εισαγωγή των STE στις οδικές μεταφορές θα πρέπει να οδηγήσει στη βελτίωση της ε, αηφορίας ε, και της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας. Αυτό το προ... Αυτές είναι οι προτεραιότητες του προγράμματος που ήθελα να σας παρουσιάσω. Ευχαριστώ. <coughs> Πρόεδρος, και τώρα θα δώσω το λόγο στον πρώτο συντονιστή Ματιά Γκρός πρώτος. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Υπουργέ και Προεδρεύοντα του Συμβουλίου. Ήδη κατά την ανάγνωση του προγράμματος εργασιών ε, του Βελγίου ε, είχαμε πει ότι είναι φιλόδοξο. Εντάξει, το λέμε. Ε, και εγώ με κάποια περηφάνεια, αλλά εν πάση περιπτώσει πρόκειται για κάποια ζητήματα εδώ που έχουν ε, περιληφθεί, τα οποία έχουν αναβληθεί εδώ και κάποιε προεδρίε. τα όσα περιλαμβάνονται. Θα τα βιώσουμε και εμείς τελικά ως προς την υλοποίηση και το ε, τι μπορεί να γίνει και ειδικότερα σε ό,τι αφορά ε, το κόστος, όχι μόνο στα μέσα μεταφοράς αλλά γενικά θα αποτελέσουν ένα από, τα, από τις κύριες παραμέτρους για τη δική μας πολιτική. Γιατί μιλάμε για μια πιο δίκαιη κατανομή των διαφορών ε, ποσοστών συγχρηματοδότησης σε αυτόν τον τομέα και ταυτόχρονα θα αποτελέσουν αυτές οι πολιτικές μια ενδιαφέρουσα πηγή εσόδων για τα κράτη-μέλη. Και ίσως ταυτόχρονα να είναι δυνατόν, ε, θα μπορέσει ενδεχομένως να είναι δυνατόν να δημιουργηθούν κάποιες γέφυρες χρηματοδότησης χωρίς να προβλέπεται αυτό το earmarking, δηλαδή η δέσμευση συγκεκριμένων κονδυλίων σε ό,τι αφορά συγκεκριμένα έργα για τα κράτη-μέλη, αλλά να δίνονται αντίστοιχα κίνητρα. Θεωρώ λοιπόν πως ε, με αυτές τις προσπάθειες η ασφάλεια στον εναέριο χώρο μπορεί να βελτιωθεί, χωρί βέβαια συγκεκριμένε αποφάσει τι οποίε ε, λαμβάνουμε, γιατί δεν έχουμε αρμοδιότητε, αλλά με κάποιε προτάσει τι οποίε ε, κάνουμε. Θέλουμε να διασφαλίσουμε λοιπόν την ε, ασφάλεια, δεν θέλουμε να αυξήσουμε το γραφειοκρατικό φόρτο εργασία. Και αυτό που θέλουμε να έχουμε είναι ένα συνεκτικό πλαίσιο, δηλαδή να μην λαμβάνει το κάθε κράτος μέλος διαφορετικές αποφάσεις, να υπάρχει δηλαδή μια συνοχή χωρίς να αποφασίζει ο καθένας, χωρίς να ε, υπάγεται σε ελέγχους. Και μιλάω εδώ για ε, τυποποίηση, για παράδειγμα σε ό,τι αφορά τον έλεγχο της μεταφοράς υγρών, στην, ε, σε πτήσεις ή τους σαρωτές σώματος. Με ε, τώρα την ε, πρωτοβουλία που ανέλαβε η Βελγική Προεδρία ε, θα εκινήσει ένα πολιετές πρόγραμμα το οποίο έδειξε με βάση και τα όσα κάναμε στο παρελθόν ότι μπορούμε να επιτύχουμε τους στόχους που έχουμε θέσει. Για αυτόν τον τομέα λοιπόν είναι πολύ σημαντικό αυτό. Εκείνο λοιπόν που είναι σημαντικό, επαναλαμβάνω, είναι να έχουμε ένα κοινό πολιετέ ε, πρόγραμμα το οποίο θα θέτει στόχου οι οποίοι είναι σημαντικοί για όλου του ενδιαφερομένου. Σήμερα το πρωί ακούσαμε την Ισπανική Προεδρία, ήταν σήμερα εδώ στην αίθουσά μα και αναφέρθηκε και στα μέτρα ασφαλεία στο σύνολό του που μπορούν να συμβάλλουν στα πλέον πλεονεκτήματα ενό κοινού ευρωπαϊκού εναέριου χώρου. Εγώ είπα ότι εύχομαι στο Συμβούλιο μερικά ηφαίστεια. Μερικά ηφαίστεια όχι μόνο στον αέριο χώρο αλλά και αλλού. Γιατί τελικά είδαμε ότι για παράδειγμα με ένα τέτοιο ηφαίστειο κάποιε αποφάσει ελήφθησαν πολύ γρηγορότερα. Για παράδειγμα σε ό,τι αφορά τον ενιαίο αέριο χώρο ε, πιο γρήγορα ελήφθησαν οι αποφάσει και αύριο ε, νομίζω έχουμε και μια τέτοια σημαντική απόφαση. Άρα λοιπόν βλέπουμε πω είναι ευκολότερο να υπάρχουν ρυθμίσει ενιαίε αντί για 27 διαφορετικές. Αύριο λοιπόν μπορούμε να έχουμε το καλύτερο ρυθμιστικό πλαίσιο. Αλλά αν εργαζόμαστε με 27 διαφορετικές, ε, διαφορετικά πρότυπα και με εκατοντάδες διαφορετικά επιμέρους εθνικά πρότυπα και στους σιδηροδρόμους αλλά και σε άλλους κλάδους τότε πραγματικά η καλύτερη ρύθμιση, το καλύτερο ρυθμιστικό πλαίσιο δεν θα μας βοηθήσει πολύ. Χρειαζόμαστε δηλαδή κοινή και καλύτερη υποδομή και χρειαζόμαστε αμοιβαία αναγνώριση αυτής της υποδομής και της τεχνολογίας ε, που χρησιμοποιούμε. Άρα λοιπόν ε, ε, ελπίζουμε πως θα μας δώσετε τη δυνατότητα να κάνουμε μια τέτοια κοινή συζήτηση. Γιατί αυτό που βιώνουμε με τους σιδηροδρόμους αυτή τη στιγμή δεν είναι ευθύνη των ίδιων των πολιτών. Είναι όμως ένα παράλογο σύστημα όταν βλέπουμε δηλαδή τις ρυθμίσεις τις οποίες καλούμαστε να εφαρμόσουμε. Άρα λοιπόν είμαστε ε, με το μέρο σα όταν λέτε ότι θα πρέπει να γίνει μια τέτοια συζήτηση. Θέλουμε να την κάνουμε με τη ελληνική Προεδρία. Η Επιτροπή ε, ήθελε να αναβάλει τη σχετική συζήτηση, δεν ξέρω για ποιου σκοτεινού λόγου δεν θέλω να το κάνω. Αλλά πραγματικά θα θέλαμε να σα καλέσουμε να ε, αρχίσουμε τη συζήτηση για αυτό το ζήτημα, το ταχύτερο δυνατόν. Το ίδιο ισχύει και για τη Λευκή Βίβλο. Μα είπατε πω θέλετε η πολιτική σα Προεδρία να συζητηθεί. Ε, και εμεί θα θέλαμε να υπάρξει μια λευκή ε, βίβλος ε, ε, που θα συζητηθεί για την περίοδο 2010-2020 μέσα στο 2010 και όχι μέσα στο 2011. Πρόκειται βέβαια για μια πρόκληση η οποία αφορά κυρίως την Ευρωπαϊκή ε, Επιτροπή και όχι την Προεδρία, αλλά θα μπορούσε να συμβάλλει η Προεδρία. Σε ό,τι αφορά τον χώρο της, των ναυτιλιακών μεταφορών, ναι, εδώ έχουμε να κάνουμε κυρίως με τον πυρήνα της ε, αποτελεσματικότητας, ε, δηλαδή αποτελεσματικότητα και καλή συνεργασία μεταξύ των διαφόρων μέσων μεταφοράς. Όχι λοιπόν ένας ανόητος ανταγωνισμός μεταξύ των διαφορετικών τρόπων μεταφοράς, αλλά αποτελεσματική συνεργασία τους. Και νομίζω πως και ο συνάδελφος Μιχάλη Κράμερ συμφωνεί με αυτή την προσέγγιση. Τέλος, οι διεθνείς συμφωνίες θα είναι σημαντικές για μας η αξιολόγηση της συμφωνίας με τις ΗΠΑ είναι κατά τη δική μου άποψη κάπως αισιόδοξη. Θεωρώ δηλαδή πως ε, η Ένωση αφού καλείται να ολοκληρώσει ε, και μέχρι το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο ε, τις σχετικέ διαβουλεύσεις να θέσει ε, πιο κατηγορηματικά κάποια ζητήματα. Δηλαδή ε, και η περίπτωση SWIFT έδειξε ότι όταν είμαστε λίγο πιο εμφαντικοί σε σχέση με αυτά που ζητάμε, μα ακούνε και καλύτερα οι Αμερικάνοι. Α λοιπόν κάνουμε κάτι τέτοιο σε σχέση με τη συμφωνία. Και τέλο. Να πω και ότι μετά την Κοπενχάγη το Βέλγιο θα χρειαστεί να προετοιμάσει το κακού. και θα πρέπει να δούμε το τι μπορούμε να κάνουμε και πώς μπορούμε να αναλάβουμε ένα πιο σημαντικό ρόλο εδώ. Γιατί μέχρι τώρα οι συζητήσεις αντιμετωπίζουν τις μεταφορές ως ένα απαραίτητο, ένα αναγκαίο κακό, αλλά ένα αναγκαίο κακό το οποίο εξασφαλίζει θέσει εργασία για περισσότερο από 10 εκατομμύρια άτομα, το οποίο έχει να παίξει ένα πολύ σημαντικό ρόλο σε σχέση με το περιβάλλον και κατά συνέπεια το οποίο μπορεί να συμβάλλει με τις κατάλληλες ρυθμίσεις στην μείωση των κομπών διοξιδίου του άνθρακα. Ε, εξ ονόματος λοιπόν της ε, πολιτικής μας ομάδας σας ε, εύχομαι ό,τι καλύτερο για τη δική σας Προεδρία και με βάση την πολύ καλή παράδοση των μικρών χωρών στην Προεδρία θεωρούμε πως πράγματι θα τα πάτε πολύ καλά και σας ευχόμαστε κάθε επιτυχία. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ Ματιέ. Σαΐτ, για τη συνέχεια. Ja, eh, meneer voorzitter, Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, το πρόγραμμα αυτό είναι φιλόδοξο αλλά και αναγκαίο γιατί οι μεταφορές έχουν ένα σωρό προκλήσεις μπροστά τους. Συμφόρηση, επίπτωση στο περιβάλλον, στο κλίμα και είναι και σημαντικός οικονομικός τομέας που δίνει δουλειά σε πολύ κόσμο. Τέλος, όλοι οι Ευρωπαίοι αντιμετωπίζουν το πρόβλημα της κινητικότητας. Η μεγάλη πρόκληση λοιπόν είναι να έχουμε ένα σύστημα πιο ενοποιημένο, πιο βιώσιμο και επιμένουμε η Κομισιόν σύντομα να προτείνει τη Λευκή Βίβλο και να μην περιμένει το τέλος της χρονιάς το 2011, γιατί το θέμα παρά είναι σημαντικό. Η Λευκή Βίβλος για τις μεταφορές θα πρέπει να αναφέρεται στο μέλλον, να έχει στόχους με νούμερα και ένα πρόγραμμα σε πολλά επίπεδα που θα εφαρμοστεί τα επόμενα έτη. Το Συμβούλιο μπορεί να εμπνευστεί από τη θέση του Κοινοβουλίου που πρόσφατα ψηφίσαμε. Για να πετύχουμε αυτούς τους στόχους χρειάζεται ένα φάσμα λύσεων. Πανάκια και λύση θαυματουργή δεν υπάρχει. Και η διάρθρωση των τιμών θα πρέπει να είναι στο πλαστάσιο μας και το ευρωσήμα, το αυτοκόλλητο, είναι, θα είναι κάτι σημαντικό και αυτό. Εμείς λέμε ας επιτραπεί στα κράτη-μέλη να διαχειρίζονται καλύτερα το κόστος της υποδομής, η εξωτερικοίευση του εσωτερικού χρέους, ε, κόστους, σε αυτό αναφερθήκαμε ήδη έτσι, ο τομέας αυτός θα γίνει πιο αποδοτικός και ταυτόχρονα θα μειωθούν και οι ζημιές που δημιουργούν οι μεταφορές. Αυτό είναι σημαντικό σε δύσκολους καιρούς του προπολογισμού που περνάμε. Θα πρέπει να μπουν νέα χρήματα στις μεταφορές. Υπολογίζω όπως όλοι μας στην Βελγική Προεδρία για να σημειωθεί μια πρόοδο στο θέμα αυτό και κατά κάποιο τρόπο μια μικρή επανάσταση μπορούμε να τη χαρακτηρίσουμε. Ας πέρασουμε τώρα στα διευρωπαϊκά δίκτυα. Συναντηθήκαμε στη Σαραγώσα, οργανώθηκε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Το συμπέρασμα είναι ότι τα μέχρι τώρα αποτελέσματα είναι περιορισμένα. Και ένα από τα μεγάλα προβλήματα είναι η χρηματοδότηση των μεγάλων έργων υποδομής στην Ευρώπη. Τα έργα αυτά για να υλοποιηθούν θα απαιτήσουν νέους και πιο δημιουργικούς χρηματοδοτικούς μηχανισμούς. Διαφορετικά όλα αυτά θα μείνουν νεκρό γράμμα και η οικονομική επίπτωση αυτών των επενδύσεων θα παραμείνει περιορισμένη. Το λέω αυτό ιδιαίτερα για τα σιδηροδρομικά δίκτυα. Αυτός ο μηχανισμός χρηματοδότησης με στα πλαίσια του ΤΕΝΤΕ έχει σημασία για το σύνολο της πολιτικής μεταφορών. Πρέπει να τονιστεί ιδιαίτερα η μεταφορά μέσω των σιδηροδρόμων με μεγαλύτερη ενοποίηση, δηλαδή να βελτιωθεί η σύνδεση που πρέπει να υπάρχει μεταξύ των χωρών, να κινούνται τα τρένα πιο γρήγορα. Αλλά δεν αρκεί αυτό. Πρέπει να, γίνει και πιο φιλικό προς το χρήση το μέσο αυτό, με ένα καλύτερο σύστημα έκδοσης εισιτηρίων, Φερρυπίν και έχουμε και το πρώτο σιδηροδρομικό πακέτο που πρέπει να βελτιωθεί. Τώρα, ασφάλεια στις μεταφορές. Περιμένουμε σύντομα ένα νέο πρόγραμμα δράσης μέχρι το 2020. 2010-2020 από την Κομισιόν. Αυτό όμως πρέπει να μεταφραστεί σε έργα, κύριε Υπουργέ. Έχουμε την πρόταση για τα πρόστιμα για παραβάσεις που έγιναν σε τρίτη χώρα. Επ' αυτού έχει αποφανθεί το Κοινοβούλιο. Προχωρώ γρήγορα στις αεροπορικές μεταφορές. Θα σταθώ σε δύο σημεία. Σε ένα σημείο μάλλον, με το οποίο δεν συμφωνούμε το Συμβούλιο, η χρηματοδότηση για τα μέτρα ασφαλείας στην πολιτική αεροπορία. Αυτή τη συζήτηση δεν μπορείτε να τη γλιτώσετε. Ξέρετε ότι το Κοινοβούλιο θέλει εναρμόνιση των μέτρων ασφαλείας. Και θεωρούμε ότι οι χώρες που θέλουν να πάρουν επιπλέον μέτρα θα πρέπει να πληρώσουν τη διαφορά. Ξέρω ότι στο Συμβούλιο δεν αρέσει αυτό, αλλά θα πρέπει να έχουμε περισσότερη διαφάνεια και στο θέμα αυτό και μια καλύτερη διαχείριση του εναέριου χώρου. Χρειάζεται να εισαχθούν ως πιο σύντομα γίνεται τα μπλοκ, τα τμήματα για τα οποία συζητήσαμε το πρωί και να διδαχτούμε από την έκρηξη του ηφαιστείου. Πιστεύουμε ότι αυτή η ιδέα μπορεί να υλοποιηθεί όλο Το πρωί ακούσαμε ότι 20 εκατομμύρια σύντομα θα δοθούν για πολλά από αυτά τα αεροπορικά μπλοκ, λειτουργικά τμήματα του ενέργειου χώρου. Και ένα σημαντικό κομμάτι θα πάει στον μπλοκ στο οποίο ανήκει και το Βέλγιο. Το Βέλγιο που λοιπόν μπορεί να παίξει ένα ρόλο ο μηχανής να δώσει το καλό παράδειγμα να κινηθούν τα πράγματα. Θαλάσσιες μεταφορές. Θετικό θετικές οι ιδέες που παρουσιάστηκαν από το Συμβούλιο στο άτυπο Συμβούλιο της Αμβέρσας. Θα πρέπει να γίνει μια καλύτερη οργάνωση μεταφοράς από τα λιμάνια προς το εσωτερικό σύνδεση με διάφορους τρόπους μεταφορών και ένα τελευταίο σημείο, τα δικαιώματα των επιβατών. Στα πλαίσια της Ισπανικής Προεδρίας σημειώθηκε ένα βήμα θετικό για μια συμφωνία για τα δικαιώματα των επιβατών ε, για τις θαλάσσιες και πλωτές μεταφορές. Μεταφορές όμως με πούλμαν και λεωφορεία ακόμα δεν έχει ρυθμιστεί το θέμα. Ελπίζουμε να υπάρξει βελτίωση σε αυτό. Να δοθεί μια μέγιστη, προστασία στα δικαιώματα αυτών των επιβατών. για τις αερομεταφορές πρέπει μια αξιολόγηση των δικαιωμάτων των επιβατών γιατί υπάρχουν ακόμα αρκετά κενά στην νομοθεσία που πρέπει να καλυφθούν. Εν κατακλείδη σας Επισημαίνω ότι έχετε πολλή δουλειά μπροστά σα. πάντως η ομάδα μας θα σας υποστηρίξει. Αν δείξετε φιλοδοξία μπορείτε να υπολογίζετε σε μας. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, ευχαριστούμε Σαΐντ. Η κυρία Κιάστερα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, για τα όσα μας είπατε θα ακούσετε αντίστοιχα πράγματα με αυτά που ήδη ακούσατε από του συναδέλφου. Ε, είναι πολύ θετικό το ζήτημα που ασχολείστε πάλι με την ε, Ευρωβινιέτα, γιατί ε, υπήρξαν προηγούμενοι συνάδελφοί σα που δεν απέλεξαν να μην ασχοληθούν με αυτό το ζήτημα, γιατί πραγματικά είναι δύσκολο και πραγματικά σα συγχαίρω για το ότι ασχολείστε και πάλι το θέτετε στην ημερησιαδέταξη, ακόμα και αν θα υπάρξουν δύσκολε συζητήσει σε σχέση με αυτό. Επίση, θα συμφωνήσω με τα όσα είπαν οι συνάδελφοι. Είχαμε πρόσφατα την έκθεση Ματσίου Γκρό σε ό,τι αφορά το μέλλον των μεταφορών και χρειαζόμαστε πράγματι επιγόντω τη λευκή βίβλο. δηλαδή έχουν, έχει δοθεί μια όθηση σε, όλα αυτά, σε όλη αυτή τη διαδικασία με αυτή την έκθεση γκρός οπότε καλό είναι να λάβουμε τη λευκή βιβλία το ταχύτερο δυνατό γιατί θα πρέπει να δώσουμε ακριβώς την έμφαση που πρέπει στις μεταφορές και ε, μ' άρεσε το γεγονός ότι αναφερθήκατε ξανά και ξανά στην εσωτερική αγορά, στην εννέα αγορά, γιατί ε, πράγματι έχετε δίκιο. Ε, δηλαδή πρέπει εδώ να προωθήσουμε κάποια ζητήματα όπως τη διαλειτουργικότητα. Ε, σε, στα χαρτιά υπάρχουν πολλά περί διαλειτουργικότητας, αλλά δεν έχουν εφαρμοστεί πολλά από αυτά. Άρα λοιπόν, εάν κάνετε κάτι σε αυτό το μέτωπο, ε, θα με χαροποιούσε πολύ. Σε ό,τι αφορά τώρα τα ευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών, τα TNT, ε, είπαμε ότι είχαμε τη μεγάλη διάσκεψη τη Αραγός, αλλά τώρα καλούμαστε να εφαρμόσουμε τα όσα αποφασίσαμε εκεί. Ε, ιεράρχηση προτεραιοτήτων σε ό,τι αφορά τα projects, τα διάφορα έργα. Αντιλαμβάνομαι ότι προφανώ πρόκειται για κάτι δύσκολο, αλλά κάπου θα πρέπει να επιτύχουμε και κάποια πρόοδο, ειδικότερα σε ό,τι αφορά και τα διασυνοριακά έργα τα οποία θα συγχρηματοδοτηθούν. Ένα ζήτημα τώρα που μας απασχολεί ειδικότερα από το ηφαίστειο και μετά είναι το ολοκληρωμένο σύστημα κρατήσεων. Για πρώτη φορά διασφαλίσαμε τα απαραίτητα κονδύλια για τη δημιουργία ενός τέτοιου ολοκληρωμένου συστήματος κρατήσεων για τους σιδηροδρόμους, για τις σιδηροδρομικές μεταφορές. Νομίζω πως κάτι τέτοιο θα ήταν πολύ καλό, πολύ ευνοϊκό για τους ε, πολίτες μας, ε, αν μπορέσουμε να επιτύχουμε εδώ κάποια πρόοδο. Τώρα, σε ό,τι αφορά γενικά τις ροές, ας το πούμε έτσι, μεταφορών, θα πρέπει να έχουμε αυτά τα ε, διαλειτουργικά τις λειτουργικές διαπαφές ας το πούμε έτσι και τα FAPS τα λειτουργικά τμήματα και το γεγονό ότι μας είπατε ότι πράγματι εδώ θέλετε να προωθήσετε και να επεκτείνετε περισσότερο και τι ε, ε, ναυτιλιακές και τι πρωτέ μεταφορές. Ναι, υπάρχουν εδώ κάποια προβλήματα ακόμα, αλλά θα πρέπει να ε, προσπαθήσουμε να τα επιλύσουμε. Υπάρχουν δηλαδή δυνατότητες, ακόμα δυναμικό που δεν έχει αξιοποιηθεί στις ναυτιλιακές μεταφορές και εναλλακτικά προς τις ε, οδικές μεταφορές θα πρέπει ακριβώς να προσπαθήσουμε να αξιοποιήσουμε αυτό το δυναμικό. Μας είπατε ότι θα έχετε αυτή τη διάστηση στην ε, Βέρσα σε ό,τι αφορά την καλύτερη ενσωμάτωση των ναυτιλιακών του πλωτών μεταφορών στο δίκτυο μεταφορών τη Ευρώπη Είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό, αλλά ο συνάδελφο Στέρξ είμαι, σίγουρο είμαι σίγουρη πω αναφέρει περισσότερα σχέση με αυτό, γιατί πραγματικά γνωρίζει πιο πολλά αυτό το ζήτημα. Και α, αυτή για τις εσωτερικέ εσωτερικές ε, οντούς, λοιπόν, η, ε, αυτό που θέλετε να κάνετε πολύ σωστό. Επίσης, ό,τι αφορά το Safe CNET, πράγματι βλέπετε τα όσα έχουμε να κάνουμε ε, από τα διάφορα φορτικά πλοία πετρελοκυλίδες και ούτω καθεξής. Ε, ίσως ε, καλό θα ήταν να αναλάβουμε κάποια δράση εδώ ούτω ώστε να αποδείγουμε τα όσα συνέβησαν στον κόλπο του Μεξικού. Βέβαια, αναφέρεται ξανά και ξανά το επιχείρημα ότι δεν αποβαίνουμε ε, σε τόσο ο Γεωτρής ε, στην Ευρώπη, αλλά πραγματικά θα πρέπει να δούμε λίγο τι ακριβώ κάνουμε στην Ευρώπη. Έχουμε ένα σχέδιο εκτάκτου ανάγκη για να προλάβουμε τέτοιες αντίστοιχες καταστροφές ε, στα δικά μα. ύδατα. Είναι κάτι που ε, σίγουρα θα θέλαμε να αποφύγουμε και θα πρέπει εκ των προτέρων να το καταπολεμήσουμε, να το προλάβουμε. Σε ό,τι αφορά τώρα τα δικαιώματα των επιβατών, εγώ είχα συμμετάσχει στον τριμερή διάλογο, χωρί όμω να επιτευχθεί τελικά εκεί μια συμφωνία και ελπίζω πως η πολιτική Προεδρία θα μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε αυτό το διάλογο γιατί δεν είναι δυνατό να έχουμε δικαιώματα για τους επιβάτες σε όλους τους άλλους ε, τομείς εκτός από τα λεωφορεία. Άρα λοιπόν ελπίζω πως πραγματικά από την δική σας Προεδρία να καταστεί δυνατό να ε, φτάσουμε σε μια συμφωνία η οποία θα είναι θα αποτελεί, θα συνεπάγεται μια μεγάλη πρόοδο για τους πολίτες μας. Ε, τώρα, σε ό,τι αφορά το χρηστιακό νέφος της τάχτης, ε, πραγματικά εδώ μας ταρακούνε σε αυτό ότι χρειαζόμαστε European Sky, χρειαζόμαστε ε, καλύτερες ε, συνδρομικές μεταφορές και μας είπατε πως θα υπάρξει μια διάσκεψη στο Bruges για τις νέες μεταφορές. Θα μπορούσατε να μας πείτε κάποια συγκεκριμένη ημερομηνία γιατί έχουμε και εμείς φορτωμένο πρόγραμμα. Καλό θα ήταν να ξέρουμε πότε θα είναι. Και σε ό,τι αφορά τις τεχνολογικές καινοτομίες κάνατε λόγο για τον Καλλιλέο είναι πολύ καλό αυτό που μας είπατε ότι θα γίνουν κάποιες αναλύσεις ε, κόστους ε, και ότι εντάξει, κάποια αρχή θα γίνει μετά από τη δική σας προεδρία, ότι παράλληλα αυτά όμως εσείς θα προσπαθήσετε να κάνετε κάποιες ε, προσπάθειες προς εκείνη την κατεύθυνση, γιατί πραγματικά όλοι περιμένουμε με μεγάλο ενδιαφέρον να ξεκινήσει η υλοποίηση αυτού του συστήματος. Και ε, τέλος έχουμε το ETS το οποίο πραγματικά έχει κάποια ωφέλη ε, πραγματικά σε ό,τι αφορά για παράδειγμα την αποφυγή των ε, κυκλοφοριακών συμφορήσεων και πρόκειται για έναν τομέα ο οποίος ε, ίσως υποτιμάει λίγο αυτό το ζήτημα γιατί μιλάμε για ένα ETS το οποίο και από πλευράς ασφάλειας και από πλευράς προστασίας του περιβάλλοντος είναι θετικό. Άρα λοιπόν ελπίζω πω υπό τη δική σας Προεδρία, αν μπορέσετε να ασχοληθείτε με όλα αυτά τα ζητήματα, θα ήταν πάρα πολύ θετικό. Σα ευχαριστώ πολύ. Καλό. Με συγχωρείτε. Λάθος, λάθος έκανα, λέει ο Προεδρό. Ο κύριο Κράμερ. Δεν πειράζει, υπάρχουν και χειρότερα, λέει ο κύριο Κράμερ. Ναι, ε, Εμεί έχουμε ήδη γνωριστεί και στη διασύνδεση τη Σαραγώσα. Μα είπατε πω έχουμε να κάνουμε εδώ με την βιώσιμη, με την ε, φόρο, το, ε, το αεφόρο, βιώσιμο μέλλον. Και πράγματι δεν έχουμε να κάνουμε ένα απλό επιθετικό προδιορισμό, μια ωραία λέξη. Α, θα πρέπει να λάβει και περιεχόμενο αυτή η λέξη. Και η Λευκή Βίβλος, ακόμα και αν περάσει γρήγορα, τίποτα δεν κάνει ακόμα. Δηλαδή αποτελεί απλά ένα παραπάνω χαρτί. Η πραγματικότητα είναι διαφορετική. Ε, μας ικανοποιεί το γεγονό ότι αναφερθήκατε στην Ευρωβινιέτα και την βάλατε στη δική σα ατζέντα γιατί ε, δύο προηγούμενε προεδρίε ούτε καν αναφέρθηκαν σε αυτό το ζήτημα στην παρουσίασή του, παρότι έχει αποφασιστεί εδώ και ένα χρόνο αλλά έχω να θέσω και σε σχέση με αυτό το ζήτημα ένα ερώτημα. Είπατε, μα είπατε ότι θα ε, το υποβάλλετε ε, το Δεκέμβριο. Δηλαδή τι σημαίνει αυτό, ότι πιστεύετε ότι δεν θα καταφέρετε τίποτα και ουσιαστικά θα δώσετε τη σκητάλη στην επόμενη Προεδρία. Δηλαδή, τι θα κάνετε ακριβώ, θα προσπαθήσετε να βρείτε το συμβασμό το Δεκέμβριο, να μα πείτε. Μετά, εσωτερήτευση των που λέμε, των, εξωτερικών, των εξωτερικών δαπανών, ναι, πράγματι ε, πρόκειται για ε, το σημείο στο οποίο ε, κρίνονται τα πάντα, το πούμε έτσι. Γιατί εδώ υπάρχει ένα πρόβλημα λέμε πως οι μεταφορές ε, είναι ευθυνές, αλλά αν θέλουμε πιο φιλοπεριβαλλοντικές μεταφορές είναι πιο ακριβές. Αυτό μιλάμε ότι, ε, ε, θεωρούμε ότι είναι ένα πολιτικό ζήτημα, μια πολιτική απόφαση. Άρα λοιπόν πρέπει να μας πείτε αν θέλετε να να ευνοείτε τις μεταφορές αυτές, τα είδη μεταφορών που έχουν αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον ή αν θέλετε να κατευθύνετε στις πιο ακριβές μεταφορές, αναλλακτικές μεταφορές. έχουμε ε, και στις ε, συνδρομικές μεταφορές αλλά και ε, στις οδικές μεταφορές κάποια ειδικά διόδια, ειδικότερα σε ό,τι αφορά φορτικά το τόνου και ούτω καθεξής, θα πρέπει να αλλάξουν εδώ κάποια τα πράγματα, κάπως τα πράγματα γιατί 30 δισεκατομμύρια ευρώ ε, πληρώνει ο Ευρωπαίος φορολογούμενος ώστε να μπορούν να ε, λαμβάνουν κάποια ειδικότερα ωφέλη οι αεροπορικές εταιρείες. Δεν μπορούμε δηλαδή όταν έχουμε την περίπτωση ε, του ηφαιστείου να εξετάσουμε μόνο τις δαπάνες για τις αεροπορικές εταιρείες. αν λαμβάνουν ο τομέας δηλαδή των αερομεταφορών 30 δις κάθε χρόνο τότε ας τα λαμβάνει και ο τομέας των σιδηροδρόμων. Μετά, εμείς κάναμε μία ανάλυση και είδαμε πως η συγχρηματοδότηση κατά 60% κατευθύνεται στις οδικές μεταφορές, 20% πηγαίνει στις δρομικέ μεταφορές και 0,9% πηγαίνει στους, ε, στα ποδήλατα, γενικά ποδηλατοδρόμου. Εμείς στο Κοινοβούλιο αποφασίσαμε ότι το 40% θα πρέπει να κατευθυνθεί προς το, ε, στους φιλοπεριβαλλοντικούς ε, Ο κ. Παρότο είχε αποδεχθεί τότε, αλλά τελικά υπήρξε μπλοκάρισμα από το Συμβούλιο και δεν πέρασε κάτι τέτοιο. Δεν μπορούμε όμως ε, να θέτουμε σε αυτούς μας ε, ε, στόχους όπως μείωση των εκπομπών κατά 20% έως το 2020 αλλά τελικά να μην επενδύουν καθόλου χρήματα στους τομείς που θα μας βοηθήσουν να επιτύχουν ένα τέτοιο στόχο. Μετά αναφερθήκατε και στην ασφάλεια των μεταφορών. Είναι σωστό αυτό, είχε συζητηθεί αυτό και στο Κοινοβούλιο πριν από ένα-δύο χρόνια ε, κυρίως ε, ε, αναφερθήκαμε στις βελτιώσεις ε, στην τεχνολογία, δεν ξέρω από εδώ ποιος κέρδισε, αλλά εν πάση περιπτώσει από πού προέρχονται τα πιο πολλά ατυχήματα από τις πολύ μεγάλες ταχύτητες και από την κατανάλωση αλκοόλ. Αλλά έχουμε, μιλάμε 40.000 νεκρούς κάθε χρόνο στην Ευρώπη. Ε, και στο τσουνάμι είπαμε ότι είχαμε 200.000 νεκρούς. Άρα τι σημαίνει αυτό ότι ουσιαστικά κάθε πέντε χρόνια στην Ευρώπη έχουμε τον ίδιο ε, ε, φόρο ζωή, νεκρούς δηλαδή από, αυτούς τους, από αυτές τις οδικές μεταφορές, από αυτές τις αιτίε. Άρα ε, λέμε ότι αφού υπάρχουν και συγκεκριμένοι περιορισμοί και στους δρόμους, ε, ίσως θα πρέπει να έχουμε και συγκεκριμένο όριο ταχύτητας και στους αυτοκινητοδρόμους. Ε, εντάξει, δεν έχουμε φτάσει μέχρι εκεί. Είπε ένα συνάδελφο εδώ, ούτε στο Αφγανιστάν έχει τέτοιο όριο ταχύτητα. Εντάξει. Εντάξει, δεν ξέρω ποια σχέση έχει τώρα το Αφγανιστάν με τη Γερμανία. σω είναι οι δύο χώρε, οι δύο μοναδικέ χώρε ε, στον κόσμο που δεν έχουν ανώτατο όριο ταχύτητα στου αυτοκινητοδρόμου. Η μόνη διαφορά ίσω που υπάρχει μεταξύ αυτών των δύο χωρών είναι ότι το Αφγανιστάν δεν έχει αυτοκινητοδρόμου. Εν πάση περιπτώσει, να βάλουμε ένα όριο. Ε, θα, θα είμαι πραγματικά ε, διαλλακτικό, θα πω 120-130 ε, χιλιόμετρα ανά ώρα. Εν πάση περιπτώσει, δεν αντιλαμβάνομαι γιατί να μην μπορούμε να κάνουμε κάτι τέτοιο εδώ. Μετά, σε ό,τι αφορά τις ε, μεταφορέ, μεταφορές, ε, το γνωρίζουμε και εμεί οι πράσινοι πως αν ε, έχουμε εδώ φιλοπεριβαλλοντική πολιτική μπορούμε να έχουμε μείωση και των σχετικών εκπομπών. το 8% λαμβάνει χώρα των μεταφορών λοιπόν στις θάλασσές μας, αλλά ένα σημαντικό ποσοστό από αυτό, το 80% δηλαδή από αυτό το 100%, ε, λαμβάνει χώρα στο ορεινό, αλλά μετά έχουμε και κάποια άλλα ποτάμια. Στον Εύα και ούτω Όπου όμω υπάρχουν πάρα πολλέ χώρε μέσα σε κάθε χρόνο 100 περίπου ημέρε όπου λόγω για παράδειγμα πλημμύρων ή οτιδήποτε άλλο δεν είναι δυνατό. υπάρχουν ε, προβλήματα σε ό,τι αφορά συγκεκριμένα δρομολόγια και γι' αυτό θα πρέπει να είμαστε σίγουροι και να λέμε ότι η εσωτερική ναυσιπλοεία ναι, μεν έχει κάποια πλεονεκτήματα, αλλά έχει και μειονεκτήματα. Υπάρχουν δηλαδή και κάποια προβλήματα. Τι σημαίνει αυτό, ότι αν θα κάνουμε επενδύσει ε, σε αυτές τις ε, πλωτέ γενικά μεταφορέ, θα πρέπει να είναι πολύ στοχοθετημένε. Θα κάνετε λοιπόν αυτό που καλείστε να κάνετε, να προωθήσετε την τη εσωτερική οδού ε, ναυσιμπλοεία. θα έχουμε για παράδειγμα δύο μικρά πλοία τα οποία θα προβαίνουν σε κάποιε μεταφορέ, θα πρέπει να έχουμε ένα τεράστιο project το οποίο θα υλοποιηθεί σε 20 χρόνια. Τώρα, οι ε, προσφυγέ κατά 22 χωρών από την πλευρά τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή επειδή δεν τήρησαν το συνδρομικό πακέτο. Είπαμε ε, ότι θα έχουμε εδώ αναθεωρημένο πακέτο, το RICAST, και αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχει ένα κράτο μέλο το οποίο θέλει να μπλοκάρει αυτή τη διαδικασία εσείς ως Προεδρεύον του Συμβουλίου θα υποστηρίξετε τον Επίτροπο ούτως ώστε να συνεχιστούν αυτές οι διαδικασίες κατά παράβαση. Γιατί μιλάμε ότι βρισκόμαστε σε ένα κράτος δικαίου στην Ευρώπη. Να μην υπάρχουν αυθαιρεσίες. Άρα λοιπόν ε, σας καλούμε να υποστηρίξετε τον Επίτροπο σε ό,τι αφορά την, ε, αυτές τις διαδικασίες. Ένα τελευταίο ζήτημα είναι ο θόρυβος. Έχουμε πει ότι ε, μπορούμε να ε, έχουμε μια τέτοια ε, ρύθμιση εδώ από την πλευρά τη Ευρώπη σε ό,τι αφορά δική μα χρηματοδότηση, μόνο σε εκείνο το σημείο. Άρα λοιπόν θα ήθελα να σα ρωτήσω, θα, θα θέλατε να υποστηρίξετε και το rolling stock, δηλαδή τη χρηματοδότηση ό,τι αφορά το θόρυβο και σε, σχέση με αυτό το τομέα. Γιατί. το να κάνουμε επένδυση σε κάποια άλλα, για παράδειγμα σε συστήματα απέδησης των αμοξοστοιχειών ή οτιδήποτε άλλο θα μπορούσαμε ναι, με, με καλύτερο τρόπο να επιτύχουμε ε, την ε, μείωση του θορύβου στις μεταφορές γενικά, πράγμα το οποίο είναι προς όφελός μας φυσικά. Συμφωνείτε με αυτό. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ τον κύριο Κράμερ και κύριο Ευχαριστώ Πρόεδρε. Τα συγχαρητηριά μου κύριε Υπουργέ για το πρόγραμμα που παρουσιάσατε. Πραγματικά ήταν μουσική για τα αυτιά μου. Αν κατορθώσετε να τα ελοποιήσετε όλα αυτά, καταπληκτικά. Και κυρίως ε, αναφέρουμε στα FABs, ε, στα λειτουργικά τμήματα ενεργείου χώρου. Θα ήθελα να τα καταφέρετε γιατί αυτό θα μας επέτρεπε να απλοποιήσουμε πάρα πολύ τη ζωή μας ε, και σε γλωσσικό επίπεδο. Τώρα, σε ό,τι αφορά την Ευρωβινιέτα, θεωρώ ότι είναι πολύ καλό το ότι θέσατε αυτό το σημείο στην ημερική διάταξη. Εγώ όπως και άλλοι συνάδελφοι το δήλωσαν, ε, θα ήθελα να συνεχίσουμε τη συζήτηση επί του θέματος αυτό. Ε, θα έπρεπε να συζητήσουμε το θέμα αυτό και σε τεχνικό επίπεδο, όχι μόνο σε πολιτικό επίπεδο. Εγώ θέλω να σας θέσω μια ερώτηση για την Ευρωβινιέτα. Αν βάλετε την Ευρωβινιέτα στην υπηρεσία διάταξη, τι θα κάνετε με τα εφιστάμενα συστήματα στις διάφορες χώρες, δηλαδή τα συστήματα των διοδίων σε Γαλλία και Ιταλία. Οι κατοχώρες εισήγαγαν μόλις ε, ένα σύστημα ε, συγκεκριμένων τελών. Τι θα κάνετε λοιπόν ε, σε σχέση με την Ευρωβινιέτα. Εγώ θα ήθελα πάρα πολύ να καταργήσουμε όλα αυτά τα διαφορετικά συστήματα γιατί πραγματικά είναι πάρα πολύ δύσκολη η κατάσταση. Ο Χρήστος τώρα πρέπει να αντιμετωπίσει 27 διαφορετικά συστήματα. Τι σκέφτεστε. Επίσης, κύριε Υπουργέ, χαίρομαι πάρα πολύ που βλέπω ότι ε, δίνεται και προσοχή στις ε, εσωτερικές πλωτές ε, οδούς. Ο κύριος Κράμερ Αναφέρθηκε ιδίω στους σιδηροδρόμους, όμως ε, θα πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη ότι πάνω από το 60% των ε, μεταφορών γίνεται από μικρά σκάφη των 150 ε, τόνων. Έτσι λοιπόν, ε, μήπως ε, θα πρέπει να σκεφτούμε και το σύστημα Μάρκο Πόλο. Υπάρχει ένα σύστημα Μάρκο Πόλο για την πρόθεση τη εσωτερική ναυσιπλοεία, αλλά το σύστημα αυτό δεν μπορεί να λειτουργήσει στην πραγματικότητα, γιατί πραγματικά η γραφειοκρατία είναι τεράστια. Και αν θέλετε να βελτιώσετε την αποτελεσματικότητα θα έπρεπε να πλουστεύσετε το σύστημα Μαρκοπόλου, να γίνει πιο προσβάσιμο. Έτσι λοιπόν, τι θέλω να σας ζητήσω κύριε Υπουργέ, να εξετάσετε αυτό το σύστημα Μαρκοπόλου και να προωθήσετε την απλούστευσή του. Υπάρχει και κάτι άλλο για το οποίο θέλω να σας ρωτήσω για τις οδικές μεταφορές. Κάποιος από τους συναδελφούς ε, συνέταξε μια εξαιρετική έκθεση σε ό,τι αφορά τα πρόστιμα και τις παραβάσεις, τις οδικές παραβάσεις και Ξέρετε ότι τα συστήματα στις οδικές μεταφορές διαφέρουν ε, τα μάλλα από χώρα σε χώρα μπορεί κάποιος να χρειαστεί να πληρώσει 180 ευρώ πρόστιμο στην Ιταλία, ενώ στη Γαλλία μπορεί να πρέπει ακόμη και να φλεξτεί για ένα έτος το άτομο και να πληρώσει 30.000 ευρώ. Έτσι λοιπόν θα πρέπει ε, ουσιαστικά να προβούμε σε κάποια προσέγγιση των ε, προστήμων για τις ίδιες παραβάσεις ε, θα ήθελα να ασχοληθείτε και με αυτό το θέμα. Επίσης να σας ευχηθώ κάθε επιτυχία. Το, σε ό,τι αφορά τώρα το θέμα της εσωτερικής νευσιπλοείας, σας εμπιστεύομαι σίγουροι ότι θα είναι πολύ καλά τα αποτελέσματα της Βελγικής Προεδρίας. Πρόεδρος. Βλέπετε ότι εν γέννη είναι πολύ θετικά αποδεκτές οι προτάσεις σας, συμμερίζονται οι συνάδελφοι της ανησυχίας σας. Έτσι λοιπόν ε, θα προτείνουμε και αυτό το ε, θέμα στους συντονιστές, όμως ε, μας περιορίζει ο χρόνος. Μόνο λοιπόν, θα σας δώσω το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ομαδοποιήσω, αν μου επιτρέπετε, τις απαντήσεις με βάση τα έξι πακέτα που σας ανάφερα στην εισαγωγή μου. Καταρχήν, η φιλοδοξία μας σύντομα να γίνει συζήτηση για τη Λευκή Βίβλο. Ξέρετε καλά ότι η Κομισιόν επιθυμεί να ξεκινήσει η συζήτηση στο Συμβούλιο του Δεκεμβρίου. Είναι λίγο αργά. Θεωρώ ότι μας συμφέρει στο εξάμεινο αυτό να έχουμε και ανταλλαγή απόψεων στο Συμβούλιο αλλά και συζήτηση με την Κομισιόν για τις προσαρμογές που θα πρέπει να γίνουν έτσι ώστε στη φάση της πρώτης ανταλλαγής απόψεων να ληφθούν υπόψη και μετά να ληφθούν υπόψη διάφορες αλλαγές. Συνεχίζω στα, στα φλαμαδικά. Περίπου ένα χρόνο πριν ξεκίνησε η προετοιμασία της Λευκής Βίβλου. Θεωρώ ότι θα πρέπει να είναι δυνατόν το Δεκέμβριο ακόμα και αν δεν έχουμε ένα τελικό κείμενο, έστω ένα έγγραφο εργασίας με τα βασικά στοιχεία, πιστεύω ότι ήδη το Δεκέμβριο θα υπάρχει δυνατότητα να γίνει μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων για να ληφθεί απόφαση μέχρι το τέλος του μηνός. Όχι για να πούμε μετά «Α, η Βελγική Προεδρία τα κατάφερε». Όχι, διότι πιστεύω ότι το περιεχόμενο της Λευκής Βίβλου πρέπει να καλύπτει όλες τις μεγάλες ιδέες του τι πρέπει να γίνει τα επόμενα χρόνια για την κινητικότητα. Η λευκή αυτή βίβλος θα ορίζει τον τρόπο συμπεριφοράς του επιτευκταίους στόχους για τα επόμενα χρόνια. Θα είναι ένα είδος σύνταγμα όλων των νομοθετικών και άλλων μέτρων που πρέπει να ληφθούν για να έχουμε μια βιωσιμότητα στις μεταφορές. Σε θέματα ασφάλειας, όλες οι θεμελιώδεις ιδέες αυτές πρέπει να εμπεριέχονται στη Λευκή Βίβλο. Θα είναι γελίο να εξακολουθούμε να συζητάμε, να μιλάμε για τη Λευκή Βίβλο, ότι είναι τόσο σημαντικό για τις μεταφορές, για την κινητικότητα και η απέξω να τα βλέπουν όλα αυτά, να ξέρουν ότι αφορά την περίοδο 2010-2020 και να δημοσιευτεί με καθυστέρηση ας πούμε το 12. Επιβάλλεται λοιπόν να ξεκινήσουμε αμέσως αυτή τη δουλειά. Δεύτερον, η, το ευρωσήμα, το αυτοκόλλητο. Όλοι μιλήσατε γι' αυτό. Πολύ μάλλον μιλήσατε γι' αυτό είπατε ότι είναι μια ιδέα η οποία αξίζει να προωθηθεί. Σας ομολογώ ότι πολλές φορές σκέφτηκα το θέμα αυτό πριν αποφασίσω να πω κάτι για το ευρωσήμα αυτό. Πολλοί στο Συμβούλιο, μάλλον υπάρχουν στο Συμβούλιο πολλές διαφορετικές θέσεις. Ανάλογα με το ποια χώρα μιλάει. Εγώ προσωπικά θεωρώ ότι και στο Κοινοβούλιο υπάρχουν διαφορετικές απόψεις για το θέμα αυτό. Για το Ευρωσήμα υπάρχουν πολλές εθνικές θέσεις και γι' αυτό είναι δύσκολο να καταλήξουμε σε ομόφωνη θέση. Ωστόσο, Επίσης θεωρώ ότι πρέπει η φιλοδοξία μας να είναι να κάνουμε μια πρόταση. Νομίζω ο κύριος Κράμερ είπε ότι πρέπει να βιαστούμε. Πρέπει να βιαστούμε. Ο χρόνος τρέχει. Εγώ νομίζω ότι δεν πρέπει να βιαστούμε για ένα τέτοιο θέμα. Θα ήταν επικίνδυνο. Υπάρχει κίνδυνος να μπερδικλωθούμε στις ιδέες μας και να πέσουμε. Θεωρώ ότι πρέπει να γίνει μια συζήτηση και μάλλον θα γίνει αυτή η συζήτηση μέχρι το τέλος του χρόνου. Καταρχήν όλοι οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αναλύσουν το θέμα αυτό από όλες τις πλευρές. Υπάρχουν, υπάρχει μια ομάδα εργασίας που μόλις τώρα ξεκίνησε τη δουλειά της για το πολύ πολύ λεπτό αυτό θέμα. Ας περιμένουμε να δούμε τι πορίσματα θα βγουν από την ομάδα αυτή εργασίας. Ελπίζω να είμαστε έτοιμοι τον Οκτώβριο ας πούμε. Εν πάση περιπτώσει, αν έχουμε υλικό, το μπορούμε να το συζητήσουμε έστω άτυπα, ας πούμε από τον Οκτώβριο και μετά. Επαναλαμβάνω για το θέμα αυτό υπάρχουν πολλές διαφορετικές θέσεις. Υπάρχουν οι θέσεις των περιφερειακών, περιφερικών χωρών και οι θέσεις χωρών που βρίσκονται στο κέντρο της Ένωσης. Εδώ ήδη έχω μια μεγάλη διαφορά. Έπειτα, σε ορισμένε από αυτέ τι χώρε υπάρχει ήδη ένα εθνικό σύστημα. Οι χώρε αυτέ θέλουν να το κρατήσουν. Δεν θέλουν να απορροφηθούν σε μέσα σε ένα γενικευμένο ευρωπαϊκό σύστημα. Και αυτό είναι που δυσκολεύει τα πράγματα για όλους μας. Δεν θέλω να προδικάσω τα πορίσματα της ομάδας εργασίας. Πιστεύω όμως ότι για το ευρωσήμα θα πρέπει να κάνουμε διάκριση μεταξύ της καταπολέμησης του θορύβου, της ρήπανσης αφενός και αφετέρου της χρήσης των υποδο... της υποδομής. Με τον α ή το β τρόπο υπάρχει κίνδυνος να τα ανακατέψουμε όλα αυτά τα θέματα. Ενώ τα θέματα αυτά συνήθως είναι διαφορετικά το ένα από το άλλο. Πρέπει λοιπόν να κάνουμε αυτή την διάκριση και να λάβουμε υπόψη μας τις ευαισθησίες που υπάρχουν στο θέμα αυτό. Μερικοί συντονιστές σωστά επέστησαν την προσοχή μας στο ότι η χρηματοδότηση και η χρήση των εισόδων αυτών είναι ένα σημαντικό δεδομένο. Αν κάνουμε τη διάκριση λοιπόν, σαφή διάκριση όμως, μεταξύ των υποδομών αφενός, συμφόρηση στην κυκλοφορία αφενός, αφετέρου την καταπολέμηση της ρήπανσης και του θορύβου, αν κάνουμε αυτή τη διάκριση, είναι πιο εύκολο τότε να δούμε πώς θα χρησιμοποιήσουμε τα χρήματα αυτά και έτσι πιο εύκολα να βρούμε μια πολιτική λύση. Δεν θέλουμε να δυσκολέψουμε τη ζωή κανενός δημοσιονομικά. Το να επιμερίσουμε λοιπόν το πρόβλημα σε δύο κατηγορίες θα μας βοηθήσει. Αναφέρθηκε ο αγγλικός όρος earmarking, να οριστεί πού θα πάνε κάθε φορά τα συγκεκριμένα κονδύλια. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Πολλοί από εσά το είπατε το θέμα αυτό της χρηματοδότησης είναι σημαντικό. Εγώ από τη μεριά μου θα προτιμούσα να έχουμε έσοδα πάνω κάτω με αυτά που έχουμε σήμερα μεν αλλά η στάθμιση των επιμέρους παραμέτρων που ανάφερα που πρέπει να ενυπάρχουν στο ευρωσήμα αυτό να αλλάξει. Δηλαδή να λάβουμε υπόψη τα επιμέρους στοιχεία τα οποία ανάφερα πριν έτσι ώστε τελικά να ικανοποιηθούν όλοι χωρίς να στοιχίζει όλη αυτή η ιστορία πιο ακριβά στο χρήστη. Μια τέτοια διαδικασία νομίζω θα καθησυχάσει όλες τις χώρες όσον αφορά το θέμα του προϋπολογισμού. Θέλουμε να πετύχουμε τη μέγιστη δυνατή εναρμόνιση στις μεταφορές. Φυσικά όμως αυτό θα πρέπει να γίνεται λογικά. Τα χρήματα που θα προέρχονται από τις μεταφορές να επανεπενδύονται στις μεταφορές και όχι αλλού. Θα επανέλθω εξάλλου στο θέμα αυτό. Για να δούμε τώρα κάτι άλλο. Την ασφάλεια. Και το μνημόνιο που θα δημοσιευτεί για τους στόχους ασφάλειας. Με το προηγούμενο δεκαετές πρόγραμμα δράσης είχαμε στόχο τη μείωση κατά 50% του αριθμού των θυμάτων. Ας δούμε τι έγινε απολογισμό του 2009. Μερικές χώρες που είχαν αρνητικές στατιστικές στο παρελθόν βελτιώθηκαν. Και στο τέλος του 2009 συνολικά θα έχουμε μια βελτίωση περίπου 36% σε σχέση με τη γενική κατάσταση και πιο συγκεκριμένα στις οδικές μεταφορές. Ελπίζω στο τέλος του 2010 η βελτίωση να είναι 40%. Θα πρέπει ο στόχος μας να παραμένει το 50%. Το πιο σημαντικό όμως είναι ότι βλέπουμε ότι υπάρχει πολιτική βούληση υπέρ αυτής της μείωσης των δυστυχημάτων και των, των ατυχημάτων συγγνώμη, και των θυμάτων. Πάση όποια και να είναι τα νούμερα, αυτό που έχει σημασία είναι να υπάρχει πολιτική βούληξη. Δεν ξέρω ποιο θα είναι ο στόχο για την περίοδο 2010 2010-2020 Θα είναι το 50%. Γιατί όχι. Αυτό που έχει σημασία όμω είναι ο αριθμό των ατυχημάτων, των νεκρών και των βαρέως τραυματισμένων να μειωθεί αρκετά. Η τάση είναι σημαντική, όχι τόσο το συγκεκριμένο νούμερο. Βέβαια, οι στατιστικές και οι συγκρίσεις μεταξύ των διαφόρων χωρών είναι ένα δεδομένο και μάλιστα ενδιαφέρον. Το επόμενο πρόγραμμα δράσης θα πρέπει να εμπεριέχει μία πολύ σημαντική παράμετρο για προστασία των ασθενών χρηστών. Στο παρελθόν αναφερόμασταν κυρίως στους οδηγούς ταχύτητα, κατανάλωση φαρμάκων ή νοπνευματοδών, τήρηση των φανοστατών, το κόκκινο, τα διάφορα μέτρα ασφαλείας, όρια ταχύτητας κλπ. Όλα αυτά αφορούν τον οδηγό. Όπως το βλέπουμε εμείς το πρόβλημα, εμείς θα θέλαμε επίσης να ασχοληθούμε και με τα συνθήματα, τα παράλληλα θύματα των ατυχημάτων αυτών δηλαδή την προστασία των χριστών, των ασθενών χριστών όπως τους λέμε, δηλαδή μέτρα που και αυτά επαναλαμβάνω θα πρέπει να υπάρχουν στη Λευκή Βίβλο για τα άτομα αυτά. Τώρα για τα διασυνοριακά μέτρα μεταφορές μεταφορών. Η σημερινή κατάσταση διέπεται από ένα έντονο εθνικό στοιχείο στις περιοχές εκατέρωθεν των συνόρων. Χρειάζεται συνεργασία όσον αφορά τον έλεγχο στις μεταφορές. Πολύ συχνά αυτό στηρίζεται σε διμερή μέτρα, σε καλό κλίμα μεταξύ αστυνομίας και λοιπά μεταξύ των αρχών δεν είναι μέτρα της Ένωσης που θα πρέπει όμως να υπάρχουν και να εφαρμόζονται αυτόματα. Να μην είναι δηλαδή διμερεί και περιορισμένα μόνο στις δύο τοπικές αστυνομίες. Αν θέλουμε να ακολουθήσουμε αυτή την πιο εναρμονισμένη μέθοδο, καταρχήν θα έχουμε προβλήματα. Προβλήματα στις θέματα της δικαιοσύνης και εσωτερικών πιο αποτελεσματικούς ελέγχους, ιδιαίτερα στις οδικές μεταφορές, σε χώρες όπου το... υπάρχει πάρα πολλή κίνηση transit, υπάρχουν πάρα πολλά φορτηγά με ξένες πινακίδες, συχνά διαπιστώνουμε ότι η έλεγχη δεν είναι αποτελεσματική και οι ποινές και οι κυρώσεις είναι ανεπαρκείς και δύσκολοι. και από εκεί και πέρα επιθυμούμε να μην εργάζονται οι χώρες σε διμερή βάση. Θα πρέπει να έχουμε ένα αυτοπροματοποιημένο σύστημα πληροφόρησης σε ευρωπαϊκό επίπεδο και αυτό σημαίνει, λόγω χάρη, τη βαλκική αστυνομία πρέπει να μπορεί να ποινικοποιήσει κάποιο που έρχεται από την Πολωνία και που χρησιμοποιεί στο Βέλγιο την πολωνική του πενική, πινακίδα ή ε, δεν θα έπρεπε να παρεμβαίνει η βελγική δικαιοσύνη. Δεν είναι αυτό βέβαια το θέμα που θέλω να συζητήσω εδώ. Το... Ο στόχος του εναρμονισμένου συστήματος θα είναι να ταυτοποιήσουμε όποιον έχει κάνει την παράβαση και να μπορούμε να λάβουμε και μέτρα για να τον τιμωρήσουμε. Όσοι παρακολούθησαν από κοντά αυτή την υπόθεση, γνωρίζουν ότι ήδη έχουμε συζητήσει πάρα πολύ το θέμα της νομικής βάσης. Ε, Κάποιο είπε κάποια μέρα ότι δεν με ενδιαφέρει αν είναι μαύρη ασπριγάτα, με ενδιαφέρει αν πιάνει ποντίκια. Έτσι λοιπόν, αυτό που μας ενδιαφέρει και μας είναι να εφαρμοστεί αποτελεσματικός έλεγχος. Πρέπει να εφαρμοστεί. Όσοι λοιπόν ε, προβαίνουν σε παρεμβάσει ε, θα πρέπει να ανακαλούνται στην τάξη και θα πρέπει και να τιμωρούνται. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να το δούμε εις βάθος αργότερα. Νομίζω ότι μου θέσατε και μια ερώτηση που έχει να κάνει με το εξής. Για το θέμα της κινητικότητας. Έχουμε ε, τις ε, χώρες ε, όπου υπάρχει ένα σύστημα εσωτερικής ναυσιπλοείας που λειτουργεί καλά. Όμως ό,τι αφορά το θέμα της διατροπικότητας, νομίζω ότι θα πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη σημασία στο οικονομικό και στο περιβαλλοντικό επίπεδο, αλλά και δεύτερον θα πρέπει να δούμε και την εσωτερική ναυσιπλοεία και να βελτιώσουμε τις συνδέσεις μεταξύ της θάλασσας και του εσωτερικού της χώρας με μεγαλύτερη χρησιμοποίηση της εσωτερικής ναυσιπλοείας. Όλα αυτά θα πρέπει όμως να τα αναπτύξουμε με ισορροπημένο τρόπο και θα πρέπει να δημιουργήσουμε και συνδέσμους μεταξύ των θαλάσσιων μεταφορών και, των, και της εσωτερικής ναυσιπλοείας. Θα πρέπει όλα αυτά να τα οργανώσουμε και σε τεχνικό αλλά και σε διοικητικό επίπεδο. Να υλοποιήσουμε τις ε, μπλε οδούς, blue lanes. Αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Σε ό,τι αφορά τώρα τις ε, ενέργειες μεταφορές, πιστεύουμε ότι έχουν ε, γίνει κάποιες πολύ σημαντικές ε, πρωτοβουλίες με τη δημιουργία του FABEX, με τη στενή συνεργασία μεταξύ στρατιωτικής και πολιτικής αεροπορίας για να μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε με καλύτερο τρόπο τους αεροδιαδρόμους. Θέλουμε να μειώσουμε την ε, χρήση της κυροζήνης, να αποφεύγεται να γίνονται παρακάμψεις από τα αεροσκάφη και θα πρέπει να προωθήσουμε και αυτό το ζήτημα εξίσου. Θα ήθελα τώρα να αναφερθώ σε κάποια συγκεκριμένα σημεία. Διεθνοποίηση, συγγνώμη, εσωτερικοποίηση του εξωτερικού κόστους. Ο κύριος Κρός αναφέρθηκε στην αναγκαιότητα να υπάρχει επιμερισμός του άχθους μεταξύ των διάφορων τρόπων μεταφοράς. Σε ό,τι διαφορά λοιπόν αυτό το εξωτερικό κόστος ε, πώς θα γίνει η δυνοποίηση θα πρέπει ουσιαστικά να έχουμε ένα level playing field ε, θα πρέπει οι κανόνες του ανταγωνισμού να είναι οι ίδιοι κάτι που δεν ισχύει σήμερα. ξέρω ότι δεν θα μπορέσουμε να έχουμε αμέσως ικανοποιητικό αποτέλεσμα. Παρ' όλα αυτά νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε μια προσπάθεια για να σημειώσουμε πρόοδο στον τομέα αυτό. Σε ό,τι αφορά τώρα την πηγή εσόδων για τα κρατημέλη, να έχετε δίκιο κύριε Κρός. Κατάλαβα τι θέλατε να πείτε. Και μάλιστα το είπατε σχετίζονται φυσικά και με τα διευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών. Υπάρχουν διασυνοριακά έργα, διασυνοριακά project, ε, τα οποία σήμερα δεν λαμβάνουν την απαραίτητη προσοχή σε εθνικό επίπεδο. Και Φυσικά θα έπρεπε να συνεισφέρει και η Ευρωπαϊκή Ένωση στο να, εξεύρουν, να εξευρεθούν καλύτεροι τρόποι και πηγές χρηματοδότησης. Εμείς από το Συμβούλιο και με το Κοινοβούλιο θα πρέπει να δούμε με ποια μέσα θα μπορέσουμε να καλύψουμε τα κενά, τους κρίκους που λείπουν για να χρηματοδοτήσουμε αυτά τα τμήματα των δικτυών που λείπουν ακόμη σε διασυνοριακό επίπεδο και επίσης θα πρέπει να βελτιώσουμε και την ποιότητα των υποδομών ανεξαρτήτως του τρόπου μεταφοράς. Θα πρέπει να υπάρξει και ισορροπία στο θέμα αυτό. Μιλήσαμε για το earmarking και τη δέσμευση των πόρων επανειλημμένος, όμως εγώ νομίζω ότι εδώ δεν μπορούμε να έχουμε αποτελέσματα μαύρα ή άσπρα. Θα πρέπει να βρούμε και μια σωστή απόχρωση του γκρι. Αναλόγως και με τις προτεραιότητες που πρέπει να γίνουν σεβαστές. Εγώ προσωπικά θεωρώ ότι θα πρέπει να υπάρχει τρόπος να οργανώσουμε αποτελεσματικά αυτή τη χρηματοδότηση ό,τι αφορά τώρα την ασφάλεια και πιο συγκεκριμένα την ασφάλεια των αερολιμένων. Γνωρίζετε ότι προσπαθούμε να αναπτύξουμε μία ευρωπαϊκή προσέγγιση, μια καθολική προσέγγιση σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Κάποια κράτη-μέλη έχουν ε, ουσιαστικά προχωρήσει στο θέμα αυτό και ελπίζω τελικά να καταλήξουμε σε μια κοινή θέση. Ελπίζω ότι όλα αυτά θα μπορέσουν να γίνουν κατά τη διάρκεια των επόμενων τεσσάρων μηνών. Ελπίζω να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε, να καταθέσουμε μία πρόταση που να δρομολογηθεί. Σε ό,τι αφορά τώρα την οδική ασφάλεια και το πολιτές πρόγραμμα, αναφέρθηκα σε αυτό. Πιστεύω ότι ακόμη και αν υπάρχει αν δούμε ότι η μείωση του 50% για το 2001-2010 δεν είναι δυνατή, θα πρέπει και πάλι να θέσουμε τον πύχη ψηλά και τα 27 κράτη-μέλη, η πολιτική των 27 κρατών μελών θα πρέπει να δηλώσουν ότι επιθυμούν σφόδρα να εργαστούν για την υλοποίηση του στόχου αυτού. Όχι μόνο για ηθικούς λόγους, αλλά και για να καταπολεμήσουμε όλες αυτές τις αρνητικές συνέπειες ε, για χιλιάδες ανθρώπους. Υπάρχει και κόστος ε, που σχετίζεται με αυτά τα ατυχήματα. Θα πρέπει να εργαστούμε όλοι μαζί. Κάποιες χώρες μας έχουν δείξει ότι υπάρχουν δυνατότητες βελτίωσης και πρόοδου μέσω των βέλτιστων πρακτικών και μέσω των συγκρίσεων που πρέπει να γίνουν και μέσω του benchmarking. Θα πρέπει λοιπόν θα πρέπει να εμπνευστούμε ένα από τον άλλο για να καταλήξουμε σε καλά αποτελέσματα. Τώρα, για τις θαλάσσιες μεταφορές. και πιο συγκεκριμένα συνεργασία μεταξύ των διάφορων τρόπων μεταφοράς. Εγώ ξέρω ότι η ΜΕΝ είναι υπέρ των συνδεδρόμων περισσότερο, η ΔΕ υπέρ των οδικών μεταφορών. Θα πρέπει όμως να μπορούμε να αναγνωρίσουμε ότι κάθε τρόπος μεταφοράς ε, έχει τα δικά του πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. Γνωρίζουμε ότι η ιστορική ναυσιπλοεία από οικονομική και οικολογική σκοπιά έχει πολλά πλεονεκτήματα. Γνωρίζουμε επίσης ότι υπάρχει το εξή πρόβλημα με την ιστορική ναυσιπλοεία, ότι χρειάζεται περισσότερο χρόνο για τις μεταφορές. Επίσης, ε, τα δίκτυα αυτά δεν είναι πολύ αναπτυγμένα. Αυτά είναι μενοκτήματα που πρέπει να τα αναγνωρίσουμε. Σε σχέση με την εσωτερική νευσιπλοεία, ξέρουμε ότι η σιδηρόδρομη είναι πολύ πιο γρήγορη. Το σιδηροδρομικό δίκτυο είναι ήδη πολύ πιο πυκνό. Και από την άλλη γνωρίζουμε ότι το σιδηροδρομικό δίκτυο δεν είναι πάντοτε τόσο ευέλικτο όπως ε, οι οδικές μεταφορές λόγου χάρη. οδικέ μεταφορές που μέρα με την ημέρα μπορούν να εξελιχθούν και φυσικά καθώς είναι πιο, δυνα... πιο προσαρμόσιμες υποστηρίζουν και την ανάπτυξη των υπόλοιπων τρόπων μεταφορά. Παρίσι, Παραδείγματο χάρη, η κολονία σε μια μέρα, δεν τη οδική οδού μπορεί να φτάσει κάποιο πολύ εύκολα, αλλά εμεί ε, θέλουμε ουσιαστικά να εξισορροπήσουμε τη χρήση των διάφορων τρόπων μεταφορά, έτσι ώστε κάθε φορά να μπορεί κανεί να προσφύγει στον τρόπο μεταφορά που ανταποκρίνεται καλύτερα στι κοινωνικέ, περιβαλλοντικέ και οικονομικέ του ανάγκε. Είναι του περιβάλλοντος. Το περιβάλλον είναι ζωτική σημασία στο πλαίσιο αυτό. Δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Κύριε Καντράουι. Θα πρέπει φυσικά η φιλοδοξία μας να είναι να επιταχύνουμε τη δημοσίευση της Λευκής Βίβλου για την οδηγία για την Ευρωβινιέτα αναφερθήκατε κι εσείς. Θα πρέπει να υπάρξει απελευθέρωση από τα κράτη-μέλη. Σίγουρα θα χρειαστούμε αυτούς τους πρόσθετους πόρους, όμως το εγχείρημα αυτό θα πρέπει να ξεκινήσει από την αρχή ότι το συνολικό άχθος δεν μπορεί να βελτιωθεί. Αν οι Υπουργοί Οικονομικών ε, βρουν ε, ένα κονδύλι που δεν χρησιμοποιείται για τις μεταφορές, αυτοί θα δουν σε τι μπορεί να χρησιμοποιηθεί αυτό το κονδύλι. Όμως εμείς πρέπει να υποστηρίξουμε το δικό μας ε, τομέα και πρέπει να ζητήσουμε να υπάρχει μεγαλύτερη ισορροπία μεταξύ των διάφορων τρόπων μεταφοράς και να χρησιμοποιούνται σωστά τα κονδύλια. Τώρα, την άπτυξη των ευρωπαϊκών δικτύων μεταφοράς. Όπως ε, σωστά είπατε, υπάρχουν περιορισμοί και εδώ τίθεται το θέμα της χρηματοδότησης, όπως ε, είπα και για τους σιδηροδρόμους ε, και για τις οδικές μεταφορές. Το να καθορίσουμε αυτή τη χρηματοδότηση θα είναι ένα εγχείρημα εξέβρεση ισορροπίας μεταξύ Συμβουλίου και Κομισιόν και ελπίζω και με την έγκριση του Κοινοβουλίου. Και στο πλαίσιο αυτού του εγχειρήματος θα πρέπει να σκεφτούμε τις τεχνικές ε, ιδιαιτερότητες, ε, τις τεχνικές προδιαγραφές του κάθε τομέα. Κυρίως για τους σιδηροδρόμους, όπως είπατε. Κάποια άλλη στιγμή, όχι σήμερα, έχουμε μιλήσει για τα ε, δίκτυα τα ηλεκτρικά που υπάρχουν στις διάφορες χώρες. Ε, είναι σημαντικό πέρα από την οικολογία, πέρα από το περιβάλλον, να δώσουμε έμφαση και στην ασφάλεια. Αν θέλουμε να δράσουμε βρεχυπρόθεσμα, θα πρέπει πρέπει η ασφάλεια να τεθεί ως προτεραιότητα. Είναι θεμελιώδους σημασίας και θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να επιμείνει στην τεχνική εναρμόνιση για να υπάρχει ασφάλεια αυτή. Η ανάπτυξη λοιπόν των υποδομών είναι κάτι σημαντικό. Και κατόπιν μιλώντας από τεχνική σκοπιά, η ανάπτυξη των δικτύων θα πρέπει να γίνει λογικά εύκολα, αλλά ποτέ δεν πρέπει να ξεχνάμε την ασφάλεια. Θα πρέπει να πάμε πολύ πιο πέρα από ό,τι έχουμε κάνει σήμερα. Σε ό,τι αφορά την αναδιατύπωση τώρα τη πρώτη δέσμη μέτρων για τους σιδηροδρόμους, Εν τω μεταξύ, είδαμε ότι υπάρχουν αρκετέ αρνητικέ αντιδράσει έναντι του δεύτερου πακέτου. Έτσι, λοιπόν, στο εσωτερικό του Συμβουλίου θα πρέπει να υλοποιήσουμε μια αρκετά διαφανή συζήτηση για τις ε, φιλοδοξίες ε, της Κομισιόν και Επίσης ε, θα πρέπει να δούμε και τι είναι έτοιμες να πράξουν οι διάφορες χώρες λαμβάνοντας υπόψη την πραγματικότητα στο σιδηρομικό τομέα και λαμβάνοντας υπόψη και το ρόλο του κάθε εθνικού συνδρομικού οργανισμού. Δεν έχει κανένα νόημα να έχουμε κάτι άριστο στο χαρτί αν δεν υπάρχει στη χώρα πολιτική βούληση και δεν ε, υπάρχουν και οι πόροι να τέθουν σε εφαρμογή τα όσα θα λέγονται στο χαρτί. Πιστεύω ότι είναι σημαντικό σε ό,τι αφορά το συνδυνομικό πακέτο να μπορέσουμε στο Συμβούλιο να έχουμε μία ανοιχτή και επικοδομητική και ειλικρινή συζήτηση. Ελπίζω ότι σε κάποιους μήνες θα μπορέσουμε να παρουσιάσουμε σχετικές προτάσεις. Και επίσης ελπίζω ότι οι διάφορες εθνικές αρχές θα έχουν επικοδομητική στάση. Θα ήθελα να αναφερθώ τώρα στην ε, επιβολή των κυρώσεων σε περίπτωση που έχουμε δύο συνολογικές παραβάσεις. Πολύ το αναφέρατε αυτό. Αναφερθήκατε και σε ε, διαφορετικά ποσά σε ό,τι αφορά τα πρόστιμα. Αναφέρατε τη Γαλλία, παραδείγματο χάρη, και κάποια χώρα της Βαλτικής. Κοιτάξτε, το σημαντικό είναι ότι όταν υπάρχει παράβαση, πέρα από το ποσό που επιβάλλεται από την εθνική νομοθεσία, να μπορεί να επιβληθεί αυτή η κύρωση. Εμένα με ενδιαφέρει καταρχήν να υπάρχει εναρμόνιση και εφαρμογή σε όλα τα επίπεδα. Τώρα αν θέλουμε όλοι να τα κάνουμε άπαξ, τελικά μάλλον διακινδυνεύουμε το να μην έχουμε κανένα αποτέλεσμα. Πιστεύω για το ημετοφάμπεκ θα μπορούσαμε να προχωρήσουμε πολύ γρήγορα Βέβαια δεν μπορώ παρά να μιλήσω για την περιοχή που μας, ε, την περιφέρεια αυτή που μας αφορά εμάς ως Βέλγιο, Μπενελούξ, Γαλλία, Γερμανία, Ελβετία και νομίζω ότι έτσι μπορούμε να διαχειριστούμε καλύτερα τον ενέργειο χώρο και ελπίζω ότι το ίδιο θα ισχύει και για τις υπόλοιπες περιφέρειες. Πραγματικά Είμαι πεπισμένος ότι πρόθεσμα θα μπορέσουμε να προβούμε σε σημαντικές βελτιώσεις. Κυρίως ε, σε ό,τι φορά τώρα τους επιβάτες. Για τα λεωφορεία, τους επιβάτες των λεωφορείων. Εδώ θα ήθελα να σταθώ στο εξής ξέρετε ότι οι μεταφορές ε, με τα λεωφορεία για τις μακρές αποστάσεις, για μεγάλες αποστάσεις, είναι ο φτηνότερος τρόπος μεταφοράς. Αν ε, τώρα θέλουμε λοιπόν να συμπληρώσουμε εδώ τους κανόνες, θα πρέπει να κατανοήσουμε ότι αν θέλουμε πιο αυστηρή νομοθεσία, θα πρέπει αυτό να έχει επίπτωση και στις τιμές. Αυτό είναι προσπέλαστο. Έτσι λοιπόν θα πρέπει να υπολογίσουμε και να γνωρίζουμε ότι στο υφιστάμενο σχέδιο, ο τομέας που αντέδρασε πρώτος ήταν οι σιδηρόδρομοι, γιατί οι σιδηρόδρομοι ε, ανταγωνίζονται τα λεωφορεία σε εθνικό επίπεδο και ο τομέας των σιδηροδρόμων με ρώτησε μάλιστα γιατί έχουμε μεγαλύτερο ρυθμό επιβατών σε σχέση με τα λεωφορεία. Υπάρχει πρόβλημα ανταγωνισμού. Αυτό θα πρέπει να το έχουμε κατά νου. Δηλαδή, ότι τα δικαιώματα των επιβατών σε ό,τι αφορά τι ενέργειε μεταφορέ, παραδείγματο χάρη, εκεί είναι πιο κατανοητά τα πράγματα. Όμω, να σα πω ότι για ε, τι μεγάλε εταιρείε, κυρίω τι μεγάλε αεροπορικέ εταιρείε, δεν μπορούμε να βρεθούμε σε μια κατάσταση που θα έχει ως αποτέλεσμα ο παγκόσμιος ανταγωνισμός με τα μέτρα που θα πάρουμε εμείς να έχει αντίκτυπο στον ανταγωνισμό, δηλαδή οι δικές μας εταιρείες να είναι λιγότερο ανταγωνιστικές ε, στη διεθνή σκηνή. Αν οι κανόνες μας είναι υπερβολικά αυστηροί, θα πρέπει να έχουμε κατά νου ότι θα έχουμε πρόβλημα ανταγωνιστικότητα. Λοιπόν, Λευκή Βίβλο, όλα αυτά τα συζητήσαμε, εσωτερική νευσιπλοεία και να περάσω στα γαλλικά. Για τα ευρωπαϊκά δίκτυα μιλήσαμε. Τώρα για τον κόλπο του Μεξικού. Ε, εντάξει, δεν θέλω να έρθω εδώ σε αντιπαράθεση με συνάδελφου που είναι αρμόδιοι για, τον, για την προστασία του περιβάλλοντος. Εάν υπάρξουν προβλήματα για τι ναυτιλιακές μεταφορέ, ε, προφανώ και θα παρέμβω εκεί. Αλλά εάν δεν συμβεί κάτι τέτοιο, ε, η Επίτροπος που είναι αρμόδια για το περιβάλλον θα πρέπει να επιληθεί αυτό το ζήτημα. Ε, είναι προφανώς σημαντικά, αλλά πραγματικά οι υπουργοί περιβάλλοντο οι επίτροποι περιβάλλοντο εκείνοι είναι αρμόδιοι και όχι εγώ. Μετά, αναφερθήκατε και στο ζήτημα, ε, ε, το κοινό σύστημα κρατήσεων. Η Επιτροπή αυτή την περίοδο προετοιμάζει κάποιες προτάσεις και προφανώς εμείς θα συνεχίσουμε αυτή τη διαδικασία αλλά η Ουγγρική Προεδρία θα κληθεί να ολοκληρώσει αυτό το πακέτο. Εμείς δεν θα προλάβουμε να το ολοκληρώσουμε από της δικής μας ε, προεδρίες Ε, μετά σε ό,τι αφορά τη διάσκεψη κορυφή θα είναι 25 και 26 Οκτωβρίου. Με ρωτήσατε πότε ακριβώς θα είναι εκείνη για τον αεροχώρο. Σε ό,τι αφορά το ETS τώρα. Ε, ναι, είναι σημαντικό αυτό το ζήτημα και ο τομέα των οδικών μεταφορών θα πρέπει να παίξει εδώ ένα ρόλο και συμφωνώ. Και επίσης ε, το ΙΤΕΣ έχει επιπτώσει στην τεχνολογία που χρησιμοποιείται στα οχήματά μα και γι' αυτό μπορούμε να επιτύχουμε εδώ και ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα εναντί άλλων υπήρων, άλλων κατασκευαστών. Ε, τώρα στον ε, κύριο Κράμερ ε, νομίζω πως απάντησα εξηγώντα δηλαδή γιατί η σχετική συζήτηση θα γίνει το Δεκέμβριο. Επίση, ό,τι αφορά του ίσου ε, κανόνε παιχνιδιού, αναφέρθηκα και σε αυτό, όπω και στι εκπομπέ διοξιδίου του άνθρακα. Πραγματικά ελπίζω δηλαδή πω εδώ η Λευκή Βίβλο θα μα δώσει τη δυνατότητα να κάνουμε κάποια βήματα παραπάνω, να επιτύχουμε κάποια πρόοδο. Ναι, μετά σε ό,τι αφορά την κατανάλωση αλκοόλ και την οδήγηση, αναφέρθηκα και σε αυτό. Εντάξει, τώρα απόφαση της γερμανικής ε, κυβέρνησης ε, αν θα επιλέξει το Ρήνο, τον Έλβα, δεν ξέρω α, τι ακριβώς θα επιλέξει είναι δικό της θέμα, εθνικής δηλαδή πολιτικής. Ε, αναφέρθηκα και στις εσωτερικές οδούς ναυσιπλοείας. και στις συνδρομικές μεταφορές αναφέρθηκα. Τώρα, σε ό,τι αφορά τον θόρυβο. Θόρυβος από τις ε, μεταφορές. Είπα και προηγουμένως πως δεν είναι σημαντική μόνο η ρήπανση εδώ και κατά συνέπεια η ρήπανση του περιβάλλοντος αλλά και ο θόρυβος που προέρχεται από τις μεταφορές. Θα πρέπει να συζητηθεί και αυτό το ζήτημα. Και Βαντάλη τώρα σε ό,τι αφορά την Ευρωβινιέτα ε, το κάλυψα. Για τα φορτικά είπαμε ότι δεν θα πρέπει να έχουμε 27 ξεχωριστά κουτάκια τα να, πρέπει να συμπληρώνουμε. Είπα και γιατί το Γαλιλαίο ως τεχνολογία είναι πολύ σημαντικό για μας, γιατί με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να επιτύχουμε την θέσπιση ενός ευρωπαϊκού συστήματος. Μέσω δηλαδή των δορυφόρων θα μπορούμε να έχουμε μια κοινή καταχώρηση, μια κοινή πιστοποίηση, χωρίς να έχουμε 27 διαφορετικές ε, καταχωρήσεις εδώ. Ναι, ε, είπατε, αναφερθήκατε και στο ε, υποστηρικτικό πρόγραμμα για τα διαλειτουργικά έργα. Ακόμα δεν έχει αναλυφθεί κάποια πρωτοβουλία σε αυτό το τομέα. Ε, ούτε προβλέπεται κάτι τέτοιο στο δικό μας ε, πρόγραμμα εργασιών, αλλά θα μπορούσα να αναφερθώ στο ζήτημα αυτό στη συνάντηση που θα έχουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πάντως, εις βάθος εξέταση αυτού του ζητήματος δεν θα γίνει κάτι δική μας Προεδρία. Σε ό,τι αφορά τα πρόστιμα, αναφέρθηκα ήδη σε αυτό δεν νομίζω πως μπορεί να αποτελέσει στόχο μας η εναρμόνιση των προστίνων που επιβάλλονται σε όλη την Ευρώπη. Ε, ε νομίζω πως ε, σας απασχόλησα αρκετά και απάντησα σε όλα τα ερωτήματα. Σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Υπουργέ. Ακούσαμε πολύ ενδιαφέρον όσα μας είπατε. Έχουμε όμως πίεση χρόνο Και ε, δεν χαιρέτησα τον Ούγκρο Υπουργό Εθνικής Ανάπτυξης, ο οποίος ήρθε και βγήκε, θα συντηρηθεί μετά από έξι μήνες. Το ξέχασα, παράληψή μου. Ευχαριστώ την κυρία Μπλίκμαν. Αλλά έχουμε εννέα άτομα που έχουν ζητήσει το λόγο ακόμη. Προτείνω λοιπόν για την κυρία Βέκμανς να ακολουθήσουμε τη σειρά εγγραφής και τις ομάδες και να περιοριστείτε Μάξιμου δύο λεπτά, αν γίνεται. Και ένα λεπτό καλό είναι. Και ο κύριος Σούπερ στο τέλος θα κλείσει την πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η συζήτηση. Τεγκράντες Πασκουά. Είστε πρώτος, παρακαλώ σύντομα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, παραδίνομαι. Ε, Θυμάστε ένα φιλμ ε, όπου ε, κατόρθωσε τελικά να ξεφύγει ο ήρωας επειδή είχε δώσει πάρα πολλές εξηγήσει. Ε, εγώ έχω πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη στη Βελγική Προεδρία. Είναι μία από τις χώρες ιδρυτές Ευρωπαϊκής Ένωσης και σίγουρα θα σεβαστείτε τις δεσμεύσεις σας, όμως οι δεσμεύσεις είναι πάρα πολύ φιλόδοξες. Εγώ νομίζω ότι συνειδητοποιείτε ότι πραγματικά εδώ ε, επιζητάτε τους μπελάδες. Γιατί ε, ο συντονιστής μας ε, έθεσε τα κριτριά μας ε, με αρκετά σαφή τρόπο. Εγώ τα προσυπογράφω, απλώς να πω δύο λόγια στο να επιμείνω σε αυτό που είπαμε Ματιέ σε σχέση με την διεθνοποίηση του εξωτερικού κόστους και να προσπαθήσουμε να βρούμε έναν επιμερισμό του κόστους. Γιατί για αυτή την Ευρωβινιέτα αναφερθήκατε στο ότι υπάρχουν διαφορές εδώ και διαφορές στο Συμβούλιο ε, δεν θέλουμε η Ευρωβινιέτα τελικά να είναι ένα παιχνίδι τιμωρίας. Πρέπει να βρούμε μια ισορροπία και έναν τρόπο συμβίωσης μεταξύ των διάφορων τρόπων μεταφορά. Εγώ χάρηκα πάρα πολύ που άκουσα τα λόγια σας. Λευκή Βίβλος. Πιστεύω ότι ε, αν διαβάσετε την έκθεση Cross μπορείτε να δείτε που είναι η συνένεση αυτής της Επιτροπής. Ε, πραγματικά εξαντλητικά είναι τα στοιχεία εκεί και νομίζω ότι συγκεράζονται οι απόψεις των ΜΕ και των ΔΕ. Τώρα για την ε, ασφάλεια της Μεταφορέ, μεταφορές με ενδιαφέρει πάρα πολύ το θέμα. Ήμουν συγγητή ε, για το πακέτο ΕΡΙΚΑ, για ένα κανονισμό και μια οδηγία και για την πολιτική χρηματοδότηση της ΕΜΣΑ θέλει να θέσει τα νέα καθήκοντα της ΕΜΣΑ, η Βελγική Προεδρία επιτάπητος. Το θέμα είναι πώς θα προβούμε στη χρηματοδότηση, να δούμε αν υπάρχουν πόροι ή όχι ή αν ε, θα πρέπει να ε, αλλάξουμε, να τροποποιήσουμε τα καθήκοντα του οργανισμού. Έτσι λοιπόν, ε, κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστούμε για τις μακροσκελείς εξηγήσεις σας, τα λόγια του ε, συντονιστή μα, ε, παρουσιάζουν τις σκέψει μας περί εξεύρεσης ισορροπία. Ε, Σα ευχόμαστε καλή επιτυχία και όταν θα έχουμε περισσότερο χρόνο θα μπορέσουμε να επανέλθουμε στα θέματα αυτά και σας εύχομαι καλή επιτυχία. Ευχαριστούμε. Η κυρία Γιάλα, ευχαριστώ πρόεδρε. Εγώ ήμουν εισηγήτρια για αυτά τα διασυνοριακά πρόστιμα. Έτσι λοιπόν θα ήθελα να σας ευχαριστήσω κύριε Υπουργέ ε, για τις προσπάθειες που καταβάλει η Βελγική Προεδρία εγκαίρως, όμως ε, φοβάμαι μήπως ε, ξανακαταλήξουμε σε αδιέξοδο, γιατί έχουμε κράτη-μέλη που θέλουν να μπλοκάρουν λόγω της νομικής βάσης. Έτσι λοιπόν, εγώ θα ήθελα η Βελική Προεδρία να ακολουθήσει μια πιο ρεαλιστική προσέγγιση, όπου θα αφήσουμε εκτό το θέμα τη ε, νομική βάση και να, να προσπαθήσουμε να σημειώσουμε πρόοδο επί των θεμάτων όπου μπορούμε να συμφωνήσουμε και να ε, χρησιμοποιούμε και ε, τα υφιστάμενα συστήματα χωρίς όμως να τα ονομάζουμε. Και έτσι λοιπόν ε, ξέρω πάρα πολύ καλά ότι εσείς θα μπορέσετε να λύσετε το γόρδιο δεσμό ε, με την νομική υπηρεσία του Συμβουλίου. Δεν βοηθά η νομική υπηρεσία της Προεδρίας να επιλύσουν το ζήτημα, αλλά τελικά βοηθά στην εμπλοκή των ζητημάτων. Έτσι λοιπόν εγώ ελπίζω να μπορέσετε να λύσετε αυτό το γόρδιο δεσμό γιατί αυτό είναι το πρόβλημα που έχουμε τώρα, χρηματοδότηση των τεντή. Ε, το εξάμεινο της Βελγικής Προεδρίας είναι θεμελιώδης σημασίας ε, για να μπορούμε να βρούμε μια διαιτησία στο ότι ε, το δίκτυο των μεταφορών για τις επόμενες δημοσιονομικές προοπτικές να είναι προτεραιότητα. Μετά από έγιναν με το ηφαίστεια και κατέρευσε όλη η Ευρώπη, ανταγωνιστικότητα, δυνατότητα επικοινωνίας κτλ. λόγω ενός προβλήματος και βασιζόμασταν σε ένα μόνο δίκτυο, δηλαδή στο αεροπορικό, το είδαμε αυτό, τώρα χρειαζόμαστε και ένα εναλλακτικό το δεύτερο δίκτυο, προφανώς του σιδηροδρόμους και επομένως θα έπρεπε στις επόμενες δημοσιονομικές προοπτικές να έχουμε ένα ταμείο, να έχουμε μία φόρμουλα μείωση του ελλείμματος, επενδύσεις ε, στα τέντη. δεν ξέρω πώς, αλλά θέλουμε από το 2014 στο 2020 οι μεταφορές σε ευρωπαϊκό επίπεδο να αποτελούν τη λύση και όχι το πρόβλημα Ευρωβινιέτα προσυπογράφω όσο είπε ο κ. Ντεγκράντε, αλλά θα ήθελα να ε, μου πείτε το εξή, εσεί δίνετε πολύ μεγάλη σημασία στι περιφερειακέ χώρε, όμω υπάρχουν και εναλλακτικέ και άλλε δυνατότητε. Εμεί θα ήμασταν διατεθειμένοι να έχουμε ω εναλλακτική πράσινου διαδρόμου, όχι μόνο πράσινου διαδρόμου από περιβαλλοντική σκοπιά, αλλά πράσινου διαδρόμου σε ό,τι αφορά την κινητικότητα και την αποδοτικότητα και τη διατροπικότητα, συντροπικότητα, με συγχωρείτε, έτσι όπου ε, ώστε όλοι οι τρόποι και οι οδικέ μεταφορέ ε, να είναι αποδοτικοί και επίσης να αναφερθώ και στο θέμα της επιμελητίας. Νομίζω ότι υπάρχει κάποια σύγχυση σε ό,τι αφορά τα αποτελέσματα των ομάδων εργασίας που έθεσε σε εφαρμογή κομισιών και θα πρέπει να αναζωογονήσουμε και αυτό το θέμα της οργάνωσης ως λύση για τις μεταφορές. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε για την παρουσίασή σας και για το ότι πριν την Προεδρία προετοιμαστήκατε για το πρόγραμμα αυτό και με μερικά μέλη της Επιτροπής μας. Ήταν πάρα πολύ χρήσιμο αυτό. Ελπίζω το Ευρωκοινοβούλιο και η Προεδρία να ασκήσουμε από κοινού πίεση στην Κομισιόν να βγάλουν αυτή τη λευκή βίβλο πριν το Δεκέμβριο. Δεν ξέρω πώς θα το πετύχουμε, πάντως από κοινού, ήδη από το Σεπτέμβριο, ας ασκήσουμε πίεση στην Κομισιόν. Τρόπος θα υπάρχει γι' αυτό. Ασκήστε πίεση και στον Επίτροπο για την Ευρω... το Ευρωσήμα. Άκουσα με προσοχή αυτά που είπατε. Πολύ ενδιαφέροντα, αλλά ως Κοινοβούλιο το earmarking είναι το σημαντικό. Ο στόχος δεν είναι να γεμίσουν τα κρατικά ταμεία. Ο στόχος είναι να είναι αποτελεσματική η χρήση του συστήματος αυτού. Βιωσιμότητα. Να δούμε ιδιαίτερα τους ιδοδρόμους πόσο αποδοτικά λειτουργούν. «30 δις επιδοτήσεις από την Ένωση και απαλού». Να το δούμε αυτό ξανά για το θόρυβο χρειάζεται η βοήθεια της Ευρώπης. Για τα φορτηγά όμως δεν έχουμε τις ίδιες απαιτήσει. Θα ήθελα στην Προεδρία σας να κάνετε κάτι παραπάνω για τα τρένα. Έχετε πολύ καλή γνώση του θέματος είναι ένα παραμελημένο μέσο μεταφοράς, χρειάζεται προσπάθεια. Ελπίζω στην Προεδρία σας να έχετε μια πιο ευρωπαϊκή φιλοσοφία. Χρειαζόμαστε πολύ περισσότερες ευρωπαϊκές και όχι εθνικές υποδομές. Κύριε Μπούλς, κύριε Πρόεδρε, εγώ δεν θα κάνω ερώτηση θα προτιμούσα να κάνω μια ερώτηση στον Υπουργό Τουρισμού, αλλά χρόνο δεν έχουμε, οπότε δεν θα ρωτήσω. Πρόεδρος, συνεχίζουμε. Πολύ σύντομα κύριε Υπουργέ, είπατε με τη δική σας παρουσίαση πως το Βέλγιο κατά κάποιο τρόπο έχει ε, προκαθοριστεί να αναλάβει την προώθηση του χώρου των μεταφορών ούτως ώστε να καταστεί μια πραγματικά ενιαία αγορά και το διαπιστώνεται στην, ε, με βάση την δική σας ε, χώρα, δηλαδή ένα, μια πυκνοκατοικημένη χώρα η οποία βρίσκεται κεντρικά στην Ευρώπη. Άρα λοιπόν εκεί και οι μεταφορέ ε, transit, διέλευση δηλαδή από άλλε χώρε είναι πολύ σημαντικέ. Άρα λοιπόν ε, ε, χαιρόμαστε με το γεγονό ότι έχετε αναλάβει εδώ να αντιμετωπίσετε τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τέτοιες κεντρικές χώρε και, το, και η Ευρωβινιέτα είναι κάτι που μας ενδιαφέρει και η εναρμόνιση στι δρομικέ μεταφορέ είναι κάτι το οποίο θεωρώ πω είναι πολύ σωστό. Δηλαδή δίκα, στα αναθεώρηση και τη σχετική νομοθεσία από το χώρο των σιδηροδρόμων. Πραγματικά σα καλώ να ακολουθήσετε αυτή την οδό. Ένα τελευταίο σημείο που θα ήθελα να θίξω στον πλαίσιο των παρατηρήσεων μου είναι αυτός ο διάλογος μεταξύ των πολιτικών από το χώρο των μεταφορών αφενός και από τους, των πολιτικών από το χώρο της, του, του γενικά περιφερειακής πολιτικής αφετέρου. Δηλαδή θα πρέπει να ε, εξετάσουμε λίγο ε, το ποιες είναι οι περιοχές ε, στόχοι 1 Δηλαδή, αν δούμε ποιε είναι αυτέ οι περιοχέ στην Ισπανία ε, και, να δούμε, και δούμε από πού ε, λαμβάνουν χρηματοδότηση σε ό,τι αφορά τι υποδομέ, να πούμε ναι, είναι σωστό, αλλά ε, να εξετάσουμε πώ ακριβώ επενδύονται, πού γίνονται αυτέ οι επενδύσει. Και αυτό ισχύει και για άλλε χώρε, όπω για την Ελλάδα ή, για παράδειγμα, για την Ανατολική Γερμανία. Εκεί θα πρέπει πραγματικά να επενδύσουμε και σε κεντρικού διαδρόμου, ώστε να έχουμε μια ενιαία αγορά στην Ευρώπη με εξαιρετική υποδομή μεταφορών. Ευχαριστώ. Uh, domnule președinte, uh, ευχαριστώ Πρόεδρε. Πολύ σύντομα κύριε Υπουργέ, καθώς η μελέτη για το Δούναβι αποτελεί ε, μέρος των εργασιών των τριών Προεδριών, ε, θα ήθελα να μου πείτε ποια είναι η προτεραιότητα που δίνεται σε αυτή τη στρατηγική. Το δεύτερο ερώτημα που θα ήθελα να θέσω είναι πώς θέλετε να αξιοποιήσετε την ε, ενδιάμεση ε, αξιολόγηση ανθρώπων των ε, δημοσιονομικών προοπτικών. Πώς θα αξιολογήσετε λοιπόν αυτήν την ενδιάμεση αναθεώρηση το ώστε τα κράτη-μέλη τα οποία δεν αξιοποίησαν αρκετού διαρθρωτικού πόρου για τι υποδομέ να μπορέσουν να το κάνουν κατά το δεύτερο ήμιση αυτή τη περίοδου. Θα ήθελα και εγώ πολύ σύντομα να πω δύο λόγια, Πρόεδρε. Καταρχήν να συμφωνήσω με την κυρία σε ό,τι αφορά τι ε, υποδομέ μεταφορών και να σα επιστήσω και εγώ την προσοχή, κύριε Υπουργέ, σε αυτό το ζήτημα. Είναι σημαντικό δηλαδή το να προσπαθήσουμε να κάνουμε εδώ κάποια πρόοδο. Ένα δεύτερο ερώτημα, σύντομο θα ήθελα να θέσω Ε, σε ό,τι αφορά την ε, έγκριση των Liner σε, σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Είσαστε θετικά διακείμενος ή δεν αποτελεί αυτό καν ζήτημα για τη δική σας πρόεδρε. Ευχαριστώ. Ε, Κυρία Λίχτεμπεργε. Ευχαριστώ. Τρία ερωτήματα έχω να θέσω κύριε Υπουργέ. Πρώτον, σε ό,τι αφορά την Ευρωβινιέτα. Όταν μας λέτε πως η συνολική επιβάρυνση για τον ε, τομέα των μεταφορών δεν θα πρέπει να αυξηθεί και ε, μιλάμε ταυτόχρονα και για την εσωτερήκευση, των internalization των εξωτερικών ε, δαπανών. Πώς ακριβώς αυτά θα υπάρξουν το ένα δίπλα στο άλλο. Εάν θέλουμε να μείνει ήδη το επίπεδο της επιβάρυνσης της χρηματοδοτικής, πώς ακριβώς θα επιλοποιήσετε την Ευρωβινιέτα. Δεύτερο, σε ό,τι αφορά την το πρωτόκολλο ε, για την, ε, τη συλλοφορία. Ε, θα προσπαθήσετε να το ολοκληρώσετε μετά από έξι χρόνια συζητήσεων. Τρίτο ζήτημα, δικαιώματα των επιβατών. Έτσι όπως αναφερθήκατε στα δικαιώματα των επιβατών, είχα την εντύπωση πως αποτελούν ουσιαστικά κάποια προβληματικά, αν θέλετε, σημεία, κάποιες ενοχλήσεις στην εύρυθμη λειτουργία των μεταφορών. Μα για να δημιουργήσουμε τον ίδιο ε, τους ίδιους κανόνες παιχνιδιού σε όλους τους κλάδους των μεταφορών. Δεν θα πρέπει να έχουμε τις ίδιες ρυθμίσεις. Κατά συνέπεια, δεν θα πρέπει να αποφύγουμε να παραμείνει το status quo στα λεωφορεία. Απαρότε αντιλαμβάνομαι ότι είναι πιο δύσκολα τα πράγματα για τα λεωφορεία, το ίδιο ίσχυε κάποτε και ε, για τους συνδρομού, το ίδιο ίσχυε και για τις ενέργειες μεταφορές. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Πολύ ε, ωραία όλοι αυτή οι φιλόδοξη στόχη, αλλά αν ε, τους ε, εξετάσω και ακούσω τα όσα είπαν οι συνάδελφοι, πραγματικά φοβάμαι ε, ε, ε, φοβάμαι δηλαδή το να αναλαμβάνουμε δράσεις, ένα σωρό δράσεις και να το υποσχόμαστε όλα αυτά στους πολίτες μας χωρίς να επιτυχάνουμε τελικά πάρα πολλά. αναφερθήκατε στα έξυπνα συστήματα μεταφορών. Ναι, είναι πολύ καλό αυτό, αλλά αυτό που με ενδιαφέρει εμένα είναι το τι ακριβώς θα συμβεί στην πράξη και πότε Εάν θέλουμε όμω ε, να έχουμε ε, ε, περισσότερες μεταφορές αλλά με, με λιγότερα οχήματα στον δρόμο τότε πραγματικά θα πρέπει να έχουμε και νέε μετρήσει σε ό,τι αφορά τα οχήματα που βρίσκονται στον δρόμο. Ποια είναι η δική σας θέση. Έχουμε ένα μικρό πρόβλημα. Και ο δείκμας μας περιμένει εδώ και πολύ ώρα με πολύ υπομονή. Και θα ήθελα να ευχαριστήσω και τους συναδέλφους οι οποίοι ήταν σύντομοι αλλά σας έθεσαν πάρα πολλές ερωτήσεις. Πώς τώρα θα απαντήσετε στις 20 ε, ερωτήσεις που σας τέθηκαν. Ε, νομίζω ότι αυτό θα μας καθυστερούσε πάρα πολύ. Όμως, ε, ίσως επειδή βρίσκεστε και κοντά, η γραφική σας εγκύτητα ίσως θα σε επέτρεπε να ξανάλθετε. να παρουσιαστείτε και πάλι ενώπιον μας, γιατί πραγματικά ο πλούτος του προγράμματος ε, και όλες αυτές οι προτάσεις ε, και η ικανότητα να ε, εκφράζεστε για θέματα που μας ενδιαφέρουν όλους προκάλεσε πληθώρα ενδιαφέροντος και μια πολύ πλούσια συζήτηση, όμως πρέπει να ακούσουμε και την Υπουργό Τουρισμού Εμείς θα επιθυμούσαμε να μπορούσατε να ξανάλθετε όταν θα επιστρέψουμε από τις καλοκαιρινές διακοπές, γιατί νομίζω ότι θα ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον να ξαναδούμε όλα αυτά, αφού θα έχουμε κάνει και διακοπές. Νομίζω όμως ότι έχετε τόσο πράγματα να μας πείτε που δεν εξαντλήθηκε το θέμα. Σας ευχαριστώ λοιπόν για το συμπέρασμα που θα ξαγάγατε. Κύριε Πρόεδρε, κοιτάξτε, όπως και να έχει, θα ήθελα να πω δύο λόγια. Γιατί, κύριε Νέμερ, αναφέρθηκε σε αυτές τις ε, τεράστιες ε, γραμμές. Mega project, mega trucks των 60 τόνων, συμπληρώνει ο Πρόεδρος. Είναι τα φορτηγά, τα πολύ μεγάλα φορτηγά. Αν θέλετε να μου τις θέσετε γραπτός, όλες αυτές τις ερωτήσεις να απαντήσω ή να ξανάρθω, ό,τι θέλετε. La volonté du président fait loi. Ah, je vous laisse Μπορείτε όμως να πείτε δύο λόγια συμπερασματικά. Όπως είπα στην εισαγωγή μου, πιστεύω ότι είναι μεγάλες οι προκλήσεις και η βούληση να προχωρήσουμε επίσης είναι μεγάλη. Νομίζω ότι μπορούμε να κάνουμε ένα βήμα προς τα μπρος αν ε, υπάρχουν επαρκές φιλοδοξίες και συνεννόηση μεταξύ Συμβουλίου, Κοινοβουλίου και Κοινοβουλευτικών Ομάδων. Και πιστεύω, και αυτή είναι η βαθιά μου πεποίθηση, ότι αν θέλουμε να μιλήσουμε για μια Ενωμένη Ευρώπη, για μια νέα αγορά, τότε οι μεταφορές διαδραματίζουν ουσιώδη ρόλο και η ενότητα αυτής της Ευρώπης δεν μπορεί να ελοπιθεί παρά μέσω ενός συστήματος μεταφορών που θα λειτουργεί καλά, αλλά και με αρμονικό τρόπο και θα έχουμε ίσω κανόνες για όλους, level playing field, δεν θα ωφελείται κάποιος τομέας περισσότερο από κάποιον άλλο, ούτε θα βρίσκεται σε μειονέκτημα. Νομίζω ότι σε μάκρο οικονομικό, περιβαλλοντικό επίπεδο και σε επίπεδο ασφαλείας θα πρέπει να εντοπίσουμε όλα τα στοιχεία που έχουμε στη διάθεσή μας για να κάνουμε κάποιες επιλογές λογικές, επιλογές που θα τις κάνουμε το επόμενο εξάμεινο, αλλά ελπίζω ότι στα τέλη της Προεδρίας μας τότε θα είναι αρκετά καθορισμένοι με σαφήνεια οι προσανατολισμοί, έτσι ώστε να μπορέσουμε να ακολουθήσουμε μία οδό και να καταλήξουμε σε ικανοποιητικό αποτέλεσμα για αυτή την ενιαία αγορά που αξίζει να υλοποιηθεί και μπορώ να σας πω ότι είναι προς το συμφέρον και της οικονομίας και του περιβάλλοντος αλλά και της ασφάλειας. Χρειαζόμαστε όλη κινητικότητα για να παραμείνει το μέσο των μεταφορών κάτι αποδεκτό στο πνεύμα όλων των Ευρωπαίων. Euh, εγώ ευχαριστώ εξ ονόματος όλων σας για αυτές ε, τις ε, παθιασμένες παρεμβάσεις και νομίζω ότι ε, εμείς είμαστε συμμαχοί σας και πραγματικά παρακολουθούμε πολύ κοντά τις προτάσεις μας και πραγματικά μας ανοίξατε την όρεξη. Έτσι λοιπόν να ξανάρθετε το φθινόπωρο. mesdames messieurs, je votre attention euh, Παρακαλώ, μπορώ να έχω την προσοχή σας κυρίες και κύριοι για το δεύτερο τμήμα της συνεδρίασής μας σήμερα το απόγευμα. je, remercie, euh, Madame Ευχαριστώ την κυρία Βέγμαντς που είναι υπουργός pourrait euh, tenir les conversations euh, dedans sans voix ou dehors à voix παρακαλώ αν θέλετε να συζητήσετε εκτός της αίθουσας. Λοιπόν, ευχαριστώ την ε, κυρία Δέκμαν της Υπουργού Τουρισμού για την επίσκεψή της στην Επιτροπή μας και φυσικά εκτιμούμε και την πρώτη φορά που υποδεχόμαστε εδώ Υπουργό Τουρισμού ως αρμόδια επιτροπή στο πλαίσιο της ε, συνθήκης της Έτσι λοιπόν, είμαστε αρμόδιοι στο επιχειρησιακό σκέλος του ζητήματος. Λοιπόν, σας ευχαριστώ για την υπομονή σας και θα σας δώσω απευθείας το λόγο. Ja, sehr geehrter Präsident, werte Kolleginnen und Kollegen. Ε, να σας πω ότι καταρχήν δεν ευθύνομαι εγώ που δεν μπόρεσε ο συνάδελφος να απαντήσει στα ερωτήματά σας ε, και χρειάστηκε να φύγει. Ε, σίγουρα θα ξαναέρθει για να συζητήσετε. σε, κάθε περίπτωση με χαρά μου βρίσκομαι σήμερα εδώ για να συζητήσω μαζί σας τις προτεραιότητες της Βελγικής Προεδρίας και να τις παρουσιάσω καταρχήν. Ε, με πεπισμένη πως η ανταλλαγή απόψεων θα είναι πολύ ενδιαφέρουσα γιατί η δική σας Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού όπως διαφάνηκε μόλις ε, τώρα έχει μια ιδιαίτερη δυναμική και ε, θεωρείται πολύ σημαντική. Ε, να σας πω επίσης ευθύς εξ αρχής ότι μετά από αυτή τη συζήτηση θα βρίσκομαι και εγώ και οι συνεργάτες μου στη διάθεσή σας για να απαντήσω σε περαιτέρω ερωτήματα και να αναφερθώ σε ζητήματα που σας ενδιαφέρουν. Ε, και τώρα ε, θα ήθελα Πρωτού αναφερθώ στο πρόγραμμα της Βελτικής Προεδρίας για τον τουρισμό να κάνω κάποιες παρατηρήσεις τις οποίες ε, ίσως δεν ακούτε για πρώτη φορά. Για παράδειγμα αναφέρθηκαν από τον δικό μας Πρωθυπουργό του Βελτιού και να πω πως ο τουρισμός για τη δική μας χώρα έχει μια ιδιαίτερη σημασία και παρότι δεν έχουν ακόμα ολοκληρωθεί, ολοκληρωθεί οι συζητήσει για τη σύσταση τη Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση του Βελγίου, ε, αυτό ε, δεν θα έχει επιπτώσει ε, στην δική μα ενασχόληση με το ζήτημα και δεν θα επηρεάσει αρνητικά το πρόγραμμα τη δική μα Προεδρία τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Είχαμε τον κατάλληλο χρόνο στη διάθεσή μα να προετοιμάσουμε αυτό το πρόγραμμα και θα το υλοποιήσουμε στο ακέραιο. Να θυμίσω όμω ότι αποτελεί ένα περιφερειακό ζήτημα, ε, ζήτημα ε, περιοχών. Ε, δηλαδή έχουμε καταρχήν τη γερμανόφωνη περιοχή εκείνη της πρωτεύουσα και της Βαλωνίας που είναι αρμόδια. Κατά συνέπεια το πρόγραμμα το οποίο θα σας παρουσιάσω σήμερα έχει συνταχθεί με συνέπεια σε συνεργασία με όλες τις περιοχές και κατά συνέπεια ε, δεν ε, υπάρχουν επιπλοκές ε, με τη μεταβατική αυτή περίοδο μέχρι τη σύσταση δηλαδή της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης του Βελγίου. Άρα λοιπόν έχουμε κάνει ό,τι μπορούμε ούτως ώστε να ανταποκριθούμε στις προσδοκίες σας απέναντι στην Βελγική Προεδρία. Οι προτεραιότητε τις οποίες έχουμε θέσει έχουν συζητηθεί και με τις άλλες δύο προεδρίες, την Ισπανία δηλαδή και την Ουγγαρία και έτσι για πρώτη φορά μετά από τη συνθήκη της Λισαβόνας ε, θα έχουμε τη δυνατότητα να εργαστούμε με αυτόν τον τρόπο και θα ήθελα με αυτή την ευκαιρία να ε, συγχαρώ ε, τον προκάτοχό μου, τον Χουάν Μισκίτα, τον Υπουργό Τουρισμό, για τη δουλειά που έκανα κατά τη διάρκεια των τελευταίων έξι μηνών, πραγματικά θέτοντας εδώ κάποια θεμέλια για την κοινωτική πολιτική. Τώρα, δεν χρειάζεται να σας υπενθυμίσω ότι εδώ ε, κινούμαστε κατά εφαρμογή του άρθρου 195 της Συνθήκης της Λισαβόνας και ε, συζητάμε λοιπόν για ε, την μελλοντική ευρωπαϊκή πολιτική τουρισμού και την ε, λήψη ιδιαίτερων συγκεκριμένων μέτρων από την, στο πλαίσιο δηλαδή αυτής της πολιτικής συμπληρωματικά προς τα εθνικά μέτρα. ο κλάδος του τουρισμού με τις 1,8 εκατομμύρια μικρομεσαίες επιχειρήσεις ε, αντιστοιχεί στο 5% του ευρωπαϊκού ΑΕΠ και το έμεσο δηλαδή το άμεσα συνδεδεμένο προϊόν καθάριση του εθνικό προϊόν αντιστοιχεί στο 10% και από πλευρά απασχόλησης το αναλογεί το 12%. Η, η ανάπτυξη εδώ στο πλοίο τη απασχόληση είναι, ε, ο ρυθμό ανάπτυξη είναι πολύ υψηλότερο από ότι ε, σε άλλου ε, κλάδου τη οικονομία και γι' αυτό υπενθυμίζω εδώ κάτι το οποίο βέβαια γνωρίζετε, ότι είναι πολύ σημαντικό ο τουρισμό, ο κλάδο του τουρισμού για την ευρωπαϊκή διάσταση, αλλά και όταν συζητάμε το πώ μπορεί να συμβάλλει ο κλάδο αυτό στην υλοποίηση των στόχων τη στρατηγική 2020. Δεν θα πρέπει να ξεχνούμε όμως ταυτόχρονα ότι ο τουρισμός όπως και άλλοι κλάδοι με τους οποίους ασχολείται πεθαμένο στο Κοινοβούλιο ε, πλήττεται από κρίσεις και συγκεκριμένα την ε, κρίση την οποία διερχόμαστε ακόμα. Όμως θα πρέπει εδώ να υπενθυμίσουμε ότι ο τουρισμός ε, βιώνει μια ταχύτερη ανάκαμψη από ό,τι αυτό συμβαίνει σε άλλους κλάδους της οικονομίας. Άρα λοιπόν και αυτό αποτελεί ένα σημαντικό επιχείρημα ως προς το γιατί είναι τόσο σημαντικός ο κλάδος του τουρισμού στο πλαίσιο της Αδηγική 2020. Στο πλαίσιο αυτό ο διατομιακός χαρακτήρας ε, του τουρισμού αφορά και πάρα πολλά επίπεδα πολιτικής, ε, για παράδειγμα και σε ε, εθνικό και σε περιφερειακό επίπεδο και επιτρέψτε μου να αναφερθώ ε, σε διάφορα παραδείγματα πολιτική ανταγωνισμού, πολιτική εσωτερικής αγοράς, πολιτική απασχόλησης, πολιτική προστασία του περιβάλλοντος, ανάπτυξη της υπαίθρου και περιφερειακή ανάπτυξη. Σε όλους λοιπόν αυτούς τους τομείς πολιτικής έχει να παίξει ρόλο ο τουρισμός αλλά και σε σχέση για παράδειγμα με την προστασία των καταναλωτών και ένας ο άλλος τομέα στου οποίου δεν θα αναφέρω τώρα. οι προκλήσει τι οποίε αντιμετωπίζει ο τουρισμό ε, σήμερα και σε επιστημονικό και σε οικολογικό και σε κοινωνικό επίπεδο είναι πολλέ και αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι ε, με τα απαραίτητα προσαρμοσμένα εργαλεία να μπορέσουμε να κάνουμε ε, ό,τι πρέπει. Και ε, μέσα σε αυτό το πλαίσιο συναντήθηκαν και οι αρμόδιοι Υπουργοί Τουρισμού και οι Υφυπουργοί τους ε, στις 15 ε, Απριλίου του 2010 στη Μαδρίτη και σε συνέχεια αυτής της διάσκεψης εγκρίθηκε ομόφωνα η δήλωση της Μαδρίτης για, μια, για ένα βιώσιμο μοντέλο τουρισμού. Και στο πλαίσιο αυτής της δήλωσης ε, τα κράτη-μέλη εξέφρασαν την βούλησή τους για την ανάπτυξη μιας τέτοιας, ε, ε, ενός τέτοιου βιώσιμου και κοινωνικού μοντέλου τουρισμού και αναφέρθηκε και ανάγκη ενός ηθικού, ενός υπεύθυνου τουρισμού, ο οποίος δηλαδή θα είναι κοινωνικός, θα είναι φιλοπεριβαλλοντικός, θα, είναι, θα σέβεται την πολιτιστική κληρονομιά και ούτω ε, Τα κράτη-μέλη ε, πρότειναν νέα εργαλεία και μια νέα πιο στοχευμένη προσέγγιση σε ό,τι αφορά τη γνώση και την γενοτομία στον τουρισμό μέσω της αξιοποίησης νέων τεχνολογιών και επίσης ε, πρότειναν την δικτύωση και την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών. Ταυτόχρονα η δήλωσή τους καλεί και την Ευρώπη να δώσει μια άλλη ορατότητα, ένα πιο έντονο προφίλ αν θέλετε σε αυτόν τον ε, τομέα. Δηλαδή να μην δημιουργεί εμπόδια σε ό,τι αφορά τις ε, ροές ε, τουρισμού αλλά να λάβει ένα ρόλο υποστηρικτικό. Η Βελγική Προεδρία χαίρεται επιχαίρεται την ανακοίνωση της Επιτροπής ε, για την Ευρώπη ως ε, το πιο σημαντικό ε, τουριστικό προορισμό στην Ευρώπη όπως παρουσιάστηκε στις 30 Ιουνίου και διαπιστώνουμε και εμείς ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έλαβε υπόψη της τις συστάσεις της δήλωσης της Μαδρίτης και ότι προέβη και σε ακρόαση με τον ε, ιδιωτικό τομέα και τις ε, ομοσπονδίες και τα δίκτυα από τον ε, κλάδο αυτό για να εμπλουτίσει περισσότερο αυτή την ανακοίνωση. Η ανακοίνωση λοιπόν αυτή έχει την πρόθεση να δημιουργήσει ένα σχέδιο, ένα πλαίσιο δράσης το οποίο θα επιτρέψει την, τον ανταγωνιστικό χαρακτήρα αλλά και τη δυνατότητα μιας βιώσιμης ανάπτυξης του τουρισμού και λαμβάνοντα υπόψη και την ε, συνθήκη της Λισαβόνας ε, προτείνονται ε, διάφορες πρωτοβουλίες οι οποίες εστιάζουν σε 4-5 βασικούς τομείς προτεραιότητα, τους οποίους θα έχετε ήδη διαβάσει θεωρώ καταρχήν την τόνωση της ανταγωνιστικότητας του τομέα του τουρισμού η προώθηση και η ανάπτυξη ενός υπεύθυνου και ενός βιώσιμου τουρισμού ως τρίτο, στόχο η ε, περαιτέρω ανάπτυξη, επέκταση του προφίλ και της ορατότητας της Ευρώπης ως ε, μια ποιοτική, ένας ποιοτικός ε, και βιώσιμος προορισμός τουρισμού και η συμπερίληψη του τουρισμού στην πολιτική και στα χρηματοδοτικά εργαλεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να εκπονήσει και να υλοποιήσει αυτό το σχέδιο δράση σε στενή συνεργασία και με τα κράτη-μέλη αλλά με και του βασικού ενδιαφερόμενου από τον κλάδο του τουρισμού. Άρα λοιπόν, ε, σε τι θα βασιστεί η Βελγική Προεδρία και τι έχουμε προετοιμάσει και έχουμε παρουσιάσει και στους δύο εταίρους μας ε, στο πλαίσιο των ε, Προεδριών. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό, είναι πολύ σαφές ε, για τη Βελγική Προεδρία ότι ακολουθούμε ένα συγκεκριμένο στόχο. Δημιουργία σαφών βάσεων για την μελλοντική ε, πολιτική τουρισμού της Ευρώπης. Δηλαδή, ποιοι θα είναι εκείνοι οι τομείς στους οποίους μπορούμε να κινηθούμε συμπληρωματικά ε, προς τις πολιτικές των κρατομελών, πού μπορούμε να δώσουμε αυτές τις δυνατότητες και αυτό θα γίνει μόλις θα λάβει η χώρα και το νέο επίσημο Συμβούλιο Τουρισμού και υπό Βελγική Προεδρία θα έχουμε ε, για πρώτη φορά ένα τέτοιο συμβούλιο και θέλουμε να δώσουμε έμφαση σε ένα τέτοιο συμβούλιο σε αυτή τη σύνθεση όπου θα, δώσουμε, θα υπογραμμίσουμε και την ανακοίνωση της Επιτροπής αλλά και την ανάγκη για τον καθορισμό των βασικών πυλώνων της μελλοντική ε, ευρωπαϊκής πολιτικής του τουρισμού. Και βασισμένη σε αυτό θα ασχοληθεί και το Ευρωπαϊκό Φόρουμ Τουρισμού, το EFT, το οποίο θα ε, λάβει χώρα τον Νοέμβριο ε, με αυτό το ζήτημα και θα εξεταστεί το πώς μπορεί το φόρουμ αυτό να ε, συμβάλλει σε συντονισμό και με τους ενδιαφερόμενους φορείς σε ανάπτυξη αυτής της πολιτικής. Αλλά εμείς θα προσπαθήσουμε να συνεργαστούμε και με τους Ούγγρους συναδέλφους που μας διαδεχτούν στην Προεδρία, ώστε να υπάρξει αυτή η βιωσιμότητα. Όμω, ε, ποια είναι πιο συγκεκριμένα τα ζητήματα τα οποία θέλει να προωθήσει η Βελγική Προεδρία. Θα σα ε, δώσω μια σύντομη επισκόπηση ω προ τα θεματικά πεδία τα οποία θέλουμε να προωθήσουμε και τα οποία ε, ελπίζουμε να οδηγήσουν σε συγκεκριμένα συμπεράσματα του Συμβουλίου. Καταρχήν, θα ασχοληθούμε με το ζήτημα το πώς ε, θα ε, προωθήσουμε όπως είπα και προηγουμένως έναν υπεύθυνο, βιώσιμο και ποιοτικό τουρισμό, πώς λοιπόν θα υλοποιηθεί αυτό ούτως ώστε ε, να αποτελέσει το διακριτικό χαρακτηριστικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να αποκτήσει και η Ευρωπαϊκή Ένωση περισσότερη ορατότητα στο τουρισμό. Μπορεί λοιπόν να αποκτήσει μεγαλύτερο, πιο έντονο προφίλ εάν τονίσουμε ακριβώς τον ποιοτικό και βιώσιμο χαρακτήρα και αν τονίσουμε και τα κριτήρια βιωσιμότητας ε, και υπευθυνότητας ε, που διακρίνουν τον τουρισμό μας. Ε, αυτό ούτως ή άλλως θα λάβει χώρα, αλλά θέλουμε να του δώσουμε ακόμα μεγαλύτερη έμφαση, να δείξουμε ε, πώς μπορούμε να κάνουμε κάτι τέτοιο συνεργασία και με κάποια προγράμματα τα οποία έχουμε κινήσει σε αυτόν τον τομέα μετά, ένα άλλο θεματικό πεδίο θα είναι ο πολιτισμός και ο Εντάξει, θα μπορούσε κανεί να βρει ότι υπάρχει ξεχωριστό φόρουμ, αν θέλετε, και ε, ξεχωριστέ ομάδε που συζητάνε τα ζητήματα πολιτισμού και κουλτούρα στην Ευρώπη, αλλά ε, δεν συζητούν τα αφορά αυτά ζητήματα τουρισμού τόσο ιδιαίτερα. Άρα λοιπόν, όταν ε, ε, μιλάμε εδώ για, την, ε, για τον ε, πολιτισμό, μιλάμε για ένα πάρα πολύ πλούσιο τομέα, ειδικότερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτή η πολιτιστική ποικιλομορφία είναι κάτι το οποίο μπορούμε να προσφέρουμε στο επίπεδο του τουρισμού. Υπάρχουν διάφορες πρωτοβουλίες που έχουν αναλυφθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τον πολιτισμό και θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν καλύτερα από τον τουρισμό. Και αυτό βέβαια θα μα ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο όταν θέλουμε να έχουμε ένα τουρισμό ο οποίος δεν είναι τουρισμός μόνο για τις παράκτη περιοχές ή μόνο για τις ορεινές περιοχές ή μόνο για τις αστικές περιοχές αλλά για ένα τουρισμό των περιφερειών, των περιοχών γενικά ε, γιατί μπορούν να υπάρξουν εδώ κάποιες νέες λύσεις, κάποιες νέες προσεγγίσεις που μπορούν να λειτουργήσουν ως ε, παραδείγματα. Για παράδειγμα, να συζητήσουμε το πώς μπορούμε την βιομηχανική μας κληρονομιά να την προωθήσουμε περισσότερο στο πλαίσιο του τουρισμού. Ή για παράδειγμα το ζήτημα των ε, πολιτιστικών ε, πρωτευουσών. Ε, όλα αυτά λοιπόν τα επιμέρους ζητήματα θέλουμε να, τα, να τους δώσουμε περισσότερη έμφαση. Μετά ένα άλλο ζήτημα στο οποίο θα μπορούσαμε να αναφερθούμε, αλλά μόνο λίγη εισαγωγή, χωρί δηλαδή να είμαστε σε θέση να εμβαθύνουμε είναι η δυνατότητα ανταλλαγή συμβέντηση των πρακτικών και ο τρόπο που θα μπορούσαμε να προβούμε σε μια ανταλλαγή πρακτικών. Η Επιτροπή προτείνει στο δικό τη έγγραφο ότι να υπάρχει μια ψηφιακή πλατφόρμα η οποία θα μπορούσε να εγγυηθεί αυτή η ανταλλαγή βελτιστών πρακτικών. αποτελεί λοιπόν κάτι τέτοιο μια καλή λύση, ένα καλό παράδειγμα, αλλά ίσω θα πρέπει καταρχήν να εξετάσουμε. Υπάρχουν άλλε δυνατότητε. Δυνατότητε ενδεχομένω τι οποίε έχουμε εφαρμόσει σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Μήπω θα μπορούσαμε να κάνουμε ένα βήμα παραπέρα. να πούμε δηλαδή ότι χρειαζόμαστε περισσότερες γνώσεις για το τουρισμό για να μπορούμε να ε, δρούμε καλύτερα και για να έχουμε περισσότερες γνώσεις χρειαζόμαστε και ανταλλαγή αυτών των βέλτιστων πρακτικών. Ποιε μεθόδου θα ακολουθήσουμε για να προβούμε σε αυτή την ανταλλαγή ε, βέλτιστων πρακτικών και απόψεων χωρί να δημιουργήσουμε περιττή ε, υποδομή και περιττό φόρτο εργασία που θα μα ευκολύνουν όμω να έχουμε καλύτερη υλοποίηση τη πολιτική τουρισμού μα. Επίσης θα προτείνουμε στα κράτη-μέλη να αναγνωρίσουν για μία ακόμα φορά το σημαντικό ρόλο που παίζει ο κλάδος του τουρισμού ε, στην οικονομία. Ναι, γνωρίζω πως ε, δεν είναι κάτι για το οποίο υπάρχουν αντιρρήσεις αλλά δεν χρειάζεται μόνος ε, να αναφέρεται σε μια βασική συνθήκη κάτι τέτοιο θα μπορούσαμε να το αναφέρουμε και εμείς πιο συγκεκριμένα ρητά και επίσης θα πρέπει να αναφέρουμε ε, την ε, προώθηση της Ευρώπης ως προορισμού για τον τουρισμό λέγοντας για παράδειγμα ότι θα μπορούσαμε να λαντσάρουμε αν θέλετε τους αυτούς μας και μέσω του διαδικτύου. Η ε, καινοτομία τώρα παίζει ένα σημαντικό ρόλο και στον χώρο του τουρισμού, όχι μόνο σε άλλους ε, τομείς. Ειδικότερα στο επίπεδο των μικρών, μικρομεσαίων επιχειρήσεων παίζει μεγάλο ρόλο η καινοτομία στον ε, τουρισμό. όπως και ανάπτυξη και αξιοποίηση νέων τεχνολογιών και εδώ πάλι οι σχετικέ ε, τεχνολογίες ICT ε, είναι σημαντικέ. Ε, επίση, ο τουρισμό έχει να παίξει ένα πολύ σημαντικό ρόλο σε ό,τι αφορά την οικοδόμηση μια κοινή οικονομική και κοινωνική ευρωπαϊκή ταυτότητα. Ε, αναφέρθηκα και μόλι τώρα και στον πολιτιστικό τουρισμό και επίση ε, στο ευρωπαϊκό του για την καταπολέμηση της φτώχειας ε, και, του κοινωνικού αποκλεισμού καλό θα ήταν να αναφερθεί και η πτυχή του κοινωνικού τουρισμού. Ο κοινωνικός τουρισμός, ο οποίος σε πολλές ε, χώρες έχει ήδη μια μεγάλη παράδοση, θέτει το ερώτημα του τι μπορεί να παράσχει ως κίνητρο η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτό λοιπόν αποτελεί κάτι το σημαντικό για την Βελγική Προεδρία. Ελπίζω να μένει περίπου το 1 τέταρτο που μου δόθηκε από τον πρόεδρο, ώστε να έχουμε τώρα ακόμα 3 τέταρτα στη διάθεσή μα κανονικά για την ε, συζήτηση. Οπότε αναμένω με ενδιαφέρον ε, την συζήτηση που θα γίνει και τα σχόλιά σα. Ευχαριστώ. Euh, τα είπατε πάρα πολύ γρήγορα, σεβαστήκατε και τις προθεσμίες. Να δώσουμε τα λόγο τώρα στο συντονιστή μας, ο κύριος Ματία Γκρός καταρχήν. Ευχαριστώ. Πρόεδρε. Ε, δύο καινοτομίες έχουμε σήμερα. Πρώτον, και εμείς για πρώτη φορά ασχολούμαστε στο πλούσιο της Λισαβόνας με τον τουρισμό και δεύτερον έχουμε μια γερμανόφωνη υπουργό για πρώτη φορά που μας μιλάει εδώ στην, ε, στις ε, Βρυξέλλες και μάλιστα μας ε, προτείνει και πολύ καλές και ενδιαφέρουσες ιδέες. Ο τουρισμός λοιπόν είναι ένας σημαντικός κλάδος και βρισκόμαστε εδώ σε μια επιτροπή η οποία ασχολείται, αν πάρουμε δηλαδή συνολικά ε, μεταφορές ε, και τουρισμό ε, με 20 εκατομμύρια απασχολούμενους. Και πραγματικά πρέπει να εξετάσουμε σε κάποιο σημείο το πώς μπορούμε να οικοδομήσουμε μια γέφυρα μεταξύ κινητικότητας και τουρισμού. Δηλαδή να μην ασχολούμαστε μόνο με την ε, βιώσιμη ανάπτυξη της ε, κινητικότητας και των μεταφορών γενικά, αλλά και ταυτόχρονα να ενδιαφερόμαστε και τη βιώσιμη ανάπτυξη του τουρισμού. Η ανάπτυξη του τουρισμού βέβαια έχει και τις ε, δικές της παγίδες, γιατί κάποιες φορές ο καθένας θέλει να εξελιχθεί τόσο αυτόνομα, ούτως ώστε τελικά να μην υπάρχει επαφή μεταξύ των διαφόρων κρατών μέλων. Εσείς λοιπόν πώς το βλέπετε, πώς, πώς θέλετε να Ξεφύγεται από αυτό το μοντέλο του να έχουμε δηλαδή αυτόν τον αυτόνομο, τον κατακαιρματισμένο τουρισμό. Πώς θα μπορούσε αυτό να επιτευχθεί και με ε, χρήση ευρωπαϊκών ε, ε, πόρων. Είναι πολύ ενδιαφέρον σε όλες αυτές οι δηλώσεις βέβαια κάθε φορά που ακούμε, αλλά τίθεται κατευθείαν και το ερώτημα του πώς θα χρηματοδοτηθούν όλα αυτά. Γιατί τελικά δεν, είναι, δεν επαρκούν μόνο οι καλές ιδέες, είναι καλές ιδέες, αλλά χρειαζόμαστε και ιδέες ως προς το πώς θα χρηματοδοτηθούν όλα αυτά. Ο κύριος ε, Μπράιν ε, Σίμψον, ε, ο πρόεδρος μας, θα είχε πραγματικά χάρη πάρα πολύ αν ήταν εδώ και σας άκουγε να λέτε πως υπάρχει σχέση, για παράδειγμα, μεταξύ βιομηχανίας και τουρισμού, δηλαδή της της κληρονομιάς που έχουμε αυτό το τομέα και πράγματι γενικά ο πολιτισμός εδώ μπορεί να μας ε, βοηθήσει. Αναφερθήκατε και στον κοινωνικό τουρισμό, κύριε Υπουργέ. Ε, και εδώ νομίζω πως ε, ένα σημαντικός υποκλάδος θα είναι ο τουρισμός για τα άτομα με περιορισμένη κινητικότητα. Μιλάμε για 120 εκατομμύρια ανθρώπου ε, στην Ευρώπη, μιλάμε δηλαδή για πολύ ε, μεγάλη μερίδα των πολιτών. Και επίσης ε, θα ήθελα να μα πείτε, έχετε αναλογιστεί καθόλου το ενδεχόμενο τη συζήτηση κοινών προτύπων, τα οποία θα ισχύουν πανευρω... πανευρωπαϊκά. Εντάξει, δεν φαντάζομαι να καταφέρετε μέχρι τα τέλη του, του έτους αυτού να επιτύχετε ένα σύστημα, για παράδειγμα, όπου τα δύο αστέρια για ένα ξενοδοχείο θα σημαίνουν το ίδιο σε όλα τα κράτη-μέλη, αλλά τουλάχιστον θα μπορούσε ενδεχομένως να υπάρξει μια συζήτηση ε, τουλάχιστον ε, σε ό,τι αφορά αυτή τη δυνατότητα ε, εναρμόνισης και σε κάθε περίπτωση να σας πω ότι έχετε εδώ μια επιτροπή η οποία πραγματικά σας, θα σας συμπαρασταθεί ούτως ώστε όχι μόνο να προτείνετε αυτές τις ιδέες αλλά και να τις υλοποιήσετε. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε Ματιά. Κύριος Αλκαντράουι. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Καταρχήν να σας ευχαριστήσω κυρία Υπουργέ για την εισαγωγική σας παρουσίαση και να σας πω ότι η δική μου ομάδα θα σας στηρίξει τα μάλλα. Ο τουρισμός είναι ένας πολύ σημαντικός τομέας, αλλά επίσης πρέπει να γνωρίζουμε ότι και μέχρι σήμερα η δική μας, το δικό μας περιθώριο λιγμών εδώ στην Επιτροπή ήταν πάρα πολύ περιορισμένο σε σχέση με όσα κάναμε στον τομέα των μεταφορών. Τώρα πρέπει να καταβάλουμε μεγαλύτερε προσπάθειε για τον τουρισμό. Πρόκειται για ένα πολύ μεγάλο τομέα που δημιουργεί πολλέ θέσει εργασία. Αμφισβήτητα η Ευρώπη στο σύνολό τη είναι ο πρώτος προορισμός παγκοσμίω, όμως δεν έχουμε μια συντονισμένη στρατηγική για να χρησιμοποιήσουμε όσο δυνατόν καλύτερα αυτό το δυναμικό. Έτσι λοιπόν θα πρέπει να καταβάλουμε προσπάθειες προς αυτήν την κατεύθυνση. Τώρα που έχει τεθεί σε ισχύ η συνθήκη τη Λισαβόνα ε, και που συμπεριλαμβάνεται ο τουρισμός στη συνθήκη αυτή ως ε, προτεραιότητα, πρέπει μέσω της ε, πολιτικής για τις μεταφορές να δούμε ποιες επιπτώσεις θα υπάρχουν και στον τουρισμό. Μοιραία θα υπάρχουν όταν μιλάμε ε, για τη βελτίωση των υποδομών, για τα δικαιώματα των επιβατών, όλα αυτά έχουν επιπτώσει και στον τουρισμό. Αλλά πέρα από αυτά πρέπει να προβούμε σε ακόμη μεγαλύτερο συντονισμό. Θα πρέπει να συλλέξουμε καλύτερα τα στατιστικά στοιχεία, κάτι που δεν είναι καθόλου απλό. Και παραδείγματο χάρη ένα ξενοδοχείο ενό αστέρα δεν είναι το ίδιο με ένα ξενοδοχείο ενό αστέρα σε μια άλλα κράτο Και επίση πρέπει να έχουμε και ολοκληρωμένε πληροφορίε. Πρέπει να υπάρχει μια πύλη για όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά θα πρέπει να τα σκεφτούμε όλα αυτά περαιτέρω. Η πρόταση που έχουμε εδώ, να υπάρχει ένα νέο σύστημα έκδοση εισιτηρίων, ε, είναι κάτι πολύ ενδιαφέρον, αλλά θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε αυτό το σύστημα και σε άλλου τομεί. Εμεί ε, θα το κάνουμε αυτό στον τομέα των μεταφορών. Εσεί, ω ε, Υπουργό Τουρισμού, θα μπορούσατε να δείτε και ποιε είναι, ποια είναι τα πλεονεκτήματα που απορρέουν για τον τουρισμό από κάτι τέτοιο. Επίσης θα πρέπει να συντονίσουμε και τη χρήση των υφιστάμενων υποδομών έτσι ώστε να γεμίζουν και τα ξενοδοχεία ή μάλιστα να γεμίζουν ε, στις ε, περιόδους ε, χαμηλής ζήτησης. Γιατί εγώ νομίζω ότι η προσθέμενη αξία της Ευρώπης είναι στο ότι εφευρίσκει και νέες ιδέες για τον τουρισμό. Επινοεί νέες ιδέες, έτσι περίπτωση χάρη, σκεφτήκαμε ε, τις πολιτιστικές διαδρομές. Υπάρχουν και άλλες ε, ιδέες που μπορούμε να σκεφτούμε για να υπάρχει τουρισμός σε όλη την Ευρώπη και φυσικά μπορούμε να βελτιώσουμε και την ποιότητα. Για να ολοκληρώσω. Πιστεύω ότι μπορούμε να κάνουμε και μια συζήτηση για την εναρμόνιση επί κάποιων θεμάτων. Πώς προτείνατε ελάχιστα κριτήρια για να βοηθήσουμε και τα άτομα με ειδικέ ανάγκες. Επίσης, ελάχιστα κριτήρια για την αξιολόγηση των ξενοδοχείων, αλλά θα πρέπει να έχουμε ένα χρονοδιάγραμμα. Τουλάχιστον να σχηματίσουμε μια ιδέα για το πόσο χρόνο χρειάζεται για να φτάσουμε σε μια καλύτερη εναρμόνιση. Σα έχουμε και φυσικά κάθε επιτυχία στο εξάμεινο τη Προεδρία σα. Και ελπίζω ότι θα έχουμε ενδιαφέροντα αποτελέσματα στα τέλη του έτους. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Μάισνερ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Χαίρομαι πολύ στη σήμερα εδώ, κύριε Υπουργέ. Ε, και εγώ πραγματικά χαίρομαι πως έχουμε αυτή τη νέα αρμοδιότητα για την ανάπτυξη του τουρισμού σε ευρωπαϊκό επίπεδο και μπορώ να φανταστώ και εγώ πολλά πράγματα γιατί ήδη έχει εξελιχθεί ο τουρισμός. Έχετε ε, πολύ δίκιο όταν λέτε πως ε, υπάρχει ένα μεγάλο κομμάτι των απασχολούμενων που ε, απασχολούνται στον τουρισμό και μόνο και μόνο για αυτό το λόγο ο τουρισμός είναι πολύ σημαντικός και γενικά οι άνθρωποι έχουν περισσότερο ελεύθερο χρόνο στη διάθεσή τους από ό,τι στο παρελθόν και αυτό θα συνεχίσει να ισχύει. Θέλουν να αξιοποιήσουν αυτόν τον ελεύθερο χρόνο που έχουν στη διάθεσή τους. Δεν έχουν πάρα πολλά χρήματα και υπάρχει και μια τάση που λέει ότι δεν θέλω να πάω εκεί που υπάρχει πολλοί κόσμος. Άρα λοιπόν τίθεται και το πρόβλημα του που ακριβώ θα πάνε όλοι αυτοί. Ε, εντάξει, υπάρχουν πολλοί οι οποίοι θα ήθελαν να πάνε στη Μαγιόρκα και να πιούν ε, κάποια ποτά, ενώ άλλοι ε, θέλουν να πάνε στα βουνά και να κάνουν κάποια extreme sports. Αλλά υπάρχει και μια μερίδα η οποία προτιμάει κάτι άλλο. Αν σκεφτώ τον εαυτό μου ή και γνωστού μου, ε, και πραγματικά για αυτούς θα πρέπει να βρούμε ε, κάποιους, ε, κάποιες εναλλακτικές τις οποίες θα μπορούσαμε να αξιοποιήσουμε καλύτερα. Άρα λοιπόν ε, σε ένα ευρωπαϊκό φόρουμ όπως αυτό που θα γίνει μπορούν να συγκεντρωθούν πολλές ε, τέτοιες ιδέες που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε πιο απτά αποτελέσματα. Και εδώ θα θέσω λοιπόν το ερώτημα πότε ακριβώς είναι η ημερομηνία για αυτό το φόρουμ και πότε θα υπάρξει το, πότε θα λάβει χώρα το, ε, Συμβούλιο ε, Τουρισμού μα είπατε το Νοέμβριο. Νοέμβριο είναι 30 ημέρε. Μπορείτε να μα πείτε πιο συγκεκριμένα μια ημερομηνία. Θα μα βοηθούσε πολύ. Κάτι τέτοιο θα μπορούσε να αποτελέσει το πρότυπο για έναν ποιοτικό και όχι θορυβόδη αλλά ήσυχο ε, τουρισμό όπως τον φαντάζονται νομίζω πολλοί άνθρωποι πλέον. Ε, προτού επισέλθω τώρα ε, σε άλλα ζητήματα. Να πω και ένα-δυο λόγια ακόμα. Ε, κοινωνικός τουρισμός, αναφερθήκατε σε αυτόν γιατί υπάρχουν και ε, άτομα τα οποία έχουν περιορισμένη κινητικότητα, έχουν κάποια αναπηρία ή δεν έχουν πολλούς πόρους στη διάθεσή τους, αλλά παρόλα αυτά θέλουν να ε, πάνε κάπου για διακοπές ε, και υπάρχουν βέβαια περίοδοι τουριστικές στις οποίες είναι τα πάντα γεμάτα και έχουν γίνει κρατήσει για τα πάντα ενώ υπάρχουν κάποιες άλλες περίοδοι που είναι νεκρές και δεν υπάρχει τίποτα. Θα πρέπει να δούμε πώς θα υπάρξει μια καλύτερη κατανομή ε, υπάρχουν πολλές ιδέες τις οποίες, τις οποίες θα μπορούσαμε να έχουμε κοινή διαχείριση, για παράδειγμα ε, βιομηχανική κληρονομιά. Εγώ είμαι, ε, ε κοντά στον Τάστρο, όπως ε, πραγματικά υπάρχουν κάποια παλιά ορυχεία εκεί που εντάξει δεν είναι κάτι ιδιαίτερα σημαντικό αλλά πραγματικά για τη δική μου περιοχή αποτελεί μια τουριστική ατραξιόν αξιοθέατο άρα λοιπόν τέτοιου είδους στοιχεία θα μπορούσαμε να τα προωθήσουμε και υπάρχει ε, η τάση πολύ έντονα στη δική μου χώρα ε, για ενδιαφέρον ε, για το μεσαίωνα. Έτσι. Κάτι τέτοιο δεν μπορεί να υπάρξει κάπου αλλού, δεν μπορεί να υπάρξει στην Αμερική εκ των πραγμάτων. Υπάρχει δηλαδή εδώ ένα τομέα ο οποίο είναι μοναδικό και υπάρχουν πάρα πολλοί νέοι οι οποίοι ενδιαφέρονται. Ε, υπάρχουν και πολλέ ταινίε κινηματογράφου, για παράδειγμα ο Χάρι Πότερ, εντάξει είναι κάτι το μεσαιωνικό, αλλά υπάρχει μια τάση για ενδιαφέρον για ε, τέτοια ζητήματα και γενικά ιστορικές αναδρομές ε, αποτελούν μια νέα τάση. Για παράδειγμα, το να ακολουθεί κανεί ε, τα αχνάρια ενός συγκεκριμένου καλλιτέχνη, ενός συγγραφέα, ενός ζωγράφου ε, στην Ευρώπη. Και είναι, συμβαίνει δηλαδή κάποιοι άπονες οι να μην επισκέπτονται μόνο συγκεκριμένα αξιοθέατα, αλλά να ακολουθούν τη διαδρομή της ζωής ενός συγκεκριμένου καλλιτέχνη. Άρα λοιπόν βλέπετε ότι έχω πολλές ιδέες και θα ήθελα να συμμετάσχω. Υπάρχουν ε, λοιπόν ε, και κάποιες, ε, κάποια αξιοθέατα, κάποιες περιοχές οι οποίες εστιάζουν περισσότερο στη φύση, δηλαδή ο κόσμος θέλει να μεταβεί στη φύση και να εξετάσει και να δει, να, να απλά τα αξιοθέατα της φύσης. Βλέπετε λοιπόν ότι εδώ επεκτείνομαι πολύ γιατί Πρόκειται για έναν ε, τομέα ο οποίος με ενθουσιάζει. Μετά, ε, παλιές ε, πολιτιστικές πρακτικές και πολιτιστικές οι παλαιότερες τέχνες αποτελούν στοιχεία τα οποία ενδιαφέρουν πολύ. Και τέλος να περάσω και στις παράκτες περιοχές γιατί και εγώ από την κάτω σαξονία προέρχομαι και υπάρχει από το 2009 ένα εθνικό πάρκο το οποίο θα μπορούσε για παράδειγμα να αποτελέσει ε, ε, για το πώς μπορούμε να συνδυάσουμε ένα παράδειγμα για το πώς μπορούμε να συνδυάσουμε από τη μία την προστασία συγκεκριμένων ε, φυσικών περιοχών με έναν μετριασμένο, με έναν φιλικό προς τα περιβάλλοντα αυτά του τουρισμού. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κυρία Μάισνερ. Και εγώ ευχαριστώ την ε, κυρία Υπουργό για την παρουσίασή της. Ε, έχουμε, είχαμε συναντηθεί και στο παρελθόν και στη δέσμευση στη Μαδρίτη και ε, να πούμε ότι ο τουρισμός μπορεί να είναι δημιουργικός και να διασφαλίσει 20 εκατομμύρια θέσεις εργασίας αλλά μπορεί να είναι και καταστροφικός. Να το πούμε και αυτό. Μπορεί να είναι καταστροφικός ο τουρισμός ε, και έχουμε δει ότι μεγάλα ε, μεγάλες ε, ζώνες ε, παράκτιες σε χώρες της Μεσογείου έχουν καταστραφεί από τον τουρισμό, από την τουριστική αξιοποίηση και ίσως θα πρέπει να γίνει μια ανάλυση ως προς το πώς οδηγήθηκαν αυτές οι περιοχές σε αυτό το τομέα, δηλαδή τουριστικές περιοχές οι οποίες πλέον δεν, δεν προσελκύουν τουρισμό γιατί έχουν καταστραφεί. Και ίσως θα μπορούσαμε να συμπεριλάβουμε το σημείο υπαριθμών 16 ε, στο δικό μας ε, τουριστικό σύστημα. Δηλαδή, όχι να λέμε το πόσο, πόσο μακριά βρίσκεται ένας ε, προορισμός μέσω μιας πτήσης, αλλά μπορούμε να, δούμε, να, να συμπεριλαμβάνουμε τι, για παράδειγμα, και πόσες ώρες χρειαζόμαστε με το τρένο ή με το πλοίο. Θα πρέπει δηλαδή να κινηθούμε υποστηρικτικά προς συγκεκριμένους συγκεκριμένα είδη τουρισμού, εάν θέλουμε τελικά να δώσουμε την ευκαιρία και στι μελλοντικέ γενιέ να μπορούν να πηγαίνουν ε, για τουρισμό. Δηλαδή, ο τουρισμό πρέπει να είναι βιώσιμο όχι μόνο από τι πηγέ που αναφέρθηκαν, αλλά γενικά εκ των πραγμάτων πρέπει να είναι βιώσιμο. Επίση, να πούμε ε, πω ε, ο ρυθμό ανάπτυξη του τουρισμού βρίσκεται στο 20% ετησίω εδώ και πολλά χρόνια, τι τελευταίε δεκαετίε. και πραγματικά έχουμε ε, ε, δει, ε, έχουμε για παράδειγμα 70.000 ποδηλατόδρομους μέσα από τη φύση, τους οποίους μπορούν πάρα πολύ να εμπιστευτούν. Υπάρχουν κάποιες διαδρομές, όπως εκείνη που, που έχει ως τελικό προορισμό το Σαντιάγο του Κοποστέλα. Και να σας πω πως ο ποδηλατικός τουρισμός ε, έχει αναπτυχθεί τόσο πολύ γιατί. Γιατί έλεγε ε, αρχικά κανεί ότι πριν από 15-20 χρόνια το που ξεκίνησε ότι ε, καλό είναι να κινείται κανεί μόνο κατά μήκο ακτών ή λιμνών ή οτιδήποτε άλλο. Αλλά μετά άρχισαν να έχουν καινούριε ιδέε και να λένε θα ήθελα να δω συγκεκριμένα ιστορικά αξιοθέατα. Ήθελα, θα ήθελα να δω για παράδειγμα να ακολουθήσω το σιδηρό παραπέτασμα, δηλαδή κάποια αξιοθέατα κατά μήκο αυτή τη αυτής της γραμμής και μάλιστα κατευθύνεται γύρω ε, κατά μήκο περιοχών οι οποίες ήταν, ε, ε, δεν ήταν καθόλου δημοφιλείς όχι μόνο για την δυτική πλευρά αλλά και για την ανατολική πλευρά. Και ε, διαδρομέ, για παράδειγμα, μέσα από τα Περινέα Είναι και αυτή μια ακόμα διαδρομή, την οποία ακολουθούν μόνο μάλλον έμπειροι υποδηλάτε. και εκεί ακριβώς όπου δεν μπορούμε να προσελκύσουμε τους ε, διάφορους ε, τουρίστες ε, μπορούμε να το κάνουμε βάζοντας κάποια τέτοια στοιχεία πολιτισμικά, ιστορικά και ούτω Μιλάμε λοιπόν εδώ για έναν τομέα ο οποίος μπορεί να προστατεύσει το περιβάλλον γιατί ακριβώς μπορούμε να έχουμε τέτοια εναλλακτικούς τρόπους τουρισμού αλλά και προωθεί και τι περιοχέ, Γιατί για το, για το Βερολίνο δεν χρειαζόμαστε κάποιο τουριστικό πρόγραμμα ούτε για τη Βαρκελόνη, ούτε για τη Ρώμη, ούτε για τη Φλωρεντία. Ε, εμεί θέλουμε να υποστηρίξουμε και να προωθήσουμε τι ε, περιοχέ εκείνε οι οποίε δεν συγκεντρώνουν τουρισμό. Δηλαδή οι περιοχέ οι οποίε ήδη βιώνουν ε, ένα αποκορύφωμα στην τουριστική ανάπτυξη δεν χρειάζονται περαιτέρω υποστήριξη. Επίση, εμεί θέλουμε να προωθήσουμε το να είναι δυνατό το ποδήλατο να μεταφέρεται σε όλα τα τρένα. Ε, εντάξει, η ΙΤΣΕΡΕ της Γερμανίας ακόμα ε, προβάλλει κάποια αντίσταση, αλλά υπάρχει για παράδειγμα το ΤΖΒ και άλλοι που έχουν αποδεχτεί αυτή τη δυνατότητα. Να ε, προτείνετε λοιπόν και αυτό, ότι υπάρχουν και άλλες δυνατότητες μετακίνησης ε, και στο πλαίσιο του τουρισμού, όχι μόνο με το αυτοκίνητο. Τέλος, σε ό,τι αφορά το ε, ε κινητικότητα, το mobility, εδώ πραγματικά συμφωνώ με ε, την ευρωπαϊκή προσέγγιση. Ε, δεν θα επιτρέπεται, δεν πρέπει να επιτρέπεται η οικοδόμηση ούτε ενό ξενοδοχείου το οποίο δεν θα προβλέπει την απαραίτητη υποδομή για άτομα με αναπηρία. Σε ό,τι αφορά παλαιότερα ξενοδοχεία, ναι, θα πρέπει να δούμε το πώ μπορούμε να κάνουμε κάποιε τροποποιήσει, αλλά κανένα καινούργιο ξενοδοχείο χωρί αντίστοιχη υποδομή. Αυτά από την πλευρά μου. Σα ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Κράμερ. Κυρία Υπουργέ, έχετε το λόγο για μια πρώτη σειρά απαντήσεων και μετά θα συνεχίσουν πάλι οι συνάδελφοι. Ευχαριστώ Πρόεδρε και ευχαριστώ όσους ε, πήραν ε, το λόγο και ε, για τα ερωτήματα που έθεσαν. Εκείνο που καθίσταται σαφές είναι ακριβώς αυτός ο διατομιακός χαρακτήρας του τουρισμού. Ο κύριος Γκρός το ανάφερε, ο κύριος Κεντουρή και η κυρία Μάρισνα και ο κύριος Κράμερα αναφέρθηκαν σε αυτό είτε πρόκειται δηλαδή για την κοινότητα γενικά, το mobility, το ποιο ρόλο μπορεί δηλαδή να παίξει εδώ ο τουρισμός, είτε πρόκειται για την ε, πολιτική περιβάλλοντος και εκεί έχει να παίξει σημαντικό ρόλο ο τουρισμός και να πούμε πως εάν η Ευρωπαϊκή Ένωση δραστηριοποιηθεί σε αυτό το τομέα του τουρισμού δεν θα δραστηριοποιηθεί στο πλαίσιο των όσων ήδη λαμβάνουν χώρα Η Ένωση δηλαδή θα δραστηριοποιηθεί μόνο εφόσον κάτι είναι φιλοπεριβαλλοντικό και μόνο εφόσον κάτι ε, επιφέρει μια προστιθέμενη αξία στα όσα ήδη λαμβάνουν χώρα σε επίπεδο κρατών μελών. Θα πρέπει αυτό δηλαδή να το θέσουμε στο επίκεντρο. Θα δραστηριοποιηθεί, θα αναλάβει δράση η Ευρωπαϊκή Ένωση μόνο εφόσον κάτι ε, δίνει επιπρόσθετη χρησιμότητα στις προσπάθειες που ήδη έχουν αναλυθεί σε εθνικό επίπεδο. Και γι' αυτό και στα συμπεράσματα θα δείτε ότι θα αναφέρεται κάτι μόνο εφόσον υπόσχεται να είναι ε, φίλο περιβαλλοντικό σε ό,τι αφορά τον τουρισμό, να, είναι, να προωθεί τον κοινωνικό τουρισμό και να έχει προσθέμενη αξία. Και από εκεί και μετά περνάω σε αυτό που ανέφεραν ε, διάφοροι ομιλητέ. Δηλαδή, θα μπορούσαμε να έχουμε μια ρύθμιση ούτως ώστε όλες οι υποδομές στον τουρισμό, ε, ξενοδοχεία και ούτω καθεξής να έχουν την κατάλληλη υποδομή για άτομα με αναπηρία. Η απάντηση είναι όχι, δεν μπορούμε να προβλέψουμε ένα τέτοιο κανονισμό, αλλά τίθεται το ερώτημα του πώς μπορούμε να έχουμε μία μεθοδολογία για την ανταλλαγή πρακτικών, λαμβάνοντα υπόψη την αρχή τη επικουρικότητα. Και να πούμε δηλαδή ότι αν θέλει η Ευρώπη να αναδειχθεί όσο ε, ο πλέον ανταγωνιστικό ε, ε, και ποιοτικό ε, τουρισμού. Να πούμε ότι αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνο εφόσον ε, πληρούνται μεταξύ άλλων και αυτά τα πρότυπα. Δηλαδή της προσβασιμότητας για κάθε άνθρωπο, δηλαδή και για άτομα με αναπηρία. Εάν θέλουμε να έχουμε λοιπόν μια Ευρώπη η οποία ακολουθεί αυτόν τον στόχο σε ό,τι αφορά το τουρισμό και θέλει να επιτύχει αυτόν τον στόχο, τότε θα πρέπει να ακολουθήσουμε αυτή την κατεύθυνση. δεν θα μπορούσαμε να έχουμε μια διάταξη την οποία θα επιβάλλουμε στα κράτη-μέλη σε αυτή τη φάση. Πρόκειται δηλαδή για μια προσέγγιση που θα λάβει η χώρα σε θελούσια βάση. Τι μπορούμε δηλαδή εμείς να προτείνουμε ως κίνητρα, πώς μπορούμε να, να δώσουμε μια όθηση στην Ευρώπη προς αυτή την κατεύθυνση. Αυτή είναι η συζήτηση που γίνεται σε αυτό το επίπεδο, σε αυτή τη φάση και να πω πως ε, στην πλειοψηφία των κρατών μελών δεν αποτελεί Κάνει ζήτημα το ότι εάν εδώ αναλάβει δράση η Ευρωπαϊκή Ένωση προφανώς θα το κάνει εφόσον πρόκειται για μια δράση η οποία είναι βιώσιμη, είναι φιλική προς τον περιβάλλον και λαμβάνει υπόψη και τέτοιες παραμέτρους. Επίσης, με ρωτήσατε πότε θα ξεκινήσει το φόρουμ 18. 18 και 19 του μήνα θα λάβει χώρα στη Μάλτα. Δεν ξέρω αν έχουμε συναδέλφους από τη Μάλτα. Δεν βλέπω κάποιον. Είναι λίγο περίεργο, αλλά δεν είναι, αν το σκεφτείτε, γιατί συμφωνήσαμε με την ε, ε, Μάλτα ότι το δικό μας Ευρωπαϊκό Φόρουμ για τον Τουρισμό θα λάβει χώρα εκεί 18 και 19 Οκτωβρίου. Το Συμβούλιο βέβαια 11 και 12 Οκτωβρίου στο Λουξεμβούργο. Τι θα μεταβούμε στο Λουξεμβούργο. Εύκολο αυτό. Αυτές είναι και οι προθεσμίες που έχουμε μπροστά μας και βέβαια θα προσπαθήσουμε να βασιστούμε στα όσα θα ε, υποθούν στο φόρουμ ούτως ώστε να έχουμε καλύτερα συμπεράσματα στο επίπεδο του Συμβουλίου για να δούμε δηλαδή ποια μέτρα υλοποίησης ε, μπορούμε να προωθήσουμε. Και χαίρομαι που μου βεβαιώσατε σήμερα εδώ ότι ο τουρισμός και η μελλοντική πολιτική τουρισμού θα πρέπει να εστιάσει ε, εκεί όπου υπάρχει και ανάγκη για ανάληψη δράσης. Θα πρέπει δηλαδή να έχουμε συγκεκριμένα κριτήρια κατά νου σε ό,τι αφορά δηλαδή τη φιλικότητα προς το περιβάλλον, σε ό,τι αφορά την ε, προσβασιμότητα για άτομα με αναπηρία, αλλά και σε ό,τι αφορά τη γεωγραφική κατανομή, να προωθούμε δηλαδή ε, περιοχές οι οποίες δεν βρίσκονται για παράδειγμα σε ορεινή περιοχή, σε παράκτη περιοχή, να προωθήσουμε λοιπόν αυτές τις περιοχές και να αξιοποιήσουμε τα όσα εφόδια στο πούμε, έχουμε στη διάθεσή μας αυτές τις ε, περιοχές είτε είναι ιστορικά αξιοθέατα είτε είναι διαδρομές ε, ε, για ποδήλατα ή για περιπάτους και το Συμβούλιο της Ευρώπης έχει ενεργοποιηθεί σε σχέση με αυτό το ζήτημα έχει δραστηριοποιηθεί δηλαδή στον τομέα αυτών των ε, διαδρομών και, ε, και ε, σε ό,τι αφορά την σημασία των περιφερειών για τη χάραξη αυτής της ευρωπαϊκής πολιτικής τουρισμού. Σας λέω ότι ναι και εγώ ως Υπουργός από συγκεκριμένη περιφέρεια γνωρίζω πόσο σημαντικό είναι να υπάρχει μια τέτοια συνεργασία και σε διαπεριφερειακό και σε διασυνοριακό επίπεδο και τα ευρωπαϊκά τα ταμεία θα χρειαστεί να παίξουν σημαντικό ρόλο όπως το έχουν κάνει και μέχρι σήμερα σε ό,τι αφορά δηλαδή την ε, δημιουργία κοινών ε, project, κοινών ε, έργων ευρωπαϊκής υποδομής και βέβαια τονίζω μία ακόμα φορά τον διατομεακό, τον γενικό χαρακτήρα του τουρισμού. αυτό είναι πολύ σημαντικό. Έτσι λοιπόν είναι και η δική μας εντολή, αυτό που καλούμαστε εμείς να πράξουμε για το χαρακτήρα που άπτεται και της περιφερειακής ε, πολιτικής και της περιβαλλοντικής πολιτικής της Ευρωπαϊκή Ένωσης και να πούμε λοιπόν ότι κατά συνέπεια θα πρέπει η μελλοντική ευρωπαϊκή πολιτική ε, τουρισμού να είναι συνεκτική και να ευθυγραμμίζεται με τις υπόλοιπες ε, πολιτικές ε, σε επίπεδο της Ευρωπαϊκής Αυτό θα προσπαθήσουμε να κάνω. Ελπίζω να απάντησα σε όλα τα ερωτήματα της ε, παρατηρήσης που έγιναν. Η εναρμόνιση των προτύπων γενικά. Εντάξει, εγώ αναφέρθηκα μόνο στα πρότυπα σε ό,τι αφορά την υποδομή για άτομα με αναπηρία, αλλά σε ό,τι αφορά τα πρότυπα γενικά, για παράδειγμα την κατηγορία των, τις διαφορετικές κατηγορίες των ξενοδοχείων, να πω πως και σε αυτό το τομέα δεν μπορεί να υπάρξει κοινή ρύθμιση σε ό,τι αφορά δηλαδή κοινά πρότυπα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η συνθήκη της Λισαβόνας δεν μας δίνει την ε, κατάλληλη αρμοδιότητα, αλλά ε, μπορεί να γίνει μια συζήτηση σε σχέση με αυτό. Δηλαδή να πούμε, το ξαναλέω, ότι εάν θέλουμε να έχουμε ένα ποιοτικό τουρισμό στην Ευρώπη, τότε θα πρέπει να έχουμε και πρότυπα επί των οποίων θα συμφωνήσουμε. Αλλά εδώ θα πρέπει να γίνει μια ανταλλαγή απόψεων, να επιτευχθεί μια συμφωνία και τελικά να υπάρξει μια ε, ε αν θέλετε, ε, συμφωνία, θελωτική συμφωνία. Δεν μπορεί δηλαδή να έχει τεσμευτικό χαρακτήρα μια τέτοια μια τέτοια προσπάθεια, αλλά θα πρέπει να προσπαθήσουμε να κάνουμε κάποιο βήμα εδώ, γιατί ε, εδώ στον τουρισμό έχει να παίξει και πολύ σημαντικό ρόλο ο ιδιωτικός τομέας. Ο ιδιωτικός ε, τομέας ε, ε, εφαρμόζει δικά του κριτήρια και υπάρχουν μάλιστα κράτη-μέλη τα οποία δεν θέτουν συγκεκριμένα πρότυπα, συγκεκριμένες προϋποθέσεις και το κάνουν οι ίδιοι κλάδοι τουριστικοί σε αυτές τις χώρες. Άρα λοιπόν ε, πρόκειται για μια συζήτηση η οποία θα πρέπει να γίνει και ε, με βάση αυτήν την προοπτική. Δηλαδή και σε συνάντηση με τον ιδιωτικό τομέα και εδώ θα έρθει να συμβάλλει το Ευρωπαϊκό Φόρουμ Τουρισμού γιατί οι ενδιαφερόμενοι φορείς, ο ιδιωτικό κλάδο έχει τη δυνατότητα να συζητήσει μαζί μα και ό,τι μπορεί να συμβάλλει στη μεγαλύτερη ορατότητα του τουριστικού κλάδου θα το δεχτούμε. Δεν θα υπάρξει δηλαδή επιφυλακτικότητα από την δική μας ε, πλευρά είναι σαφές ότι και εδώ ή ε, ο κλάδος, ο ιδιωτικό κλάδος θέλει να συμμετάσχει ενεργά στη σχετική συζήτηση. Σας ευχαριστώ. Euh, Ας περάσουμε τώρα στο δεύτερο γύρο. Έχουμε έξι ομιλητές, δύο λεφτά maximum. γιατί ο υπουργό έχει υποχρεώσει. Θα χρειαστεί να φύγει. Κύριε Χάνερα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, χαίρομαι που έχετε θέσει τόσο φιλόδοξους ε, στόχους ε, για τη δική σα ε, Προεδρία και για το γεγονό ότι δίνετε έμφαση στον πολιτιστικό τουρισμό και στον ιστορικό ε, τουρισμό, γιατί αυτά τα είδη τουρισμού είναι πολύ σημαντικά και για δική μου χώρα, την Αυστρία. Θα ήθελα να επιτύχουμε αυτόν τον ε, στόχο, δηλαδή μια κοινή ευρωπαϊκή πολιτική στην οποία μπορούν να συμμετάσχουν και να συμφωνήσουν όλα τα κράτη-μέλη. Ε, πέραν αυτού, τα όσα ε, προγράμματα τα οποία θα συζητήσουμε, και εδώ έχετε την υποστήριξή μα, θα χρειαστεί να συζητήσουμε και τα τη χρηματοδότησή του. Θα ήθελα να σα ρωτήσω, εσεί είστε υπέρ του να υπάρξει μια χρηματοδότηση ενό συγκεκριμένου, ενό ξεχωριστού κεφαλαίου ε, για τον τουρισμό στον προπολογισμό τη Ένωση. Στη διαφορετική περίπτωση θα μιλάμε μόνο για πιλωτικά ε, project. Δεν θα έπρεπε να δημιουργηθεί ένα ξεχωριστό κεφάλαιο στον προπολογισμό. Επίσης, Ε, σε ό,τι αφορά την ε, ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εκεί διαβάσαμε έστω και λίγο έμεσα ότι υπάρχει και το ζήτημα ε, των ροών των τουριστών κατά τη διάρκεια των διακοπών, των περιόδων διακοπών και διαπιστώνουμε ότι υπάρχουν πάντα κάποιες ε, περίοδοι οι οποίες και για τον κλάδο αλλά και για τους ίδιους τουρίστες είναι ε, ιδιαίτερα μεγάλη ζήτηση και κάποιες άλλες νεκρές ε, περίοδοι οπότε θα πρέπει εδώ να κάνουμε μια προσπάθεια να υπάρξει μια κατανομή. Αντιλαμβάνομαι ότι δεν είναι κάτι το οποίο μπορούμε να λύσουμε μέσα σε μια μέρα, αλλά να δούμε, να αρχίσουμε να εξετάζουμε σιγά σιγά το τι μπορούμε να κάνουμε και να δούμε αν υπάρξει και η βούληση από την πλευρά των κρατών μελών να κάνουν κάτι τέτοιο. σε κάθε περίπτωση αναμένω με ενδιαφέρον την έργα που θα αναλάβουμε. Merci Madame Rader. Madame euh, qui nous a généreusement laissé son intervention tout à l'heure. Πριν είπατε δεν θέλετε να μιλήσετε, τώρα έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Χαίρομαι που μου δίνει η ευκαιρία με την Υπουργό να κάνουμε μια συζήτηση καλά διορθωμένη για τον τουρισμό από την συνθήκη της Αβώνας και μετά Έχουμε αρμοδιότητες για τον τουρισμό. Από την Πορτογαλική Προεδρία του 2007 και μετά μέχρι σήμερα το Συμβούλιο δεν ασχολήθηκε με θέματα του τουρισμού. Αυτό είναι πολύ εύγλωτο για τη στάση των κυβερνήσεων και πόσο ενδιαφέρονται για τον τουρισμό. Μας παρουσιάσετε ένα σωρό ενδιαφέρουσες ιδέες. Γραπτά μας δεν έχω δει τίποτα. Εγώ περίμενα ένα πρόγραμμα στην ιστοσελίδα σας, ας πούμε, της Προεδρίας σας. Συγκεκριμένες προτάσεις υπάρχουν. Θα τις διαβάσω όταν θα είναι διατυπωμένες γραπτά, για να δούμε και αν είναι δυνατόν εφαρμοσμούν, βέβαια. Αναφερθήκατε στο ετήσιο φόρουμ που φέτος θα το οργανώσετε στη Μάλτα Λίγο περίεργο αυτό είπατε. και εγώ το βρίσκω πάρα πολύ περίεργο. Στο παρελθόν αυτό το ετήσιο φόρουμ γινότανε πάντα στη χώρα της Προεδρίας. Και ήταν μια μεγάλη ευκαιρία για μας, γιατί πρόκειται για μια περιφερειακού χαρακτήρα πολιτική και δεν άκουσα για ποιο λόγο θα γίνει στη Μάλτα φέτος. Θα ήθελα να μου πείτε αν ξέρετε γιατί. Ασχοληθήκατε με, θίξατε πάρα πολλά θέματα τα οποία είναι όλα ενδιαφέροντα, διαφυσβήτητα. Ωστόσο, θα πρέπει να δούμε λίγο το θέμα του τουριστικού μάρκετινγκ. και την ανάγκη συνεργασία συνοριακών περιοχών. Εγώ ε, κατοικώ στο Λιμπούργο στο από την βελγική πλευρά και μας ενδιαφέρει η συνεργασία με την άλλη πλευρά. Ολλανδία, Βαλονία, Γερμανία. Έτσι, με αυτή την καλή συνεργασία, την διασυνοριακή, όλοι ωφελούμαστε. Δεν αρκούν επενδύσεις δηλαδή μόνο σε μία συγκεκριμένη περιοχή. Χρειάζεται συνεργασία μεταξύ περιοχών που βρίσκονται γύρω-γύρω από έναν κοινό σύνορο. Θα μπορούσε να γίνει μια μελέτη, μια ανάλυση. Τι εμπόδια ακόμα υπάρχουν που πρέπει να τα υπερπηδήσουμε αν θέλουμε μια ανταγωνιστική, τουριστική δραστηριότητα. Είναι είδος βίζας, είναι φόρου, τι υπάρχουν που θα πρέπει να καταργηθούν. Μιλάω για άχρηστα εμπόδια. Ευχαριστώ. Πρόεδρος. Και τώρα το λόγο στην κυρία Γιάλα Σάντερς. Ευχαριστώ, Πρόεδρο. Συγγνώμη, έπρεπε να βγω γιατί με πήραν τηλέφωνο από την Ισπανία. Καταρχήν σα ευχαριστώ πολύ κύριε Υπουργέ και φυσικά να σας καλωσορίσω στην Επιτροπή αυτή. Εγώ εδώ έχω μία μικρή παράθεση που λέτε μία συνένεση για να οικοδομήσουμε μια πολιτική για τον τουρισμό έτσι ώστε η Ένωση να αποκτήσει τα δημοσιονομικά μέσα προς αυτή την κατεύθυνση. Πάρα πολύ μου άρεσαν τα όσα δηλώσατε γιατί το να μιλούμε για ένα δημοσιονομικό μέσο για τον τουρισμό ε, ουσιαστικά υποστηρίζει αυτό που λέμε εμείς ότι πρέπει ο τουρισμός να έχει τα δικά του μέσα και φυσικά ε, στο παρελθόν είχαμε και κάποιους συνομιλητές οι οποίοι το αρνούνταν αυτό. Έτσι λοιπόν χαίρομαι πάρα πολύ που το δηλώνετε σε αυτό. Σας υποστηρίζω 100%. Είναι πολύ γενναία αυτή η δήλωση. Τώρα, πέρα από την ανακοίνωση που παρουσιάσατε εσείς ως βάση για το πρόγραμμα της Βελγικής Προεδρίας, εγώ νομίζω ότι η Προεδρία ουσιαστικά έχει δύο ε, προτεραιότητες. Έχουμε τους ε, ηλικιωμένους οι οποίοι ε, έχουν πάρα πολύ ελεύθερο χρόνο και έχουν και δυνατότητα να επενδύσουν. Ε, υφίσταται αυτή η δυνατότητα, ίσως να είναι μέτρια, αλλά υφίσταται και είδαμε ε, ότι στην Ισπανία ε, η πρόθεση του τουρισμού και της κινητικότητας έχει μάλλον το ότι ταξιδιεύουν τα άτομα αυτά έχει πάρα πολύ μεγάλες επιπτώσεις στην υγεία τους. Έτσι λοιπόν, αυτή η δυνατότητα που έχει ο τουρισμός ε, κατά τη διάρκεια ε, των ε, χαμηλών περιόδων, όπως τις λέμε, να γεμίζουν τα ξενοδοχεία μέσω εκδήλωσης διάφορων ενδιαφερόντων για την γαστρονομία, για την πολιτιστική κληρονομιά κτλ. Αυτό είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον και έχουμε και τους αναδιόμενους ε, τουρίστες. Έχουμε ε, το θέμα των θεωρήσεων ε, ή το πρόβλημα του μάρκετινγκ, πώς θα προωθήσουμε την Ευρώπη ως ένα παγκόσμιο προορισμό. Εγώ σας υποστηρίζω σε όλα αυτά στις σκέψεις που εκφράσετε σχετικά με τα ζητήματα αυτά. Και επίση συμφωνώ με το ότι πρέπει να έχουμε κάποια πρότυπα σε ό,τι αφορά την ποιότητα αλλά και την εξομοίωση και θα πρέπει να μιλάμε και για ε, κάποια πρότυπα σε ό,τι αφορά τους επαγγελματίες του κλάδου. Στην Ισπανία, παρά το ότι έχουμε πάρα πολύ καλές σχολές τουρισμού και πολύ καλούς επαγγελματίες, ε, υπάρχει αυτή η ιδέα ότι οποιοδήποτε μπορεί να κάνει αυτή τη δουλειά. Όχι, δεν είναι αλήθεια κάτι τέτοιο. Εγώ νομίζω ότι θα ήταν πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε ένα είδος ε, τουριστικού εράσμους, δηλαδή να υπάρχουν κάποιε επαγγελματικέ ε, ανταλλαγέ. Είδαμε στην γαστρονομία λόγου χάρη υπήρξε πάρα πολύ μεγάλη αύξηση στην ανταλλαγή μεταξύ Γάλλων και Ισπανών. Δεν ξέρω τώρα ποια άκουσα καλύτερη, αλλά μπορούμε να έχουμε αυτού του είδου τι ανταλλαγέ, ε, έτσι ώστε να ενισχυθεί ο τουρισμό μέσα από αυτή τη διαδικασία. Σα ευχαριστώ. Ευχαριστούμε την κυρία Γιάλα. Ο κύριος Δεγκράντε Πασκουάλ. Να ευχαριστώ πρόεδρε. Καλώ ήρθατε κυρία Υπουργέ στην Επιτροπή αυτή. Χαίρομαι που σας ε, ξανασυναντώ αφού είχα τη δυνατότητα να παρευρεθώ μαζί στη Μαδρίτη σε κάποιε ημερίδε πολύ ενδιαφέρουσε. Θα είμαι σύντομο για να μην επαναλάβω πολλά από τα θέματα που αναφέρθηκαν από τους συναδέλφους. Ε, εγώ Είχα σκεφτεί ότι σε κάποια στιγμή κρίσης ε, μπορεί πραγματικά ο τουρισμός να είναι το εφαλτήριο για να οδηγηθούμε στην ε, ευημερία. Συμφωνώ με το μοντέλο του τρίου των Προεδριών, ε, το οποίο προωθεί την κοινωνική αλληλεγγύη και επίσης συμφωνώ και με τη θεώρηση της Βελγικής Προεδρίας. Ε, είναι φιλόδοξο το πρόγραμμά σας, ε, είναι, ε, είναι πολύ μεγάλο το πολιτικό βεληνικές, θέλετε να συνσφέρετε στην προώθηση της ποιότητας ζωής, της δημιουργίας της εργασία, στην οικονομία, την εφορία, τα μέσα μεταφοράς, την κινητικότητα και το περιβάλλον. Τίποτα λιγότερο, τίποτα περισσότερο. Πάρα πολύ φιλόδοξο το πρόγραμμα. Στην ανακοίνωση της 30ης Ιουνίου η Κομισιόν επίσης έθεσε ε, ένα πολύ φιλόδοξο στόχο, αλλά ε, έχουμε και την πτυχή της επικουρικότητας. Η επικουρικότητα δραματίζει πολύ μεγάλο ρόλο αυτή τη στιγμή. Εδώ μιλάμε για εναρμονίσεις, για συντονισμούς και πρέπει να έχουμε κατά νου ε, δεν λέω ότι δεν το είπατε εσείς, απλώς λέω ότι πρέπει να, να θυμόμαστε ότι το άρθρο 195 της συνθήκης αποκλεί κάθε εναρμόνιση ε, για ε, σε νομοθετικές διατάξεις. Όμως, ποιος είναι ο ρόλος που έχετε να διαδραματίσετε εσείς, αφού ο Επίτροπος Γιάννη, σαφή τα είπε τα πράγματα και είπε ότι δεν, θέλουν να δεν θέλει να υπάρχουν εμπλοκές σε τομείς όπου έχουμε επικουρικότητα. Εσείς τώρα θα έπρεπε να δείτε πώς μπορείτε να εξορροπήσετε τα διάφορα συμφέροντα των κρατών για να προωθήσετε τον ευρωπαϊκό τουρισμό αυτό είναι πάρα πολύ λεπτό ω αποστολή. Ξέρετε ότι ο ε, τουριστικό τομέα δουλεύει πάρα πολύ ο ένα τον άλλο μεταξύ κρατών και είναι ανταγωνιστέ τα κράτη. Έτσι λοιπόν ε, πολλές φορές αυτή ενοποίηση ενό κοινού τουρισμού θα μπορούσε να αποφέρει κάποια μειονεκτήματα. Είναι ιδιαίτερα πολύπλοκη και δύσκολη κατάσταση, Όμω, αν τα καταφέρετε, εγώ θα σα χειροκροτήσω. Εγώ πραγματικά πιστεύω ότι είναι δυνατό κάτι τέτοιο. Σα ε, προσφέρω την υποστήριξή μου. Πιστεύω ότι είμαστε σε μία πάρα πολύ σημαντική στιγμή και πάλι να σας πω καλή επιτυχία και καλή δουλειά. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον κύριο Δεγκράντες. Ευχαριστώ κύριε Υπουργέ για αυτήν την περιεκτική παρουσίαση που κάνετε για αυτό το πολύ περίπλοκο ζήτημα. Δεν υπάρχει μάλλον κανένας άλλος κλάδος ο οποίος να αναπτύχθηκε ε, τόσο πολύ, τόσο αλματοδός κατά τελευταίες δεκαετίες σε ό,τι αφορά τη δυνατότητα αλλά και τη βούληση των άνθρωπων να ταξιδέψουν. Ε, πράγμα βέβαια το οποίο σχετίζεται και με την ενοποίηση της Ευρώπης ε, και την κατάρριξη των συνόρων αφενός αλλά και ε, με τον περισσότερο ελεύθερο χρόνο που έχουν οι άνθρωποι στη διάθεσή τους, το πράγμα βέβαια το οποίο εξαρτάται και από την οικονομική τους κατάσταση. Έτσι λοιπόν προέκυψε ένας τουρισμός τον οποίο ακόμα και σήμερα αποκαλούμε βιομηχανία του τουρισμού και μιλάμε για ένα κλάδο ο οποίος πλέον αποτελεί οικονομικό παράγοντα αφού ε, συμβάλλει με σημαντικό ποσοστό στο ΑΕΠ. Άρα λοιπόν σε ό,τι αφορά την τουριστική ανάπτυξη δεν νομίζω πως θα πρέπει να χρηματοδοτηθεί με περισσότερα κονδύλια γιατί αυτή ήδη λαμβάνει χώρα. Υπάρχει δυναμισμός. Εκείνο που σωστά είπατε και εσείς που θα πρέπει να γίνει είναι να αξιοποιηθεί καλύτερα και να υπάρξουν τέτοιες δράσεις η ε, ε, τουριστική υποδομή. Τώρα, εάν αναλογιστούμε και όταν συζητάμε το μέλλον του τουρισμού, ε, είναι σαφές ότι προφανώς και αναφέρεται και στη συνθήκη της Λισαβόνας ακριβώς λόγω της αυξανόμενης σημασίας του. Και το ερώτημα που τίθεται είναι κατά πόσο μπορούν να εξοικειωθούν ο ένας με, ε, τον άλλον ε, οι άνθρωποι στις διαφορετικές ε, χώρες ή αν τα ταξίδια τα οποία γίνονται γίνονται για την απλή επίσκεψη ενός συγκεκριμένου αξιοθέατου ή προκειμένου κάποιος να περάσει για παράδειγμα στο άλλο ημισφαίριο μία μικρή περίοδο αφού λοιπόν έχουμε να κάνουμε ένα σημαντικό οικονομικό παράγοντα και υπάρχουν ολόκληρες ε, περιοχές οι οποίες έχουν βασίσει την ε, οικονομία τους ε, στον τουρισμό, αντιλαμβανόμαστε ότι υπάρχουν και σαφείς κίνδυνοι. Δηλαδή να υπάρχει ένα είδος μονοκουλτούρας, δηλαδή μονοσδιάστατης κουλτούρας σε ό,τι αφορά τον τουρισμό. το ότι ακριβώς έχει αναπτυχθεί σε ένα είδο βιομηχανία ο τουρισμό. καταδεικνύει ακριβώς ότι δεν έχουμε διαχειριστεί πάντα με τον σωστό ε, τρόπο την ε, τουριστική ανάπτυξη και ε, συχνά δηλαδή έχουμε βασιστεί απλώς και μόνο στη σύμπτωση και όχι σε ένα σωστό σχεδιασμό. Βλέπουμε δηλαδή να αυξάνεται ο ατομικό, ο εξατομικευμένο ε, τουρισμό ε, και για παράδειγμα, εγώ στην ε, δική μου πόλη στο Βερολίνο βλέπουμε ρυθμού ετήσιους ανάπτυξη τη του 20%, ανοικοδόμηση ξενοδοχείων σε κάθε γωνιά, ενώ ο κλασικό, αν θέλετε μαζικό τουρισμός που το μόνο που θέλει είναι παραλία και ήλιο έχει μειωθεί δραστικά σε ορισμένες περιοχές 20 30% υποχώρηση Στου ε, αριθμού των επισκεπτών, πράγμα βέβαια το οποίο ε, δημιουργεί και μεγάλε κρίσει το οποίο τι απασχόλησε σαν γιατί και οι προορισμοί του οποίου επιλέγουν οι τουριστέ έχουν αλλάξει. Άρα λοιπόν εδώ σε αυτό το επίπεδο θα πρέπει να προσπαθήσουμε να θέσουμε ένα πολιτικό πλαίσιο όπως το περιγράψατε και ο οποίος αναφέρεται, αριθμείται στην ε, σχετική ανακοίνωση της Επιτροπής. Εκείνο όμως που θα πρέπει να γίνει και εδώ έρχεται, πρέπει να συμβάλλει η Ευρωπαϊκή Ένωση, ε, με μια εξέταση του πώς ακριβώς έχει εξελιχθεί ο τουρισμός, πού έχουν ε, παγιωθεί ορισμένες ε, τάσεις και πού έχουν προκύψει νέες, ούτως ώστε να οργανώσουμε με σωστό τρόπο τη δική μας πολιτική. Και πέρα από την Οικονομική Επιτροπή, η δική μας Επιτροπή είναι εκείνη που είναι κατεξοχήν αρμόδια για τον ε, τουρισμό, γιατί προφανώς χωρίς κατάλληλα μέσα μεταφοράς και σωστή οργάνωση δεν μπορώ να ταξιδέψω, άρα λοιπόν πρέπει να υπάρχει ε, συσχέτιση ε, μεταξύ μεταφορών και τουρισμού. Είναι λοιπόν ένα διατομιακό, κλασικό διατομιακό ζήτημα ο τουρισμός που αφορά αφενός την προσωπική ανάπτυξη, ατομική ανάπτυξη του κάθε ανθρώπου, αφετέρου την γνωριμία μεταξύ των ανθρώπων, μετά ως ένα τρίτο στοιχείο Ω ε, παράγοντα οικονομική ανάπτυξη, και ω ένα τέτοιο στοιχείο ένα ε, βιώσιμο ε, κλάδο τη οικονομίας και για το μέλλον. Άρα λοιπόν μπορείς, μπορεί να αποτελέσει ο τουρισμό πράγματι μια σημαντική πρόκληση για την Ευρώπη. Ευχαριστώ κυρία Δέλερ. κυρία Τικάου, παρακαλώ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Σας ευχαριστούμε κύριε Υπουργέ για την παρουσία σας εδώ σήμερα. Πολύ σύντομα. Θα ήθελα να σας ρωτήσω άλλη Βελγική Προεδρία. Θα συνεχίσει την πρωτοβουλία που αναλήφθη από την Ισπανική Προεδρία για τον κοινωνικό τουρισμό. Το πρόγραμμα Καλυψό ολοκληρώθηκε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Επρόκειτο να παρουσιάσει κάποιες κατευθυντήριες γραμμές σε σχέση με τον κοινωνικό τουρισμό στα κράτη-μέλη αλλά θα ήθελα να μας πείτε αν η Βελγική Προεδρία θα δώσει συνέχεια σε αυτή την πρωτοβουλία και στο ίδιο πλαίσιο. Να υπογραμμίσω το ότι σήμερα πολύ λίγα άτομα με ειδικέ ανάγκες ε, ταξιδεύουν, όχι μόνο για να μεταβούν από το ένα μέρος στο άλλο, αλλά δεν πηγαίνουν σε κρουαζιέρες λόγω χάρη ή σε τουρ. Έτσι λοιπόν, γι' αυτό θα πρέπει να σκεφτούμε και πέρα από τις μεταφορές, θα πρέπει να σκεφτούμε γενικά ποια είναι τα δικαιώματα των ατόμων αυτών στο εσωτερικό του τουριστικού κλάδου και κάτι ακόμη σε σχέση με τα πακέτα. Τα οργανωμένα ταξίδια. Η Κομισιόν ε, έχει υποσχεθεί ότι θα αναθεωρήσει τη σχετική οδηγία Είχαμε μία συζήτηση στην Ολομέλεια, η οποία συζήτηση το θέμα εισήχθη από την Επιτροπή ΕΜΚΟ και θέλω να ρωτήσω ποιες είναι οι προοπτικές στον τομέα αυτό. Έχετε κάποιο χρονοδιάγραμμα κατά νου ή το έχετε συμπεριλάβει στο πρόγραμμα της Βελγικής Προεδρίας. Ευχαριστούμε κύριε Τικάου. Να σας ξαναδώσω το λόγο κύριε Υπουργέ να προσθέσω κι εγώ μια-δυο ερωτήσεις που έχω κατά νου. Όσα υπόθηκαν είναι ενδιαφέροντα. Ακούσαμε τίποτα και ο Γιώργο Τζάιλερ για το ότι ο τουρισμός είναι κάτι εγκάρσιο και πολυτομεακό εξού και μεγάλη δυσκολία να τον εντάξουν τον τουρισμό στις πολιτικές. Τώρα, η πρώτη μου ερώτηση αφορά ένα θέμα που αναφέρθηκε από την κυρία Γιάλα. Δεν υπάρχουν ε, φορείς ή πολιτικά μέσα στο ιστορικό αυτού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ούτε της Κομισιόν, δηλαδή στο ιστορικό των οργάνων μας δεν υπάρχουν ειδικοί πολιτικοί φορείς για το τουρισμό. Βρίσκουμε ε, ότι στην ε, Κομισιόν ε, και στο Κοινοβούλιο το βρίσκομαστε σε διάφορα ρυθμιστικά σημεία, όμως όταν ε, θέλουμε στη συνέχεια να υποστηρίξουμε τις δράσεις για τις οποίες μιλήσαμε, λέμε πού θα βρούμε τα κονδύλια στα διάφορα ταμεία στα διάφορα ταμεία για τη γεωργία, για το περιβάλλον κτλ. Έτσι λοιπόν νομίζω ότι ε, είναι σαν να κάνουμε φιλανθρωπία εδώ για να το δώσουμε στα ορφανά. Γιατί δεν μπορούν να πάνε να αγοράσουν καινούργια παιχνίδια στο μαγαζί. Έτσι λοιπόν ε, υπάρχει ένα πραγματικό πρόβλημα. Εσείς σκοπεύετε από κοινού με την Κομισιόν μήπως ε, να σκεφτείτε να δημιουργήσουμε μία δομή εργαλείων πολιτική, οικονομική που να επιτρέπει να εξεύρουμε αυτά τα μέσα ε, για να θέσουμε σε εφαρμογή τις Πολιτιστικέ πολιτικές και επίση έχετε την εντύπωση ότι υπάρχει μια εσωτερική για μια εξωτερική αγορά στην Ευρώπη που δεν έτσι διασφίσει, γιατί ε, στο εσωτερικό της Ευρώπης εξακολουθεί να βρίσκεται η μεγαλύτερη αγορά και δεν νομίζω ότι θα απευθυνθούμε με τον ίδιο τρόπο στους Βορειοαμερικανούς ή στους Βραζιλιάνους. Έχετε, ή στους Κινέζους, έχετε λοιπόν ε, την ε, πρόθεση να διαφοροποιήσετε την εσωτερική αγορά από την εξωτερική αγορά ή μήπως ε, θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για το άνοιγμα της αγοράς. Και νομίζω ότι εδώ πολύ σωστά υπόθηκε ότι υπάρχει και ανταγωνισμός μεταξύ των κρατών. Και δύο τελευταία σχόλια. Κάτι για την κατάρτιση. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε ένα πρόγραμμα κατάρτισης ε, για τα τουριστικά επαγγέλματα, γιατί πάρα πολλές οι άνθρωποι αυτοί είναι ιδιαίτερα αιρεσιτέχνες και ξέρετε ότι αυτό προκαλεί προβλήματα γιατί έχει αντίκτυπο και στην αποδοτικότητα του τομέα, στην κερδοφορία και επίση. Ε, μήπως θα προτεθεί κάτι για το περιβάλλον γιατί πράγματι ο τουρισμός μπορεί να αλλάξει τον τουρισμό αλλά το περιβάλλον Μπορεί να αλλάξει επίση και τουρισμό. Βλέπουμε ότι έχουμε την κλιματική αλλαγή και κάτι τέτοιο μπορεί να έχει επιπτώσεις ε, ε, για τον τουρισμό που μπορεί να έχουμε στη Μεσόγειο ή στο Βορρά. Κάτι τέτοιο προοδευτικά εντάσσεται στην πραγματικότητα. Και σας δίνω το λόγο κύριε Υπουργέ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να ξεκινήσω από το τέλος των ερωτήσεων για να αναφερθώ και σε κάποια ζητήματα τα οποία είχα θίξει στην αρχική μου παρουσίαση. Ε, προφανώς λοιπόν ο τουρισμός αποτελεί μια πολιτική η οποία είναι πολύ σημαντική για πολλούς και εδώ ε, στο Κοινοβούλιο αλλά και για πολλούς άλλους. Ε, δηλαδή μιλάμε για μια αναπτυξιακή οικονομική πολιτική η οποία είναι σημαντική για πολλού και έχει λάβει αυτή τη σημασία και μέσω της συμπεριληψή του τουρισμού ε, στη συνθήκη της Λισαβόνα. Αλλά πάντα, πάντα ε, υπό ε, την αρχή της επικουρικότητας έχει συμπεριληφθεί η συνθήκη της Λισαβόνα, ο τουρισμό. Μιλάμε για έναν ε, ε, τομέα της ε, συνένεση, μη δεσμευτικό τομέα και προφανώς είναι φιλόδοξη η Βελική Προεδρία σε σχέση με τα όσα προτείνει γιατί αυτό που θέλουμε να επιτύχουμε είναι το καλύτερο δυνατό. Το τι θα πετύχουμε στο τέλος είναι κάτι το διαφορετικό αλλά είναι σαφές και από τη συζήτηση ότι εάν θέλουμε να έχουμε έναν επιτυχή τουριστικό κλάδο στην εσωτερική μας αγορά αλλά και προς τα έξω θα πρέπει να έχουμε συγκεκριμένες κατευθύνσεις τις οποίες θα, θα θέσουμε κατευθύνσεις, προσεγγίσεις τις οποίες θα προωθήσουμε και τις οποίες θα πρέπει να αποτυπώσουμε και στα συμπεράσματα του Οκτωβρίου. Ε, είναι κάτι το διαφορετικό όταν ε, συζητάω για την εσωτερική αγορά ή όταν συζητάω για την ε, εξωτερική ας πούμε αγορά για άλλες χώρες. Και αυτό το αναφέρει και η ανακοίνωση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εάν θέλουμε να δώσουμε περισσότερη ορατότητα στην Ευρώπη, εννοούμε ορατότητα στην Ευρώπη απέναντι στου ανθρώπου εκτό Ευρώπη. Πώ θα το επιτύχουμε αυτό, όχι μέσω dumping ε, στις ε, τιμές, ε, για να πάρουμε ένα κακό παράδειγμα. Όχι, μπορούμε να το επιτύχουμε μόνο προτείνοντας ποιοτικό βιώσιμο περιβαλλοντικό ενδιαφέροντα τουρισμό, ο οποίος ε, είναι κατά συνέπεια καλύτερος από αυτό που μπορεί κάποιος να βρει σε μια άλλη περιοχή. Και αυτό ακριβώς αναφέρεται και στην ανακοίνωση και αυτό είναι, που συμφωνήθηκε και από τους ε, υπουργού στη Μαδρίτη. Αυτός είναι και ο στόχος τον οποίο προσπαθούμε να προωθήσουμε. Και σε αυτό το πλαίσιο έχουν να παίξουν σημαντικό ρόλο ε, οι παράγοντες στους οποίους δεν ανέφερα γιατί πραγματικά δεν είχαμε αρκετό χρόνο στη διάθεσή μας ε, ε, όπως αυτοί που αναφέρθηκαν από τον πρόεδρο για παράδειγμα πληροφορίες, ενημέρωση, εκπαίδευση. Προφανώ και αυτά έχουν να παίξουν σημαντικό ρόλο όταν λέμε ότι θέλουμε να προτείνουμε ποιοτικό τουρισμό. Χρειάζομαι δηλαδή κατάλληλο εκπαιδευμένο προσωπικό. Μετά ε, κοινωνική συμβατότητα αν θέλετε του ε, τουρισμού. Επένδυση δηλαδή εδώ και πάλι στο προσωπικό, στην επαγγελματική κατάρτιση. Εδώ έχουμε κάποια χρήσιμα εργαλεία τα οποία ήδη υπάρχουν σε ευρωπαϊκό επίπεδο και θα μπορούσαμε να φανταστούμε την ασωματώση του τουρισμού σε, αυτούς τους, ε, σε αυτά τα εργαλεία. Για παράδειγμα όταν συζητάμε περιφερειακά προγράμματα ή όταν βλέπουμε ότι μπορεί πράγματι να ενσωματωθεί η πτυχή του τουρισμού σε ένα τέτοιο πρόγραμμα. Ε, επίσης, ε, ε, λαμβάνω υπόψη αυτά που είπε ο Πρόεδρος σε ό,τι αφορά δηλαδή και την, τα διαρθρωτικά τα και την ανάπτυξη ότι θα πρέπει να δούμε ακριβώς πού βρίσκεται η ευρωπαϊκή πτυχή και πού είναι ιδιαίτερα σημαντικός ο τουρισμός. και ότι ε, η πτυχή του τουρισμού θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη σε διάφορα επίπεδα αποφάσεων τα οποία λαμβάνονται στο επίπεδο χάραξη τη πολιτική. Για παράδειγμα, ε, σε σχέση με την προστασία των καταναλωτών, σε σχέση με την ε, οδηγία για τα οργανωμένα ταξίδια. Και εκεί βλέπουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι εκείνη η οποία δίνει κάποιε γενικέ κατευθυντήρε γραμμέ για το τι πρέπει να γίνει. Και ε, Προφανώς και υποστηρίζουμε ε, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε σχέση με, μια, με τη σχετική της εδώ προσπάθεια αλλά χωρίς να μπορώ να σας πω κάτι πιο συγκεκριμένο, ο συνάδελφός μου που είναι αρμόδιος ε, έχει έρθει σε επαφές ε, με την εταιρεία Ρέντιν και συνεργάζεται μαζί της ώστε να προωθηθεί αυτό το ζήτημα. Ε, μιλάμε λοιπόν για σημαντικά εδώ θέματα ε, αναφερθήκαν και μια σειρά από παραδείγματα για την κινητικότητα. Μπορούμε λοιπόν σε διαφθορτικό επίπεδο να προωθήσουμε αυτά τα ζητήματα ε, και ε, αναφέρθηκε γι' αυτό ότι θα πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη να υπάρξει μεγαλύτερη προώθηση, μεγαλύτερη ορατότητα του τουρισμού. Εάν λέμε ότι χρειαζόμαστε μια τέτοια ποιοτική, μια πολιτική ποιοτικού και βιώσιμο τουρισμό. Αυτά τα στοιχεία δηλαδή συγκαταλέγονται σε μια τέτοια πολιτική χωρί όμω να μιλάμε για εναρμόνιση. Δεν θέλουμε δηλαδή να έχουμε έναν ενιαίο κλάδο, βιομηχανία, τουρισμού, γιατί κάτι τέτοιο θα ήταν εντελώ διαφορετικό ε, με αυτό που θέλουμε να κάνουμε. Πολλοί δηλαδή οι οποίοι ε, προώθησαν ε, μια ενιαία προσέγγιση τελικά έχασαν κάποιες από τις μεγαλύτερες ευκαιρίες που είχαν στη διάθεσή τους όταν υπήρχε δηλαδή πολύ μεγάλη εναρμόνιση μεταξύ διαφορετικών περιοχών. Όχι. Δεν χρειαζόμαστε εναρμόνιση. Θέλουμε να διατηρήσουμε πάση θυσία την ποικιλομορφία, την διαφορετικότητα μεταξύ των περιοχών μα, γιατί αυτό αποτελεί το πλέον σημαντικό χαρακτηριστικό μα. Αυτό είναι που θέλουν οι περιοχέ. Αυτό είναι και το στοιχείο που έχουν κατανοήσει πολύ καλά πλέον οι ε, τουριστικοί στα κράτη-μέλη. Γνωρίζει δηλαδή ο κλάδο το τι μπορεί να πουλήσει και τι δεν μπορεί να πουλήσει. Είναι ένα ζήτημα δηλαδή εμπορικότητα του, του, του, του τουριστικού προϊόντος. Από εκεί και μετά αυτό δηλαδή στο οποίο, ε, αυτό για το οποίο συζητούμε είναι η ποιότητα την οποία θα πρέπει να δώσουμε ε, στον τουρισμό σε αυτές τις περιοχές για να επιτύχουμε κάτι περισσότερο. Σε ό,τι αφορά το Ευρωπαϊκό Φόρουμ Τουρισμού το οποίο θα λάβει χώρα στην ε, Μάλτα αναφέρθηκε από τη συνάδελφο ε, μπορεί να ακούγεται λίγο περίεργο, αλλά δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό, δηλαδή να διοργανώνεται σε χώρα διαφορετική από την ε, διοργανώτρια χώρα. Και δεν λαμβάνει χώρα στις Βρυξέλλες γιατί είχε λάβει χώρα πέρυσι στις Βρυξέλλες. Δηλαδή η Τσεχία πέρυσι είχε διοργανώσει το Ευρωπαϊκό Φόρουμ Τουρισμού στις Βρυξέλλες. Εμείς λοιπόν αποφασίσαμε να λάβει χώρα στη Μάλτα λόγω και της ε, πολύ, καλ, ε, πολύ καλής συνεργασίας που έχουμε με τη Μάλτα, Μάλτα και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν θεωρήσαμε δηλαδή πως αποτελεί κάτι το αρνητικό. Ε, δείχνει κάτι τέτοιο μάλιστα ότι το Βέλγιο ειδικότερα σε ό,τι αφορά ζητήματα συνεργασίας βρίσκεται πολύ ψηλά και πραγματικά θεωρώ πως είναι κάτι το χρήσιμο. Κάτι το χρήσιμο και για το πρόγραμμα ε, της ίδιας της Βελικής ε, Προεδρίας. Τώρα, σε σχέση με ένα ακόμα ε, ζήτημα που αναφέρθηκε, ναι, σε ό,τι αφορά την εξωτερική αγορά πρέπει να αυξήσουμε την ορατότητα της Ευρώπης, όπως προαναφέρθηκε, θα μπορούσαμε να έχουμε μια κοινή παρουσίαση είναι εργαλεία τα οποία μπορούμε να προωθήσουμε, αλλά το κυριότερο είναι προφανώς να βελτιωθούμε ως προς το τι ακριβώς παρουσιάζουμε προς τα έξω. Και ε, εδώ βρισκόμαστε σε επαρχές μιας χάραξης, της χάραξης μιας ε, ευρωπαϊκής ε, πολιτικής. Αυτό ίσως είναι δηλαδή, το πιο σημαντικό καθήκον μας. Να δημιουργήσουμε μια σαφή βάση για τη χάραξη της πολιτικής μας. Ε, το είπα και στην αρχική μου παρουσίαση ότι αυτή είναι η προτεραιότητα της δικής μας πολιτικής προεδρίας, δηλαδή η δημιουργία μιας σαφούς βάσης. Γιατί έχουμε πολύ διαφορετικές ε, προσλήψεις σε τι ακριβώς συνίσταται η πολιτική τουρισμού. Διαφορετικές λοιπόν αντιλήψεις ανάμεσα στα κράτη-μέλη και θα πρέπει κατά συνέπεια να βρούμε μια ομοφωνία εδώ, μια συνένεση. Εμείς ε, κινούμαστε εδώ μη δεσμευτικά. Και ε, απαντώντας στο ερώτημα του γιατί ακόμα δεν έχουν δημοσιευτεί κάποια έγγραφα οι non-papers ε, είναι οφείλεται στο γεγονό ότι 30 ε, Ιουνίου δημοσιεύτηκε η σχετική ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής οπότε εργαζόμαστε τώρα πολύ εντατικά επί αυτής, αυτού του εγγράφου βάσης ε, το οποίο θέλουμε να συζητήσουμε και το οποίο θα, θέλουμε, θα θέλαμε να παρουσιάσουμε στο Συμβούλιο των Υπουργών ε, τον Οκτώβριο. Και σας είπα ήδη το τι πιστεύουμε πως θα πρέπει να συμπεριληφθεί σε κάθε περίπτωση στα συμπεράσματα που θα προκύψουν ε, από το Συμβούλιο. Σε ό,τι αφορά τον κοινωνικό τουρισμό, να σας πω ότι χαίρομαι και εγώ πολύ για το γεγονό ότι έχουμε την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής απέναντι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δηλαδή ότι πράγματι όλοι αντιλαμβάνονται αυτή την ανάγκη το να δώσουμε εδώ μια συνέχεια και σε σχέση με το πρόγραμμα Καλύψο. Ε, εμείς λοιπόν θέλουμε να δραστηριοποιηθούμε στον χώρο του κοινωνικού τουρισμού και γι' αυτό υποστηρίζουμε και τη σχετική πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που αναφέρεται στην ανακοίνωση, δηλαδή να δοθεί συνέχεια στο πρόγραμμα Καλυψό με την εστίαση σε τέσσερις ε, συγκεκριμένε ε, ομάδες ε, στόχους, ηλικιωμένους, ομάδες, άτομα με αναπηρία, οικογένειες με χαμηλό εισόδημα. Έτσι λοιπόν προσπαθούμε να έχουμε και κάποια συγκεκριμένα, κάποια απτά συμπεράσματα σε ό,τι αφορά τον κοινωνικό τουρισμό σχετικά με το πώς μπορεί να δραστηριοποιηθεί εδώ η Ευρώπη. Ε, τώρα, ας περάσουμε σε ένα από τα πιο αγαπημένα αν θέλετε ζητήματα και των Ευρωβουλευτών και των Υπουργών τη χρηματοδότηση γιατί είναι πολύ ωραίες όλες αυτές οι ιδέες τις οποίες ανταλλάξαμε ε, και τις οποίες σας ανατείνασα αλλά το ζητούμενο είναι πώς μπορούμε να υλοποιήσουμε αυτές τις ιδέες ποιες δυνατότητες έχουμε στη διάθεσή μας ε, ε Προφανώ οι δημοσιονομικές προοπτικές για την περίοδο μετά το 2013 θα είναι εκείνη που θα, α, ε, κατά την οποία θα χρειαστεί έτσι, να εστιάσετε σε αυτό το ζήτημα. η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήταν πολύ προσεκτική σε σχέση με αυτό το ζήτημα στη δική της ε, ανακοίνωση και αυτό βέβαια το έκανε ε, για σαφείς λόγους. Θα πρέπει δηλαδή να επιτύχουμε καταρχήν μια διατήρηση των χρηματοδοτικών εργαλείων των προοπτικών κατά συνέπεια που έχουμε ε, σε αυτή τη φάση στη διάθεσή μας, δηλαδή ας είμαστε και λίγο πραγματιστές σε ό,τι αφορά την πολιτική μας. Εμείς από την πλευρά τη ε, δική μα ε, Προεδρία θα προσπαθήσουμε να προωθήσουμε αυτού του στόχου και σε κάθε περίπτωση ο τουρισμό. Εφόσον έχουν συμφωνήσει επί τη τη Λισαβόνα τα κράτη-μέλη, θα πρέπει τα κράτη-μέλη να συμφωνήσουν πω ναι, θα πρέπει να δραστηριοποιηθεί εδώ η Ευρωπαϊκή Ένωση συμπληρωματικά προ τα όσα πρότουν τα κράτη-μέλη. Και ναι, θα χρειαστεί να υπάρξουν χρηματοδοτικά εργαλεία, ταμεία για τον τουρισμό. Τώρα το ποια ακριβώς μορφή θα λάβουν δεν το ξέρουμε ακόμα, δεν μπορούμε να το συζητήσουμε ακόμα, αλλά ό,τι άλλο ε, πούμε θα ήταν τελείως αντιπαραγωγικό και θα ερχόταν σε αντίθεση με τα όσα είπαμε. Η συνθήκη της Λισαβόνας προβλέπει κάτι συγκεκριμένο και κατά συνέπεια θα πρέπει να το τηρήσουμε. Άρα θα πρέπει να προσπαθήσουμε να βρούμε εδώ μία συνένεση μεταξύ των 27 κρατών μελών, ούτως ώστε να λάβει την ορατότητα που χρειάζεται ο τουρισμός και στο επίπεδο της χρηματοδότησης. Αυτά. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Υπουργέ για την πρώτη αυτή επαφή για ένα θέμα που αξίζει τον κόπο να το ξαναδούμε. Μας πείσατε, βλέπουμε τις δυσκολίες θεσμικές, δημοσιονομικές, προβλήματα φαντασίας, αλλά υπάρχουν και μεγάλες προοπτικές. Και όλοι οι συνάδελφοι θα τα σκεφτούν όλα αυτά τους επόμενους μήνες, ιδιαίτερα το καλοκαίρι των 1,5 μήνα, στις διακοπές τους διακοπές μελέτης όπου επιτόπου θα μελετήσουν τα πρακτικά προβλήματα που τίθενται από την κινητικότητα, την υποδοχή, γαστρονομικά θέματα, ήλιος, κλίμα, ποδηλασία κλπ. Ευχαριστούμε πολύ.